Good afternoon, colleagues. Καλησπέρα, συνάδελφοι, λέει η πρόεδρος. Καθίστε παρακαλώ. Έχουμε πολλή δουλειά, αλλά θα είναι το απόγευμα αυτό πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε μια ανταλλαγή απόψη που υπόσχεται πολλά. First, uh, let me greet our uh... Οπότε πρώτα πρώτα να καλωσορίσουμε τους προσκεκλημένους μας. Θα γίνει ανταλλαγή απόψεων το απόγευμα με τον Σερ Julian King που είναι ο Επίτροπος για τα θέματα ασφαλείας. Έχουν επίσης τον ε, πρέσβη Τη Εστονίας που αντικαθιστά τον κύριο Άνβελ τον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου. Τον ε, Δεκέμβριο θα παρουσιάσει νομοθετική πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να βελτιωθεί η διαλειτουργικότητα του EDPS. Και η Προεδρία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότειναν μια τριμερή ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή μας, ώστε να προπαρασκευάσουν αυτήν την νομοθετική πρόταση. Άρα, δώσουμε στον κύριο Καρτέλ, τον κύριο Πρέσβη, τον λόγο, ο οποίος θα μας εξηγεί τι ανάγκε των κρατών μελών. Στη συνέχεια δε, τη σκητέλη θα πάρει ο Επίτροπος Κίνγκ, θα μας πει τις λύσεις που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις ανάγκες που θα καλυφθούν τις ανάγκες των κρατών μελών. Στη συνέχεια δε θα γίνει ανταλλαγή απόψεων. Πρώτα πρώτα η, η πρέσβη, η πρέσβηση Τάρελ θα λάβει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμοι βουλευτές. Κύριε Επίτροπε, να ευχαριστήσουμε την Επιτροπή που οργάνωσε τη σημερινή εκδήλωση για την διαλειτουργικότητα που θα εμπλέξει Συμβούλιο, Επιτροπή και Κοινοβούλιο και οργάνωσε αυτήν τη συνάντηση και πριν εμείς κατεβάσουμε την πρότασή μας. αυτό αποδεικνύει το πόσο σημαντικό θα είναι αυτό το νομοθέτημα ούτω ώστε οι βάσεις δεδομένων να λειτουργήσουν όπως πρέπει πρώτα-πρώτα. Ε, συγγνώμη εκ μέρους του Υπουργού μας, του κυρίου Άνβελτ, είναι ο υπουργό Εσωτερικών μας, αλλά ασθένιζε. Ο Νοέμβριος είναι σκληρός, δύσκολος μήνας στην Εστονία. Πολύ πιο σκληρός και αν ελέγχει το συνδυασμό από εδώ στις Βρυξέλλες. Οπότε για να αρχίσουμε τη σημερινή συζήτηση με κάποια δήλωση για να εξασφαλίσουμε τη λειτουργία της ζώνης ε, Σέγγεν χωρίς ε, έλεγχο στα εσωτερικά σύνορα. Αυτός είναι ο βασικός μας στόχος και όπως ξέρετε διακυβεύεται πάρα πολύ το μέλλον της επίτευξης αυτού του στόχου. Οπότε για να τα καταφέρουμε θα πρέπει οι αρχές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεργαστούν και για να διευκολυνθεί αυτή η συνεργασία έχουμε ήδη στήσει κάποια συστήματα πληροφορικής και θα συνεχίσουμε τα μέσα επόμενα χρόνια προς την κατεύθυνση αυτή έχοντας και άλλα συστήματα πληροφορικής. Έχουμε όλοι γίνει μάρτυρες ε, πάρα πολύ εντόνων κατά όλων μας των κοινωνιών όσον αφορά την διερεύνηση εγκλημάτων, καταπολέμηση τρομοκρατίας και θα πρέπει να δούμε τι διάδραση υπάρχει μεταξύ των συστημάτων πληροφορικής μας και, και ακριβώς πώς είναι δομημένα αυτά. Άρα η κατάσταση επιδέχεται ακόμα πολύ δουλειά. Και εμείς οι Εστονοί θέλουμε να μιλούμε με έργα και όχι με λόγια. Έχουμε ετοιμάσει ένα βίντεο το οποίο θα προβληθεί ευθύ αμέσω από τους συνεργάτες μας.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 Uh, Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε και θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Γη. Uh, Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας τα πει ο κύριος. Κίνη και κατόπιν θα ακολουθήσει η συζήτηση. Uh, well, well, thank you, Chair, uh, honourable members. Uh, it... Ευχαριστούμε. Να συνεχίσουμε Πρόεδρε, αγαπητοί κύριοι βουλευτέ, η δική μου ε, συνεισφορά δεν θα είναι τόσο ζωντανή, ε, αλλά θα προσπαθήσω τέλος πάντων και να συνεχίσω τα όσα έχουμε επανειλημμένα συζητήσει για κάποια από αυτά τα θέματα και ελπίζω ότι θα κάνουμε κάποια βήματα πρόοδου ακόμα και πριν υποβάλουμε επισήμως την νομοθετική πρόταση ακριβώς όπως ελέγχθη να τα συζητήσουμε τότε βέβαια ενδελεχώς με Αλλά όπως προαναφέρθηκε έχουμε τις χώρες ε, πρώτης γραμμής που προσθέτουν τα σύνορα, καταπολεμούν το έγκλημα, αλλά εμείς θα πρέπει να συντονιστούμε σε ευρωπαϊκό, σε ενωσιακό επίπεδο και να έχουμε κάποιο εργαλείο σημαντικό για αυτό το έργο να εξασφαλίσουμε ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υπάρχουν πλήρες πληροφορίες, ακριβείς, αξιόπιστες και προσβάσιμες. Θεωρώ ότι έχουμε σημειώσει αρκετή πρόεδρο όσον αφορά το νέο σύστημα, αυτό που χθες παρουσιάστηκε στο Συμβούλιο. Ευχαριστούμε και την Προεδρία και όλους τους άλλους όσοι βοήθησαν. Ε, ε, κυρία Πρέσβη, εσάς και την Προεδρία σας. Επίσης έχουμε το αίτιος και ξέρω ότι σας ενδιαφέρει πολύ και για αυτό σας ευχαριστούμε για όσα κάνουν και ελπίζουμε μέχρι το τέλος του να έχουμε συμφωνήσει. Επίσης έχουμε κάποιες άλλες προτάσεις για να αναβαθμίσουμε τα υπάρχοντα συστήματα, το σύστημα πληροφοριών του Σέγγεν για αγνοούμενους, για έγκλημα της Eurodac για νόμους μετανάστες, το έκρης για καταδικασμένους από τρίτες χώρες και χρειάζεται να σημειωθεί και να κατέληψει συμφωνία. Πρόσφατα, ακριβώ όπω έλεγε το βίντεο, χρειαζόμαστε ισχυρά θωρακισμένα σύνορα, ευφυή σύνορα, να κλείσουμε τα ε, τυχόν κενά που υπάρχουν, αλλά τέλο πάντων, ακόμα και αν συμφωνήσουμε για όλα αυτά τα ζητήματα, ακόμη θα υπάρχουν κάποια θέματα, θα υπάρχουν κάποιε ασυμβατότητε μεταξύ κάποιων συστημάτων, ε, τα οποία δεν επικοινωνούν όπω θα έπρεπε. Ε, Σύνοριοφύλακε, δικαστικέ αρχέ, διοικητικέ αρχέ θα πρέπει να έχουν πρόσβαση ταχεία στα δεδομένα που χρειάζονται για να μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά του. Θα πρέπει επομένω να διευκολύνουμε όλε αυτέ τι αρχέ, να παίρνουν τι πληροφορίε πιο γρήγορα, πιο απλά και πιο κατανοητά. Και ένα παράδειγμα Τώρα ελέγχουμε όλου όσου θέλουν να μπουν στο έδαφο Ευρωπαϊκή Ένωση, χρησιμοποιώντα το SIS. Αλλά δεν είναι πάντοτε εύκολο να γίνει ο ίδιο έλεγχο σε άλλε βάσει δεδομένων, όπω το σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις το Visa. Οπότε δεν μπορούμε να έχουμε καποιούς παράλληλη έρευνα στο Eurodac και στο VISA. Και όταν κάνει κάποιον έλεγχο η αστυνομία με κάποιον από τρίτη χώρα που δεν έχει ταξιδιωτικά έγγραφα, τσεκάρει τι γίνεται ως το, το, το όσον αφορά τη μετανάστευση. Αλλά αν θέλουν να δουν και αν αυτό έχει διαπράξει κάποιο ε, έγκλημα μικρή βαρύτητος θα πρέπει να μπορούν να μπουν στην ε, βάση δεδομένων αλλά όταν έχουμε κάποια πιο βαριά εγκλήματα η τρομοκρατία η αστυνομία τότε δεν μπορεί να δει τα, τις λαθρομετανέθευσεις στο Eurodac ούτως ώστε να μπορέσει να μπει στη βάση δεδομένων για το ποιοι έχουν ε, θεώρηση διαβατηρίου ε, και έτσι να τσεκάρει το ΒΙΣ. Και αυτοί από τις τρίτες χώρες ε, πολλές φορές έχουν άλλες ταυτότητες και τις χρησιμοποιούν ανά, ανακράτος μέλος. Οπότε γι' αυτό και θα πρέπει και αφού περάσουν οι προτάσεις που θα υποβάλουμε να πρέπει να συνεχιστεί η δουλειά γιατί υπάρχουν ε, αυτού του είδους οι νεκρές γωνίες όπως υπήρχε, υπάρχουν αυτά τα κενά και άρα θα πρέπει να ε, δούμε το ότι οι υπηρεσίε που οποίες για το έργο μας θα πρέπει να έχουν την πλήρη εικόνα. Αυτό σημαίνει ότι οι τρομοκράτες αλλά και οι άλλοι εγκληματίες θα μπορούσαν να κρυφτούν πίσω από πολλαπλές ταυτότητες, από πλαστές ταυτότητες, οπότε και αναλάβουν υπόψη ότι αυτό έχει ήδη συμβεί. Να, ας πούμε ε, στην περίπτωση της επίθεσης των Μοκαδί στο Βερολίνο. Οπότε ελπίζουμε να προχωρήσουμε με τη, και με τη δική σας βοήθεια και είπαμε ότι αυτό είναι ανάγκη και αφορά όλο τον κόσμο. Έχουμε επίση την ε, πρόταση αυτή για τη διαλειτουργικότητα που θα κατεβάσουμε και έτσι αυτό το που θέλουμε να κάνουμε να καλύψουμε αυτέ τι ανησυχίε, τι μέρημνε και οπότε επεξεργαζόμαστε την πρόταση εδώ και αρκετό καιρό. Τα έχουμε πει επανειλημμένα μαζί και έχει γίνει όσον αφορά τα νομικά, τα τεχνικά, τα επιχειρησιακά θέματα ε, συζήτηση και έχουμε και την ε, ομάδα ψηλού επίπεδου εδώ και 12 μήνες έχουμε διαβουλευτεί με εμπλεκόμενους ε, κράτη-μέλη και συνεχίζεται η δουλειά σε τεχνικό επίπεδο και επίσης συνεχώς ε, ενημερώνουμε και εμπλέκουμε την γραμματεία της Επιτροπής σας. Και όταν ε, τα συζητήσαμε τον Μάιο, όπως θα θυμάται η Πρόεδρος, είχαμε πει ότι θα πρέπει να γίνει κοινή συζήτηση των τριών θεσμικών οργάνων, ούτως ώστε να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Έγινε αυτό έγινε και χθε το απόγευμα. Πολύ εξημών είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε, να μιλήσετε πάντων σε κάποιους ειδικού και εμπειρογνώμονες επίσης. Το τελευταίο εξάμεινο έγιναν ε, πολλές διαβουλεύσεις οπότε και επιβεβαιώθηκε η προσέγγιση που είχαμε χαράξει σαν πορεία αρχές του έτους και είπαμε θέλουμε ένα κεντρικό σύστημα για ασφάλεια, για τα σύνορα, για τη διαχείριση αυτών των θεμάτων που θα πρέπει να έχει διαλειτουργικότητα και για, τις, ε, και για το, το, το ΒΙΣ, ε, το EXIT, ε, το ETIAS, το οποίο το καινούργιο σύστημα που προτείνεται, το έκρις για καταδικασμένους από τρίτες χώρες για να τα πετύχουμε αυτά χρειαζόμαστε να συνδυάσουμε τα εξή τρία. Ε, να υπάρχει προσβασιμότητα στις διοικητικές αρχές ε, σε αυτά τα κεντρικά συστήματα ταυτόχρονα και να προστατεύονται τα κάποια δικαιώματα πρόσβασης τα οποία να, μην αλλάζουν αυτοί οι κανόνες πρόσβασης δηλαδή και να μπορούμε να έχουμε συνδυασμένα αποτελέσματα σε μία και μόνη οθόνη. Οπότε αυτό, αυτή, αυτή η πύλη ε, να μας δίνει την ευκαιρία για καλύτερη πρόσβαση και να είναι πιο παραγωγική η διαδικασία αυτή επίσης να υπάρχει ένα εργαλείο για τα δακτυλικά αποτυπώματα ούτως ώστε οι αρμόδιες αρχές να μπορούν να τσεκάρουν όλα τα συστήματα που έχουν τέτοια δεδομένα με το πάτημα ενός κουμπιού και βέβαια με την επιφύλαξη των ισχυών των δικαιωμάτων προσβασιμότητας ή σε αυτά τα συστήματα ανάλογα με το που μπορεί κανείς που δικαιούται να ε, προσφύγει, που μπορεί να ψάξει αλλά αυτό με παράδειγμα τρόπο επίσης ε, να υπάρχει κάποιο είδου κοινό μητρό για αποθήκευση των βασικών ε, στοιχείων των φυσικών προσώπων για όλα αυτά τα συστήματα και έτσι να μπορούμε να δούμε αν κάποιος ε, έχει διαφορετικές ταυτότητες που έχουν καταχωρηθεί στις διαφορετικές βάσεις δεδομένων. Τώρα πέραν από αυτά τα, τα, τους τεχνικούς άξονες που σας είπα έχουμε και άλλα θέματα που έχουν σχέση με, την, ε, με τις επεξεργασίες, με τις διαδικασίες ε, για την πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων. Λένε οι εθνικές αρχέ ότι έχουν πολλές δυσκολίες όταν θέλουν να επαληθεύσουν την ταυτότητα κάποιου από τρίτη χώρα στην επικράτειά τους. Όταν ε, δεν θέλει, δεν μπορεί κάποιος από τη χώρα να παρουσιάσει κάποια έγγραφα, δεν μπορούν οι αρχές να δουν τι γίνεται, να επαληθεύσουν τι ισχύει με τα υπάρχοντα συστήματα, ούτε και με το Eurodac, παρά μόνο εάν γίνει έλεγχος ε, στα πλαίσια της διαχείρισης μετανάστευσης. Ε, αυτό δεν είναι σωστό. Θα πρέπει να έχουν τα μεσαιεθνικές αρχές να δουν αν έχει διαπραχθεί κάποια απάτη περί την ταυτότητα στην επικρατειά τους και ε, έτσι θα πρέπει να έχουμε μια αναλογικότητα αστυνομικού ελέγχου στην ε, ζώνη Σέγγεν, χρησιμοποιώντα την δυνατότητα αυτή που να μα προσφέρεται. Ακριβώ όπω είπε η κυρία Πρέσβη, ούτω ώστε να μπορούμε να έχουμε αξιοποίηση του συστήματο Σέγγεν. Και στην ομάδα υψηλού επίπεδου θέλουμε να δούμε ποιε είναι οι δυσκολίε των αστυνομικών όταν θα καταπολεμήσουν ε, το βαρύ έγκλημα ή την τρομοκρατία όσον αφορά την πρόσβαση σε βάση δεδομένων για να εντοπιστεί κάποιο ε, θύμα ή θήτης. Επίσης θα έχουμε να έχουμε πιο ευφύη συστήματα και βέβαια όντως χρειάζεται να αναθεωρήσουμε τις κείμενες διατάξεις και τους κείμενους κανόνες και τα είπαμε ως Επιτροπή στην αρχή του έντος ότι θέλουμε πιο ενοποιημένους ε, κωδικοποιημένους κανόνες τέλο πάντων για την πρόσβαση σε αυτά τα συστήματα. Ούτε δεν θέλουμε τα δικαιώματα πρόσβασης να τροποποιηθούν. Το θέμα είναι πώς ασκούνται τα εν λόγω δικαιώματα και πώς θα χρησιμοποιηθούν πιο αποτελεσματικά. Έλεγχη ταυτοτήτων, ε, εφαρμογή του νόμου, Όλοι αυτοί οι έλεγχοι μας απασχολούν στην εκπόνηση της νομοθετικής πρότασης και είναι και η αξιολόγηση των επιπτώσεων ε, Τη άσκηση των θεμελιών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων στον ιδιωτικό βίο. Εάν επομένω συγκριθούν όλες αυτές οι προτάσεις και αλλάξουν σχετικέ διαδικασίες, θα εξασφαλίσουμε στο όλα αυτά να ισχύουν ε, με συμβασμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων και με αναλογικότητα και πάντως μπορώ να σας πω ήδη από τώρα ε, σε άλλε γραμμέ ποια ωφέλη βλέπουμε θα προκύψουν από αυτά τα μέτρα που θα θέλαμε να μας βοηθήσουν να εξασφαλίσουμε την ε, ε, πληρότητα, την ακρίβεια των δεδομένων, ε, ποιοτικά δεδομένα να είναι και έτσι να μπορέσουμε να μην έχουμε κατάτμιση των αποθηκευμένων πληροφοριών σε συστήματα που είναι αποσυνδεδεμένα και οι εθνικές αρχές να μπορούν να επισημάνουν τις πάντες περί ταυτότητα, και αυτοί που είναι στην πρώτη γραμμή όπως οι συνοριοφύλακες αλλά και οι δικαστικές αρχές να μπορούν να έχουν γρήγορα τις πληροφορίες που χρειάζονται για να επιτελέσουν το έργο τους. Όλα αυτά με αναλογικότητα όπως επιβάλλεται από τα θεμελιώδη δικαιώματα και η προστασία των δεδομένων και βέβαια με τήρηση των προβλεπωμένων ως δικαιώματα πρόσβασης. Και εμπλεκόμενοι πέραν άλλων όπως σας είπα είναι και αυτοί που θα ωφεληθούν από το την υπηρεσία εποπτείας ε, και από την υπηρεσία προστασίας των δεδομένων. Ε, και έτσι θα έχουμε μία αρχιτεκτονική όπως θέλουμε που θα καλύπτει όλες τις σχετικές μέρημνες και δεν μιλούμε για συγχώνευση των επιμέρους συστημάτων ούτε θα προτείνουμε συλλογή περισσότερων δεδομένων θέλουμε να αξιοποιηθούν περισσότερο τα υπάρχοντα δεδομένα λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιώματα ε, που ήδη προβλέπονται και έτσι θα αναβαθμίσουμε την ε, ασφάλεια, προς τα, τα σύνορα, θα διασυνορική απάτη θα καταπολεμηθεί, γενικά οι εγκληματίες, θα γίνει η Ευρώπη ασφαλέστερη στα πλαίσια ενός στεγανού ε, πλαισίου. Ε, αυτό θέλω ο κόσμος και πιστεύω ότι έχουμε τώρα την ευκαιρία να πετύχουμε αυτό το οποίο επιδιώκουμε με αυτές τις προτάσεις τις οποίες θα σας παρουσιάσουμε τον Δεκέμβριο και σας ευχαριστώ. Η Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πολύ τον Επιτροπό. Ας περάσουμε τώρα στη συζήτηση. Τέσσερις έχουν ζητήσει το λόγο μας τώρα. Okay, uh, first who asked for the floor was uh, Mr. Lopez Aguilar. Please. Ο κύριος Λόπεθ Αγγιλάρ, παρακαλώ. Thank you, Commissioner King. Thank you, Cecil, for your availability. Σας ευχαριστούμε, Επιτροπέ Κίνγκ, για την βούλησή σας να έρθετε εδώ στο Κοινοβούλιο και να ανταλλάξετε απόψεις ε, με τους ευρωβουλευτές για αυτή την πιο σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί ποτέ σε αυτό το τομέα. Η ζήτηση υπάρχει εδώ και χρόνια. Πλέον έχουμε αποκομίσει και εμπειρία. Οι συμφωνίες που έχουν συνεχθεί στο παρελθόν από έναν περιορισμένο αριθμό κυβερνήσεων ε, του σημερινού χώρου δικαιοσύνης και ασφάλειας πριν τη θεσμοθέτησή του, πριν τη συνθήκη της Λισαβόνας. Είχαμε ήδη εμπειρία λοιπόν ορισμένων κυβερνήσεων που κάλυπταν αυτή τη ζήτηση και κατέληγαν σε πολιτικές και τεχνικές συμφωνίες ανταλλαγής δεδομένων σχετικά με τις ε, και έρευνες και διαδικασίες και τα ποινικά μητρώα. Θα ήθελα να μας ε, πείτε δύο λόγια για την εμπειρία που έχετε λάβει εσείς υπόψη από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και δεύτερον, η εμπειρία μας δείχνει διδάγματα που πρέπει να συνεγάγουμε από τα κράτη-μέλη όπου έχουμε διαφορετικές ε, αρχές επιβόλης του νόμου και διαφορετικά επίπεδα αρμοδιοτήτων. Έχουμε λοιπόν μια αποκέντρωση των ε, πολιτικών ασφαλείας όπως στο Βέλγιο και στην Ισπανία για παράδειγμα όπου η διαλειτουργικότητα των δεδομένων μεταξύ διαφορετικών αστυνομικών δυνάμεων δεν έχει ακόμα διασφαλιστεί σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι η Επιτροπή έχει λάβει υπόψη αυτά τα διδάγματα. Προκειμένου όταν θα έχουμε την νομοθετική πρωτοβουλία να επανεξετάσουμε το σύνολο του συστήματος για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ε, δυσλειτουργίες. Να αντιληφθούν λοιπόν. Ευχαριστώ. Thank uh, Ευχαριστούμε κυρία Ζίπελ. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό το βιντεάκι που μας παρουσίασε η πρέσβης Εστονίας ήταν πραγματική έμπνευση και όπως πάντα όταν μας παρουσιάζει ο Επίτροπος Κίνγκ τα στοιχεία της λειτουργικότητα, όλα είναι εντυπωσιακά. Όμως, συνεχίζοντας ε, από τα όσα είπε ο συνάδελφος, κάποιες φορές έχουμε την εντύπωση ότι ιδίω τα κράτη-μέλη είναι υπέρ της ιδέας της διαλειτουργικότητας γιατί αυτό τους δίνει τη δυνατότητα ε, να κρύβουν έτσι κάτω από το χαλί ορισμένα εσωτερικά προβλήματα και τις λειτουργίες. Ακούσαμε τον Επίτροπο Κίν για κάποια προβλήματα που προέρχονται από το παρελθόν. Στι περισσότερε περιπτώσει το πρόβλημα δεν ήταν ε, η έλλειψη διαλειτουργικότητα. Απλώ αρχές στο εσωτερικό των κρατών μελών δεν αντίλασαν πληροφορίες μεταξύ τους ή απλώς ξεχνούσαν να εισαγάγουν πληροφορίες στις ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων. Αυτά τα προβλήματα δεν λύνονται με τη διαλειτουργικότητα. Αντίστοιχα και το θέσαμε και σε ορισμένα μέλη το ζήτημα της ποιότητας των δεδομένων. Δεν μιλώ για την τεχνική ποιότητα των δεδομένων όπως είναι τα τακτικά αποτυπώματα για παράδειγμα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να επιληθεί έτσι κι αλλιώς να υπάρχει ομοιόμορφη ποιότητα αυτών των δεδομένων. Αλλά τίθεται και το ζήτημα. Τι είδους δεδομένα και σε ποια φάση της έρευνας τα εισάγουμε στο σύστημα. Για παράδειγμα, όταν μιλούσαμε για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, από την αρχή ήταν σαφές ότι αυτό δεν αφορούσε τα μικρά ε, ίσονος σημασίας αδικήματα. Τι ισχύει τώρα όμως εμπροκειμένο, ότι υπάρχει σοβαρή υποψία εναντί ενός ατόμου, κάποιες υποψίες, υπάρχει γνώση ε, αξιόπινων πράξεων, πράξεων. Όπως και να έχει, το σημείο, το χρονικό σημείο μπορεί να διαφέρει, καθώς και το επίπεδο και αυτό οδηγεί σε κατακαιρματισμό των προσπαθειών καταβάλλονται προσπάθειες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ελπίζω και από το Συμβούλιο, να το οργανώσει όλο αυτό καλύτερα για να έχουμε τους ίδιους ορισμούς, τα ίδια ποιότητα, την ίδια ποιότητα δεδομένων, όχι μόνο για τα τεχνικά στοιχεία, αλλά ευρύτερα. Και σε ό,τι αφορά την ανάλυση της κατάστασης και λυπάμαι που το επαναλαμβάνω. Ξέρω ότι δεν είναι ευρωπαϊκή αρμοδιότητα, αλλά σε ό,τι φορά την ανάλυση καταστάσεων και δεδομένων για να δούμε ποιες πληροφορίες θα πρέπει να ε, ανέβουν σε όλες τις βάσεις δεδομένων, κάποιες φορές υπάρχουν κενά και στη δράση των ε, αρχών επιβολής του νόμου στα κράτη-μέλη, σε ό,τι φορά τον αριθμό των υπαλλήλων, την πιστοποίηση, τα προσόντα και ίσως σε ένα βαθμό εδώ ε, μπορεί η διαλειτουργικότητα να μας βοηθήσει σε ό,τι φορά την επεξεργασία δεδομένων, αλλά όχι στην ανάλυση τους, εάν δεν υπάρχει συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Κοέλιο, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους ε, δύο ομιλητές για τις παρουσιάσεις τους. Έχω ορισμένες γενικές παρατηρήσεις. Πρώτον, για το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών Schengen, το SAIS, το οποίο είναι και θα παραμείνει το κύριο σύστημα ε, στους τομείς ε, του ελέγχου των συνόρων και της ασφάλειας ε, στην επικρατειά μας. Δεν θέλω να περιευτολογήσω εδώ, απλώς ήθελα να πω ότι οι αλλαγέ ε, του πεδίου εφαρμογή θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και τι ιδιαιτερότητε και το σημερινό ρόλο του συστήματο στο ευρύτερο πλαίσιο διαχείριση πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, αυτό το μελλοντικό πακέτο για τη διαλειτουργικότητα την χάνει επεξεργασία εδώ και πολύ καιρό τώρα. Έχουμε και εκθέσει στι ομάδε ψηλού και η Επιτροπή τον έφερε προηγουμένω. Ανακοινώσει της Επιτροπής, μελέτες και τώρα σίγουρα θα έχουμε και μελέτες αντικτύπων. Αυτό θα μας επιτρέψει να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα όλων των συστημάτων. Επομένως, οι προτάσεις ε, για την λειτουργικότητα θα πρέπει πρώτα απ' όλα να έχουν δύο στόχους τη διασφάλιση της συνοχής μεταξύ όλων των πληροφορικών συστημάτων της Ένωσης και να παρέχουν τα καλύτερα τεχνολογικά εργαλεία για τον τελικό χρήστη. Φυσικά πάντα με σεβασμό προς τα θεμελιώδη δικαιώματα. Τα λεγόμενα silos ήταν στις περισσότερες περιπτώσεις ε, μια δυνατότητα και όχι τεχνικός περιορισμός στην αρχική φάση των ε, συστημάτων. Τώρα, όπως είπε σωστά ο Επίτροπος, δεν χρειάζεται να τα συγχωνεύσουμε. Χρειαζόμαστε ένα εργαλείο το οποίο θα επιτρέπει τις ε, ταχύτερες και πιο αποτελεσματικές αναζητήσεις και στα δύο συστήματα με πλήρη σεβασμό προς την νομική τους βάση. Η ενιαία οθόνη αναζητήσεων θα είναι ένα καλό παράδειγμα ε, πιο αποτελεσματικών εργαλείων προς τους ε, τελικούς χρήστες. Η διαλειτουργικότητα δεν είναι αυτός ο σκοπός, ούτε μπορεί να αξιοποιηθεί ως αποδιαπαπέως τράγος από τα κράτη-μέλη για να καλύψει την ε, έλλειψη εμπιστοσύνη μεταξύ τους. Πρέπει πάντα να υπάρχει και βούληση και διάθεση ανταλλαγή πληροφοριών. Αλλιώ δεν έχει νόημα. Και κάτι τελευταίο, Επίτροπε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή και εσάς προσωπικά ε, που έχετε προσκαλέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμμετέχει πλήρως σε αυτές τις διαδικασίες και ελπίζουμε να συνεχιστεί αυτή η επικοδομητική προσέγγιση. Ευχαριστούμε κυρία Γκριζμπέκ παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για την πολιτική μας ομάδα αυτό το θέμα αντιστοιχεί σε ένα αίτημα το οποίο έχουμε εκφράσει εδώ και πολλά χρόνια να υπάρχει καλύτερη ποιότητα και συνοχή των μέσων που έχουμε στη θέση μας για την ανταλλαγή πληροφοριών προκειμένου να έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα και ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις ε, προσπάθειες που έχει καταβάλει. Είναι σαφής η συνοχή που υπάρχει, η σαφήνεια, όπως ανέφερε και ο συνάδελφος Κίνγκ. Θέτει λοιπόν στη διάθεση ε, των εμπειρογνωμόνων ένα σύστημα το οποίο θα είναι ε, καθόλου επιχειρησιακό για να εξυπηρετεί τους πολίτες και προ του ίδιου του συστήματος ε, Σέγγεν. Συμφωνώ με αυτά που είπαν οι συνάδελφοι και περιμένω με ενδιαφέρον να ακούσω τις απαντήσεις. Δύο ερωτήσεις τεχνικής ε, φύσεως. Είπατε ότι έχουμε δύο συστήματα με δύο διαφορετικές βάσεις, με διαφορετικούς στόχους. Όταν υπάρχει ένα θετικό αποτέλεσμα hit, στα συστήματα. Ε, οι αρχές πώς έχουν πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες και ποιος ακριβώς ε, δίνει αυτή την πρόσβαση. Ποιες είναι οι δικλείδες ασφαλείας ως προς αυτό το μηχανισμό. Μετά, φαντάζομαι συμφωνείτε όλοι ότι δεν είναι το θέμα η ποσότητα, αλλά η ποιότητα των πληροφοριών. Και αυτό μας επαναφέρει στο γνωστό ερώτημα της ε, λειτουργίας ε, και της πρακτικής εφαρμογής των κρατών μελών. Αν δηλαδή τα κράτη-μέλη δεν εισάγουν ε, εγκαίρως και ορθώς τα απαραίτητα στοιχεία, πώς ε, περιμένετε να λύσετε αυτό το πρόβλημα. Γιατί δεν φταίει τελικά το μέσο της διαλειτουργικότητας, το οποίο είναι σημαντικό από μόνο του, δεν θα λύσει όμως από μόνο του αυτό το πρόβλημα. Μπορεί να είναι τεχνικό αυτό το ζήτημα, αλλά ουσιαστικά θέλουμε την συνοχή και την αποτελεσματικότητα. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι να προσθέσετε ως προς αυτό. Ευχαριστούμε κυρία Κοράτσα Μπίλτ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Χαιρετίζουμε και στηρίζουμε το έργο της Επιτροπής για τη Δηλειτουργικότητα και τις ε, βάσεις ε, δεδομένων ασφάλειας ε, για τα σύνορα. Τα περιμένουμε εδώ και καιρό όλα αυτά. Ε, συμφωνείτε μαζί μου κύριε Πίτροπε ότι το θέμα δεν είναι μεγαλύτερη πρόσβαση στα δεδομένα, αλλά η καλύτερη αξιοποίηση της διαθέσιμης πληροφορίας ε, με όλε τι δικλείδε ασφαλεία που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εμεί χαιρόμαστε που υπάρχει η προστασία δεδομένων ε, και η προστασία των θεμελιών δικαιωμάτων. Γιατί σκοπό είναι η προστασία του πολίτη αλλά και με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην καταπολέμηση του δυσμηριακού εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Συμφωνώ με την πρότασή σας. Είπατε ότι δεν είναι το θέμα η συγχώνευση των βάσεων δεδομένων, αλλά ε, να άρουμε τα στεγανά μεταξύ των βάσεων δεδομένων, να υπάρχει λοιπόν μία επαφή και συνοχή μεταξύ τους. Θέλουμε να μας βοηθήσετε να εξηγήσουμε στους πολίτες ότι όλα αυτά δεν αντίκεινται στην προστασία των ε, ε, του προσωπικού βίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, αλλά και προς τα κράτη-μέλη. Όπως είπε η Μπριγκίτε, υπάρχει μία πραγματική έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών σε ό,τι αφορά την ε, ανταλλαγή πληροφοριών. Εντάξει, αυτό δεν ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη, μην τους βάλουμε όλους στο ίδιο τσουβάλι, αλλά πέραν τη διαλειτουργικότητας πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη βούληση και θέληση συνεργασία από τα κράτη-μέλη. Και να διαβεβαιώσουμε βέβαια ότι όλα αυτά θα γίνουν ε, με τον πιο υπεύθυνο τρόπο από όλα τα κράτη-μέλη. Ευχαριστούμε ο κύριος Λέναρτς. Ευχαριστώ πολύ και εσάς κυρία Πρέζη καθώς και εσά, κύριε Επίτροπε καθώ βέβαια και τι ε, Υπηρεσίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την θαυμάσια τεχνική παρουσίαση που παρακολουθήσαμε χθες. Κάπου χθε το βράδυ, γύρω στι 7.30. Πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Βεβαίω η διαλειτουργικότητα είναι σημαντικό βήμα προ τα εμπρό, έτσι ώστε να γίνεται η βέλτιστη δυνατή χρήση των συστημάτων και οι πληροφορίε που διαθέτουν να χρησιμοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την ασφάλεια όλων μας. Μου άρεσε πολύ και το βίντεο κλιπ. Έλεγε κάπου ότι ίσως είναι ε, βαρετό και τεχνικό. Εμένα μου αρέσουν αυτά τα πράγματα. Δεν χρειάζεται να είναι εντυπωσιακά τα βίντεο αυτά. Ας είναι όσο βαρετό και τεχνικό θέλει, αλλά να μας βοηθεί να κάνουμε τη δουλειά και να την κάνουμε σωστά, που αυτό σημαίνει πρώτα ότι δεν θα χρειαστεί να επανεφεύρουμε τον τροχό, όπως είπε σωστά άλλωστε ο Επίτροπος. Πολλή δουλειά έχει γίνει και πολλή δουλειά γίνεται ακόμη. Μιλήσαμε για Aedias, Eurodac ή FCS και όλους τους σχετικούς φακέλους που είτε πέρασαν και από εμά εδώ ή τα έχουν ακόμα άλλοι αρμόδιοι στα γραφεία τους και δεν ήταν πάντοτε εύκολο να τα περάσουν από το Κοινοβουλίο, όμως μπορέσαμε να καταλήξουμε σε πολύ επικοδομητικές συμβιβαστικές λύσεις. Μιλήσαμε για την διαλειτουργικότητα των συστημάτων, η DPS λέει ότι αν θέλουμε να τα κάνουμε σωστά τα πράγματα χρειαζόμαστε νέα νομική βάση για πολλά από τα συστήματα αυτά. Αυτό είναι κάτι προς το οποίο κινούμεθα. Υπάρχει τρόπος ε, ίσως να υπάρξει μια πιο οριζόντια προσέγγιση ή θα αντιμετωπίσουμε στους επόμενους μήνες τα όσα συζητήσαμε έως τώρα έτσι ώστε να παραμείνουμε μέσα στα πλαίσια της διαλειτουργικότητας. Δεύτερο, η μέχρι τώρα προσέγγιση για να εξασφαλίσουμε ότι οι ιδέες που διαθέτουμε λειτουργούν στην πράξη, έχουν σχέση με την ποιότητα των δεδομένων και ίσως να μην παρακολούθησα καλά, κάπου, κάπου μιλήσατε για ένα data warehouse, για μια αποθήκη δεδομένων. Μπορεί να πει κάτι στην έκθεση. Και τέλος είπατε ότι οι χώρες μελή χρειάζονται εργαλεία, μηχανισμούς για να αντιμετωπίσουν την απάτη ταυτοτήτων στις επικρατείες τους. Άκουσα προχθές, την προηγούμενη εβδομάδα, τις ειδήσει από τις κάτω χώρες. Χρειάζεται λοιπόν όχι μόνο να διαθέσουμε στις χώρες μέλη τα μέσα για την αντιμετώπιση, αλλά και να τα χρησιμοποιήσουν τα μέσα αυτά. Τα δακτυλικά αποτυπώματα στα διαβατήρια, ήδη από το 2009, χάρη στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, περιλαμβάνονται για να αντιμετωπιστούν ε, ε, να αντιμετωπιστούν απάτες ταυτότητα αλλά δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ στι 100 χώρε. Πρέπει να βρεθεί τρόπο, μηχανισμοί, ώστε τα ε, εργαλεία που διαθέτουμε να χρησιμοποιούνται πράγματι στην πράξη. Ο κύριος Άλμπρεχτ των Πρασίνων, συμφωνώ με πολλά από τα όσα είπατε ω τώρα και ιδίω με τον κύριο Κοέλιο, που νομίζω ότι τόνισε ιδιαίτερα την συγκεκριμένη ιδέα του όλου κόνσεπτ της διαλειτουργικότητα, γιατί μπορούμε να μιλήσουμε για διαλειτουργικότητα με πολύ διαφορετικό τρόπο ο καθένας, Χωρί να συμφωνούμε επί της ουσίας. Συμφωνώ πολύ σχετικά με το ότι υπάρχει πραγματική προστιθέμενη αξία να υπάρχει ένα σημείο διατομής, interface και τεχνική διαλειτουργικότητα των συστημάτων, ώστε τα δεδομένα να μπορούν να ταλάσσονται με ταχύτητα και να χρησιμοποιούνται με αποτελεσματικό τρόπο όσα δεδομένα είναι διαθέσιμα. Από την άλλη μεριά συμφωνώ με το γεγονός ότι αυτό θα πρέπει να γίνεται χωρίς να αλλάξει η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων. Αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό, διότι για να υπάρξει νομιμοποίηση για τις δράσεις αυτές, αυτή χρειάζεται, έτσι ώστε πράγματι το μήνυμα να είναι μήνυμα εμπιστοσύνη ότι υπάρχουν καλύτερα δεδομένα και όχι ότι αναζητούμε νομικέ βάσει. Θα ήθελα να ακούσω επίσης σχετικά με περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις ιδέες που κατατίθενται γιατί η διατομή έρευνας είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που ακούστηκε εδώ συστήματα δηλαδή που συνομιλούν μεταξύ τους γιατί αυτό βεβαίω είναι πάλι κάτι άλλο. Και τα συστήματα έχουν διαφορετικούς σκοπούς. Συστήματα και τράπεζες δεδομένων έχουν και διαφορετικά data set. Και εμείς ως νομοθέτες έχουμε αποφασίσει ότι ένα συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων εξυπηρετεί ένα συγκεκριμένο σκοπό και άλλο σύνολο δεδομένων άλλο σκοπό. Γι' αυτό και χρειάζεται να ισχύουν οι αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητα, Αν όμως τα συστήματα συνομιλούν μεταξύ τους καθημερινά, χωρίς ξεκάθαρη ένδειξη για το πώς θα πρέπει να γίνεται αυτό και το εάν θα υπάρχουν οι αναγκαίες, τα αναγκαία εχέγγυα, υπάρχει ε, κίνδυνος ε, να υπονομευθούν οι, ε, δια, οι ε, διατάξεις αυτές της ασφαλείας. Ευχαριστώ κυρία Βερζιά. Ε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ επίσης για όλους τους παρεμβάντες σήμερα καθώς και χθες που μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε καλύτερα τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν έχω καταλάβει καλά, η διαλειτουργικότητα θα καταλήξει στην δημιουργία μιας διατομής, μιας interface, δηλαδή που θα επιτρέπει σε κάθε ένα από τα συστήματα να υπάρχει πρόσβαση σε αυτό δηλαδή με ένα κλικ να προσεγγίζουμε πληροφορίες σχετικά με ασφάλεια, διαχείριση των συνόρων και καταπολέμηση της ε, παράνομης μετανάστευσης. Επομένως, τρεις στόχους που μέχρι τώρα ήταν ξεχωριστοί. Θέλω να μάθω λοιπόν πώς θα επιτευχθεί ε, να γίνονται σεβαστές οι αρχές της αναγκαιότητας και αναλογικότητας εν προκειμένου. Και σε ό,τι αφορά τα συστήματα, αλλά και σε ό,τι αφορά την πρόσβαση των διαφόρων αρχών στα διάφορα συστήματα. Διότι αναλόγως με τα συστήματα η πρόσβαση από πλευρά αρχών δεν είναι ίδια και οι διάφορες αρχές δεν έχουν πρόσβαση στις ίδιες πληροφορίες αναλόγως με το σύστημα. Μας λέτε ότι δεν θα γίνουν νέες συλλογές δεδομένων μέσω της διαλειτουργικότητας. Ωραία. Αλλά όταν εξετάζει κανείς τις διάφορες ε, μεταρρυθμίσεις για το CIS, CIS Retour, OAS, ETIAS, όλα αυτά τα συστήματα δηλαδή, έχω την αίσθηση ότι τα πλήθη νέων προφοριών δεν σταματούν να αυξάνονται. Αυτό δεν είναι διαλειτουργικότητα, αυτό είναι τροποποίηση των διαφόρων συλλό. Το αποτέλεσμα όμως εν τέλει είναι το ίδιο και ιδίω διότι δημιουργείται το CIS Return και εκεί ορίζεται ένα έγκλημα το οποίο είναι η παράνομη διέλευση των συνόρων, αδίκημα δηλαδή, και για τα αδικήματα τα οποία μπορούν να διώκονται στα πλαίσια του CIS, αυτά βαρύνονται με ένα έξτρα δίκημα που αφορά το πρόσωπο το οποίο είναι ύποπτο να... Μα πώς θα οριοθετηθεί εδώ το πλαίσιο, Σε ό,τι αφορά την ποιότητα. Διερωτώ με, όπως και άλλοι, σχετικά με την ευθύνη των χωρών μελών για το θέμα αυτό. Το σύστημα που έχουμε τώρα προβλέπει ότι οι χώρες δίνουν τις πληροφορίες. Πώς λοιπόν βελτιώνεται η ποιότητα όταν δημιουργείται ένα interface και ποιος είναι ο έλεγχος επί των πληροφοριών που χορηγούν οι χώρες μέλη. Και η τελευταία μου ερώτηση, και θα σταματήσω κυρία Πρόεδρε, τι γίνεται με την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων όταν δεν γνωρίζουμε ποιο είναι το ποιόν των εισαγωμένων πληροφοριών και δεδομένων. Και προστασία των δεδομένων χρειάζεται αν υπάρξει ένα σφάλμα ας πούμε στην εισαγωγή στο σύστημα. Και για να το βλέπω θετικά θα πω και λίγο περισσότερο. Το σύστημα διαλειτουργικότητας πώς θα επιτρέπει την διευκόλυνση της διόρθωσης των ενδεχομένων σφαλμάτων που έχουν παρισφρήσει το σύστημα. Εάν καν αυτό είναι δυνατό. Ευχαριστώ κυρία Στίβενς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους δύο ομιλητές για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση σε ό,τι αφορά την διαλειτουργικότητα. Οπότε κατάλαβα, η ομάδα πραγνωμών υψηλού επίπεδου και η τελική έκθεση εξετάζουν ακριβώς αυτή τη διαλειτουργικότητα προκειμένου με μία ε, απλή αναζήτηση θα έχουμε διαφορετικά αποτελέσματα στην ίδια οθόνη. Ε, περιμένω με ενδιαφέρον ε, το προσχέδιο πρότασης της Επιτροπής στα τέλη της χρονιάς. Όμως, ποιες είναι οι τεχνικές προδιαγραφές ε, για να πετύχουμε αυτή τη διαλειτουργικότητα διαφόρων βάσεων δεδομένων. Υπάρχουν οι απαραίτητε τεχνικέ εξελίξει για να γίνουν όλα αυτά με ασφαλή, αξιόπιστο και οικονομικά αποδοτικό τρόπο. Η διαλειτουργικότητα είναι σημαντική και σε ό,τι αφορά τη βιομετρική ταυτοποίηση. Υπάρχουν δυσκολίες προς το παρόν με ε, τα δυσανάγνωστα ονόματα ή κάποιες φορές και με τις ταυτότητες. Οπότε είναι πολύ καλό όλο αυτό να γίνει με τα βιομετρικά στοιχεία. Όμως, κύριε Κίνγκ, ε, προβλέπετε ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα για την ε, θέσπιση ενός τέτοιου συστήματος. Κάποιες ε, προτάσεις, ερωτήσεις έχω ακόμα. Στρέφω όμως στο διερμηνέα της αγγλικής νοηματικής. Ποια Ποιε είναι οι πιθανές απτές υλικέ και άλλες βελτιώσεις μπορούμε να πετύχουμε σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματο, τη διαχείριση συνόρων, των εξωτερικών συνόρων, τη διαχείριση της ε, νόμιμη και παράτυπη μετανάστευση. Μετά, η εφαρμογή οποιασδήποτε πρόταση ε, θα ωφελήσει όλα τα κράτη-μέλη με τον ίδιο τρόπο. Πόσο ετερογενή θα είναι η ε, υλοποίηση της πρότασης από τα κράτη-μέλη και θα υπάρξουν κράτη-μέλη που θα έχουν προβλήματα, προβλήματα ε, πρακτικής εφαρμογής και πώς θα αντιμετωπιστούν. Θα αυξηθούν οι κίνδυνοι ε, διαδικτυακής ε, επίθεσης. Ποια επιπρόσθετα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα μπορεί να υιοθετήσει ο Ιουλίζα και από ποια κράτη-μέλη. Υπάρχουν σαφείς δεσμοί μεταξύ προβλημάτων και λύσεων που προτείνονται από την ε, ομάδα ψηλοεπιπέδου. Οι στόχοι αυτών των προτάσεων ξεκαθαρίζονται σε σχέση με τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί. Και τέλος, μπορούν να υπάρξουν ε, και παρενέργειε ή ανεπιθύμητε επιπτώσει ε, αυτών των συστάσεων τη ε, ομάδα υψηλού επίπεδου ε, ω προ τα θεμελιώδη δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών. Για παράδειγμα, στον ιδιωτικό βίο και στην προστασία δεδομένων. Πώς μπορεί να μετριαστεί αυτός ο κίνδυνος ανεπιθύμητων παρενεργειών μέσω τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων σε επίπεδο κρατών μελών ή και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία και κύριος Φως. You didn't ask for Ζητήσατε το λόγο, έτσι δεν είναι. Α, καλώς τότε, η κυρία Γκόμες. Νομίζω μιλούν και οι δύο ταυτόχρονα. Κυρία Γκόμες, είχαμε και χθε το ίδιο θέμα. Δεν θέλω να σας ρωτήσω για τη διαλειτουργικότητα, αφού τα είπαν οι συνάδελφοί μου. Διαλειτουργικότητα σημαίνει και βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων προσώπων που διέρχονται τα σύνορά μας. Αλλά έχουμε όμως και μέρη, τμήματα που δεν υπάρχει έλεγχος ή πάντως ε, είναι ελαττωματικός. Και δεν υπάρχει και καθόλου διαλειτουργικότητα. Για παράδειγμα, ιδιωτικά αεροσκάφη που προσγειώνονται σε μικρά αεροδρόμια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση προερχόμενα από τρίτες χώρες και ουδής ενδιαφέρεται να συλλέξει δεδομένα περί πληρωμάτων, επιβατών, φορτίων. Μπορεί τα φορτία αυτά να είναι από όπλα και ναρκωτικά μέχρι ανθρώπους ή χρήματα. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Μην το παρακάνουμε με τη διαλειτουργικότητα όταν ταυτόχρονα Α, και το PNR δεν λειτουργεί εκεί, έτσι είναι. Ενώ λοιπόν άνθρωποι με λεφτά, είτε δικά τους λεφτά, είτε των εγκληματικών τους οργανώσεων, στην ουσία βγάζουν τη γλώσσα σε όλη τη δουλειά που κάνουμε εδώ ε, με την ε, μανία αυτή που έχουμε ελέγχου, των συνόρων. Ευχαριστώ κύριε Γκόμης. Ε, επανέρχομαι στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα. Και πρώτα η πρέσβης κυρία Κάλια. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ήθελα να τονίσω εξ υπαρχής πόσο αρμονικά συμβεί η Επιτροπή με το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο με την Επιτροπή και αυτό είναι πραγματικά αξιέπαινο. Τώρα όμως μετά από τις πρώτες αυτές ερωτήσεις των Ευρωβουλευτών μπορώ να πω ότι πολλοί εξημών των Ευρωβουλευτών συμφωνούν. Άκουσα τις ε, παρατηρήσεις σας και συμφώνησα με τη σκέψη που εκφράσατε όπως του κ. Κοέλιο. Θα μπορούσα να συμφωνήσω με ολόκληρο το κείμενο της δηλώσεώς σας. Ε, θα ήταν σαν να τα είχε πει και το ίδιο το Συμβούλιο τα πράγματα αυτά. Και βεβαίως και πολλοί άλλοι εξημών Τονίσατε και εσείς αυτό που θέλουμε να τονίσουμε και εμείς, ότι η διαλειτουργικότητα δεν είναι μαγικό ραβδάκι, μακάρι να ήταν. Μακάρι να είχαμε κάτι το οποίο θα έλυνε όλα τα προβλήματα που έχουμε αμέσως. Όμως, η διαλειτουργικότητα είναι μια απλή τεχνική βελτίωση της χρήσεως των δεδομένων. Όπως είπε και ο κ. Σκόλιο, εξυπηρετεί τον τελικό χρήστη. Κάποιο άλλο είπε, ήταν και πολλοί ομιλητέ δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώ ποιο, πάντω κάποιο είπε ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ των, υπάρχουν διαφορέ, μάλλον μεταξύ των χωρών μελών, δεν είναι όλε το ίδιο πρόθυμε να μοιραστούν τι προφορίες του με άλλου. Μιλείτε σε μια ιστονή, μην το λησμονείτε αυτό. Εμεί θεωρούμε ότι η διαλειτουργικότητα είναι το φυσικότερο πράγμα του κόσμου. Δεν έχουμε απολύτω κανένα ιδεολογικό πρόβλημα με τη διαλειτουργικότητα ε, δίνουμε και μεγάλη ε, προσοχή ε, στην φύλαξη των συνόρων μέσω των μηχανισμών αυτών. Έχω τώρα και ένα άλλο παράδειγμα από άλλο τομέα που έχει όμως σχέση. Γνωρίζετε ότι από τα μεγαλύτερα προβλήματά μας είναι στη Μεσόγειο, στην κεντρική Μεσόγειο αλλά και στην ανατολική μεριά της Μεσογείου όπου προσπαθούμε να φτιάξουμε μια καλύτερη συνοριοφυλακή με διάφορες επιχειρήσεις που λειτουργούν εκεί. Operations δηλαδή. Και ε, με σημαντική ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ ε, στρατιωτικών, αστυνομικών και πολιτικών αρχών. Και αυτό είναι το στοιχείο εμπιστοσύνης ή έλλειψης εμπιστοσύνης. Και βλέπω ότι υπάρχει βελτίωση. Δημιουργείται μεγαλύτερη, βαθύτερη εμπιστοσύνη μεταξύ των χωρών μελών καθημερινά και με όλες αυτές τις τεχνικές λύσεις οι οποίες θα βελτιώσουν την καθημερινή μας πρόσβαση και τα αποτελέσματα που αποκομίζουμε, ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε και το ψυχολογικό μέρος αλλά και τις τεχνικές ε, απαιτήσει. Κάποιος μίλησε για την EU-LISA, για τον οργανισμό EU-LISA που είναι ένας οργανισμός που έχει ως σκοπό να προβληματίζεται και για την ποιότητα των δεδομένων. Έχουμε συνεργαστεί μαζί τους, υπάρχει ένα είδος οδικού χάρτη για τη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων. Η διαλειτουργικότητα δυστυχώς δεν θα λύσει όλα τα προβλήματα, όμως θα λύσει ένα ελάχιστο των προβλημάτων που είναι οι απαιτήσει του 21ου αιώνα. Και όταν κάποιος μίλησε για συνομιλία των συστημάτων μεταξύ των. Φοβούμαι ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο σημείο αυτό. Τα συστήματα δηλαδή που συνομιλούν μεταξύ των χωρί την δική μα παρέμβαση θα σήμαινε τεχνητή νοημοσύνη, η οποία είναι βεβαίω στην ατζέντα μα και ίσω μάλιστα να ενσκύψει ταχύτερα από ό,τι πιστεύουμε, αλλά για την ώρα μιλούμε ακόμη για ανθρώπου οι οποίοι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα, στι πληροφορίε στην βάση την οποία έχουμε θεσπίσει και συμφωνήσει εμείς. Η Επιτροπή νομίζω θα εξηγήσει την πρόταση και το περιεχόμενό της. Ευχαριστώ κυρία Πρέσβη. Σεις τώρα κύριε Επιτροπέ, ορίστε. Ευχαριστώ, αλλά και για τις ερωτήσεις ευχαριστώ. Να βλέπουμε τι ενδιαφέρον υπάρχει. Και στη συνέχεια των όσων είπε η κυρία Πρέσβης Ναι, είναι θέματα τεχνικά, είναι θέματα καμιά φορά βαρετά και καμιά φορά ακατάληπτα. Οπότε να μία πρόκληση. Να ένα από τα προβλήματα είναι το να τα εξηγήσουμε, να εξηγήσουμε τι κάνουμε, γιατί δεν κάνουμε. Δεν πρόκειται να λύσουμε όλα τα προβλήματα σήμερα με τις προτάσεις για την διαλειτουργικότητα ούτε ποτέ θέλαμε να πούμε ότι σήμερα αυτά θα λυθούν με τις προτάσεις για τη διαλειτουργικότητα. Απλώς θέλουμε να εκμεταλλευτούμε όσο γίνεται περισσότερο τις βασιστομένο που έχουμε. Όχι κύριε Γκρεγκόμης, δεν θα μπορέσουμε να άρουμε όλα αυτά τα κενά που επισημάνατε. Αντίθετα, εσείς με το έργο σας θα μας βοηθήσετε σε σχέση με αυτά τα κενά και είπαμε να αλλάξει η λειτουργία των υπαρχουσών βάσεων δεδομένων, δεν πρόκειται να φτιάξουμε νέες ε, βάσεις δεδομένων. Όχι, δεν θα ε, γίνει συλλογή περισσότερων ε, ε, στοιχείων περισσότερων δεδομένων. Υπάρχουν διαχωριστές δηλαδή αποφάσεις για την κάθε ε, βάση δεδομένων και εσείς κάθε φορά ε, με την νομοθετική διαδικασία ελέγχεται. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι όταν όλα έχουν συμφωνηθεί σε σχέση με την συλλογή των δεδομένων οι πληροφορίες που συλλεγεί να χρησιμοποιούν με αποτελεσματικότητα και πολλοί από εσά, όπως ο κύριος Λόπες Αγκουιλάρ, η κυρία Ζήπελ επίσης, Είπατε ότι ναι, όλα αυτά ενδιαφέροντα, αλλά τι γίνεται με τα κράτη-μέλη, τι γίνεται με τα κενά σε σχέση με το πώς διαχειριστούνται τις πληροφορίες στα κρατημέλη. Ναι, και εδώ έχετε δίκιο και θα συνεχίσουμε, συνεργαζόμαστε μαζί σας και σε αυτό το μέτωπο. τι τι λειτουργικότητα έχουν να κάνουν με τις βάσεις δεδομένων, τις πανευρωπαϊκές και σε σχέση με το τι θα κάνουμε ως προς τα κρατημέλη τα έχουμε ήδη συζητήσει και θα τα ξανασυζητήσουμε. Θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε την πλήρη εφαρμογή, την πλήρη υλοποίηση των όσων ε, συμφωνούμε να χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που έχουμε και για τις ε, διαδικασίες η παραβάση θα πρέπει να λάβουν τις ευθύνες στο κράτη-μέλη και όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών, χρηματοδότηση, άριστες πρακτικές, ε, εκπαίδευση. Θα πρέπει να βρισκόμαστε και να τροποποιούμε ό,τι τυχόν χρειάζεται, γιατί είπαμε ότι στην ε, καρδιά των προσδοθειών μας είναι το σύστημα πληροφοριών Σέγγεν. Άρα θα πρέπει το σύστημα αυτό να θωρακιστεί, να αναβαθμιστεί και όπως είπαμε θέλουμε να θεσπιστεί η υποχρέωση ε, ανταλλαγής πληροφοριών για την αντιμετώπιση της ε, τρομοκρατίας. Να αξιοποιήσουμε τεχνολογία, να προωθήσουμε τη χρήση των ε, automatic, των αυτόματων loaders των δεδομένων και επομένως όλα αυτά να γίνονται αποτελεσματικά αλλά και γρήγορα. Προς τα εκεί θα πάνε οι προσπαθειές μας αλλά επίσης για τα συστήματα που υπάρχουν αυτό που θέλουμε είναι να τα αξιοποιήσουμε περισσότερο. Οπότε και Έτσι θα ενθαρρύνουμε την ανταλλαγή πληροφορών των κρατών μελών. εδώ μιλούμε για ένα αρετό κύκλο. Για να αυτές οι κοινέ πλατφόρμες είναι πιο αποτελεσματικές, πιο χρήσιμες και οι υπηρεσίε μεταναστές, οι υπηρεσίε αλλοδαπών, οι συνοροφίλε, όλοι αυτοί, εάν αυτοί τώρα ωφεληθούν από όλα αυτά, ή τότε τα κράτη-μέλη θα έχουν κίνητρο ανταλλαγή πληροφοριών. Το είπαμε, το έχουμε ξαναπεί και πριν από σήμερα. Αλλά έτσι θα αποδώσει η προσπάθεια. Τώρα για τη διαλειτουργικότητα υπήρξε κάποια ερώτηση που αφορά και την πρότασή μας. Εμείς συνεχίζουμε να μελετούμε κάποιες απόψεις, δηλαδή το πώς ε, θα προωθήσουμε τις ιδέες σας, τις χθεσινοβραδινές. Ε, τα συζητούμε με τους εμπειρογνώμονες, θα τα συζητήσουμε άλλη φορά. Όχι, σήμερα δεν είμαστε έτοιμοι. Ε, και δεν προτείνουμε πάντως νέες νομικές βάσεις για τα υπάρχοντα νομοθετήματα. Έχουμε προσέγγιση οριζόντια. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε κάποιες αλλαγές στις ισχύουσες διαδικασίες για τα συστήματα που υπάρχουν. Εκεί γι' αυτό θα πρέπει και εμείς εντελεχώς να τα συζητήσουμε όσον αφορά την ε, εφαρμογή της πρότασης που θα παρουσιάσουμε. Θέλουμε να έχουμε διαφάνεια. Δεν θα αλλάξει τίποτα σε σχέση με τα δικαιώματα πρόσβασης. Ποιος δικαιούται να έχει πρόσβαση σε κάποια πληροφορία. Αυτό όμως που θέλουμε να διερευνηθεί και ακόμα δεν έχει παγιωθεί λύση το τι θα κάνουμε είναι το αν μπορούμε να βελτιάσουμε κανόνες και διαδικασίες για το πώς ασκούνται τα δικαιώματα πρόσβασης στις πληροφορίες. Δηλαδή, χρειάζεται πάντοτε να υπάρχει προτέρα διαβούλευση πριν κανείς κάνει κάποιο έλεγχο σε κάποια άλλη βάση δεδομένων, ίσως ε, ε, υπό κάποιες περιστάσεις αυτό θα πρέπει να γίνεται πιο γρήγορο και να μην περάσει από μια τέτοια διαβούλευση. Δηλαδή όχι κανείς να μπορεί να δει πληροφορίες που δεν δικαιούτο, αλλά να μπορεί να συμβουλευτεί τα σχετικά στοιχεία πιο γρήγορα, με πιο σύντομη διαδικασία. Αυτά θέλουμε να συζητηθούν. Εάν τώρα, το οποίο είναι και πιθανό, να έχουμε κάποια πρόταση για συντόμευση των διαδικασιών με το σύστημα HIT no HIT στο οποίο αναφέρθηκε η κυρία Γκρισμπέκ εάν λοιπόν γίνει αυτό τότε θέλουμε να έχει καταστεί σαφές ότι αυτή μας η πρόταση θα γίνεται υπό την επιφύλαξη των όσων σήμερα ισχύουν ως προϋποθέσεις πρόσβασης στις πληροφορίες. Το κείμενο το σχετικό θα είναι σαφές ότι για να συνεχίσει κανείς ε, την έρευνα αφού βρήκε κάτι, αφού έκανε ένα hit στα στοιχεία θα πρέπει όποιος τα κάνει αυτά να δικαιούται την πρόσβαση στις επιζητούμενες πληροφορίες αν χρειάζεται φερρυπίν δικαστική άδεια, άλλου είδους ε, έγκριση, άδεια, ό,τι προβλέπουν ε, τα ε, νομοθετήματα που προβλέπονται, που υπάρχουν τέλος πάντων. Δεν θα αλλάξουν τόσο προβλήματα για τα σχετικά δικαιώματα τώρα. Όσον αφορά την αποθήκευση των δεδομένων που κάποιος το ανέφερε, θα διαπιστώσετε ότι αυτό καλύπτεται από την πρόταση Λίσα. Δεν το ξεχάσαμε το θέμα. Είναι τμήμα της προσπαθίας μας για αναβάθμιση της ποιότητας των δεδομένων και της πρότασης Λίσα. Τώρα όσον αφορά ε, κάποιο είδου παραπλάνηση που ανέφερε ο κύριος Άλμπριχτ. Ναι, όντως δεν θα πρέπει με τη φρασιολογία μας να παραπλανούμε. Όταν λέμε να μιλούν τα συστήματα μεταξύ τους, το λέμε έτσι, διότι προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να εκφράσουμε την επιθυμία μας να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο των πολλαπλών ταυτοτήτων που είναι κατοχρημένα στα διάφορα συστήματα. Και όπως είπα, Έχουμε προτάσεις για αυτό το μητρό δεδομένων οπότε θα αποκλειστεί η περίπτωση το να έχει κάποιου διαφορετικές ταυτότητες χρησιμοποιώντας τα πολλά συστήματα χρησιμοποίησα αυτή τη γλώσσα για να σας παραπλανήσω αυτό εννοούσα δεν ήθελα να εννοήσω κάποιο είδου συνεχή διάδραση μεταξύ των συστημάτων ούτω ώστε να παρακάμψει κανεί του κανόνες για την προσβασιμότητα. Τίποτα από όσα θα προτείνουμε δεν θα παρακάμπτει τα όσα προβλέπονται. Ελπίζω ότι ε, έστω και εν μέρει σας καθησύχασα. Κορατσαμπίλ, να έχετε δίκιο. Πρέπει να τα πούμε ξεκάθαρα όποτε εξηγούμε ότι με τίποτε δεν θέλουμε να ε, παρέμβουμε στα του ιδιωτικού βίου. Είπαμε για διαφορετικέ ταυτότητε, είπαμε για τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών. Αυτά όλα θα πρέπει να ισχύσουν. Θέλουμε να έχουμε ε, περισσότερη υποστήριξη στο έργο των συνοροφυλάκων, των διοικητικών αρχών, γενικότερα με τι βάσει δεδομένων. Ελπίζω κάπω σα βοήθησε και την επόμενη φορά που θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση και να συζητήσουμε επί τη βάση συγκεκριμένων μα προτάσεων. Οπότε και θα μπορέσω να απαντήσω περισσότερε από τι ερωτήσει Φερρυπίν τη κυρία Στίβεν για το ποιο είναι ο κίνδυνο να μην υπάρχει ωφέλεια ή ποιε θα είναι οι ωφέλειε. Θα μπορέσουμε να έχουμε την αξιολόγηση που θα συνοδεύει την πρότασή μας. Και βέβαια θα έχουμε και το σχετικό χρονοδιάγραμμα. Και σας ευχαριστώ την προσοχή σας. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Θα δώσουμε το λόγο στον ε, κύριο Βιβορόφσκι, αναπληρωτή επόπτη του EDPS, για να μας παρουσιάσει την πρόσφατη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σχετικά με το συνεχιζόμενο έργο στον τομέα της ε, διαλειτουργικότητας στην ε, ασφάλεια και δικαιοσύνη possible. Okay. okay. Well, Ωραία λοιπόν. Έχουμε 15 λεπτά στη διάθεσή μας. Άντε 20. Να κλέψουμε για ένα πεντάλεπτο από το επόμενο θέμα. Παρακαλώ να μην ξεπεράσει τα 10 λεπτά για να γίνει και μια συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, σα ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τη δυνατότητα που μου δίνετε να σας μιλήσω για το ζήτημα της διαλειτουργικότητας ε, των συστημάτων που χρησιμοποιούνται στον τομέα της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Θέλω σήμερα να σας παρουσιάσω ε, τα βασικά μηνύματα του εγγράφου προβληματισμού που έχει ε, υπογράψει ο Ευρωπαίος Επόπτης Ζωβάνι Βουταρέλη πριν από μερικές ημέρες. Η DPS ως ε, αρχή προστασίας δεδομένων των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων αναγνωρίζει τη διασύνδεση των ε, δημοσίων πόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως την φυσιολογική εξέλιξη των πληροφορικών συστημάτων. Είμαστε βέβαιοι ότι και οι άλλες διαστάσεις της διαλειτουργικότητας των ηλεκτρονικών ε, υπηρεσιών με τα επιμέρους συστήματα σίγουρα θα τύχουν ε, ενδελεχούς εξέτασης όταν θα ε, αναλύσουμε τις λύσεις και από τους αρχιτέκτονες του συστήματος, τους χρήστες, τον νομοθέτη και σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο. Γνωρίζουμε ότι επί της αρχής σκοπός είναι η ανάπτυξη αποτελεσματικής και αποδοτικής συνταλλαγής πληροφοριών προκειμένου να υπάρχει η σωστή πληροφόρηση την σωστή στιγμή. Έτσι ξέρουμε ότι η συζήτηση που κάνουμε σήμερα είναι ένα μόνο βήμα ε, στην ε, μακρά αυτή συζήτηση για την ε, αξιοποίηση των δεδομένων που ε, διατηρεί η δημοσιοδιοίκηση. Αυτό δεν είναι ε, προκαλεί έκπληξη σε εμά, ούτε είναι κάτι που φοβόμαστε. Εμείς θεωρούμε ότι η διαλειτουργικότητα μπορεί να μας βοηθήσει να καλύψουμε ανάγκες των αρμόδιων αρχών αξιοποιώντας ε, τα πληροφορικά συστήματα μεγάλης κλίμακας και να περιορίσουμε το ε, κόστος αυτών των συστημάτων. Επίσης, ε, μπορεί να ωφελήσει την προστασία δεδομένων Έχουμε και παράδειγμα τα διασυνδεδεμένα πληροφορικά συστήματα που έχουν συναφείς στόχους και περιέχουν παρόμοια ή ταυτόσημα δεδομένα. Ε, μπορούμε έτσι με την ανταλλαγή στοιχείων να περιορίσουμε τον όγκο και το κόστος ε, των πληροφορικών συστημάτων. Εισάγεται έτσι και το λεγόμενο privacy by design σε όλη τη συζήτηση της διαλειτουργικότητας στον τομέα της ασφάλειας και της δικαιοσύνης και σε όλο αφήγημα των πληροφορικών συστημάτων των 21 ου αιώνα. Ενδέχεται έτσι να υπάρξει και αλλαγή στην επεξεργασία των ε, προσωπικών δεδομένων, γι' αυτό ενδεχομένως να χρειαστούν και τροποποιήσει της νομικής βάσης, ε, και πάντα με σεβασμό προ τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ιδίω ε, νέα ή τροποποιημένη επεξεργασία δεδομένων θα πρέπει να προσδιορίζεται ξεκάθαρα στα σχετικά νομικά μέσα και να είναι αναλογική ε, σε σχέση με τους ξεκάθαρους στόχους. Για να έχουμε περισσότερες πληροφορίες για την ευρωπαϊκή νομοθετική πρόταση, θεωρούμε ότι μία πλήρης ε, μελέτη αντικτύπου της διαλειτουργικότητας για τα μελώδη δικαιώματα και για την προσωπικό βίο και την προστασία δεδομένων είναι κάτι κέρια σημασία. Έχουμε ακούσει ήδη το έργο της ομάδας υψηλού επίπεδου και έχουμε συμμετάσχει σε αυτές τις ε, προσπάθειες. Και τα συμπεράσματα της έκθεσης της DPS ελήφθησαν υπόψη από την ομάδα της Ωστόσο, θα πρέπει να έχουμε κατά νου αυτές οι τρεις προτάσεις που έχουν τεθεί επιτάπητος και έχουν υιοθετηθεί από το Συμβούλιο. για τα βιομετρικά στοιχεία, την κοινή πύλη και το κοινό αποθετήριο. Είναι μόνο η αφετηρία της συζήτησης και για άλλες υπηρεσίες που θα προτεθούν στο μέλλον. Γιατί όσο περισσότερες επιλογές έχουμε στο μέτρο της λειτουργικότητας και της διασύνδεσης, τόσο περισσότερες ε, εφαρμογές θέλουμε να αξιοποιήσουμε. Να σταθώ σε ορισμένα σημεία για τη διαλειτουργικότητα και τις προσδοκίες μας. Αναφέρεται η διαλειτουργικότητα ως η δυνατότητα διαφορετικών πληροφορικών συστημάτων να επικοινωνούν μεταξύ τους. Συχνά θεωρείται μόνο τεχνική έννοια, όμως εμείς πιστεύουμε ότι δεν μπορούμε να το αποσυνδέσουμε από το θέμα της αναγκαιότητας της ανταλλαγής πληροφοριών, της ε, πολιτικά επιθυμητής ε, ανταλλαγής ε, δεδομένων και το καθεξής. Πάντα λοιπόν πρέπει να προκύπτει από έναν πολιτικό διάλογο και χαιρόμαστε που ξεκινάει τώρα. Να επενθυμίσουμε την έννοια της διαλειτουργικότητας με τις διάφορες προεκτάσεις της ε, στη συζήτηση ε, για τη δημόσια διοίκηση. Εκεί πολύ σωστά αναφέρεται ότι η διαλειτουργικότητα είναι η ικανότητα των οργανώσεων να έρχονται σε επαφή για ε, αμοιβαία αποφελή στόχους με ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσης μεταξύ των οργανώσεων. Όλα αυτά θα πρέπει να τα έχουμε κατά νου. Όταν εξετάζουμε την ε, σημασιολογία της διαλειτουργικότητας που ανέφερε η κυρία Σίπελ, ότι με τον ίδιο ορισμό θα πρέπει να έχουμε λοιπόν ε, το ίδιο νόημα, την ίδια ερμηνεία σε όλες τις χώρες και όλα τα συστήματα οργανωτική διαλειτουργικότητα και η νομική διάσταση. Παρατηρούμε ότι για να καταστεί δυνατή η ε, ανταλλαγή πληροφοριών, αυτό αποτελεί μοχλό ανάπτυξη και περαιτέρω ανταλλαγή. Όσο περισσότερε δυνατότητε έχουμε, τόσο περισσότερα πετυχαίνουμε λοιπόν. Αυτό ανέφερε και ο Επίτροπο Κίνγκ προηγουμένω. Η διαλειτουργικότητα λοιπόν καταρχήν ε, καθιστά πιο αποτελεσματικούς ε, τους υφιστάμενου κανόνες. Όμως, για παράδειγμα, το ευρωπαϊκό, η ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης που θέλει ε, να θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βοηθήσει τις αστυνομικέ αρχές να κάνουν αναζητήσεις σε πολλά, πολλές βάσεις ταυτόχρονα και όχι σε κάθε μία ξεχωριστά. Αυτό σημαίνει ότι οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται κατά αυτόν τον τρόπο θα είναι περισσότερες από ό,τι σήμερα. Δεν είμαι σίγουρος αν τελικά δεν θα έχουμε περισσότερες βάσεις δεδομένων ή επιπρόσθετες πληροφορίες. Χρειάζεται λοιπόν ε, η συνέργεια, αλλά που μπορεί να οδηγήσει και σε νέες πληροφορίες. Κατανοούμε ταυτόχρονα ότι τώρα ή στο μέλλον η Επιτροπή θέλει να παρατείνει τις δυνατότητες ε, ανταλλαγής ε, των δεδομένων. Η μελέτη αντικτύπου μιλάει για τον αντίκτυπο της ε, αξιοποίησης βιομετρικών στοιχείων. Αντίστοιχα, μπορεί να υπάρχουν και άλλα στοιχεία, ονόματα, ε, ημερομηνίε γέννηση που μπορούν να υπάρχουν στι βάσει δεδομένων και την ε, συνδεδεμένη του ε, χρήση. Αυτό μπορεί να επιτρέπει την ε, ταυτοποίηση ε, με αριθμητικά αλλά και βιομετρικά στοιχεία. Αυτό που μόνο του δεν είναι κακό. Είναι ένας από τους στόχους που θέλουμε να πετύχουμε, όμως πρέπει να έχουμε κατά νου ότι ε, έτσι δημιουργούμε νέα πληροφορία. Κάποιες φορές οι αρχές προστασία δεδομένων επικρίνονται ότι είναι ότι είναι βαρετέ και λένε τα ίδια και τα ίδια. Αλλά αυτό είναι ο σκοπό μα. Αυτό είναι ο ρόλο μα. Πρέπει να είμαστε βαρετοί. Αυτό θα κάνω και πάλι και να λέω ότι τα προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να τυχάνουν ε, δίκαιη επεξεργασία για ειδικού σκοπού. Θεωρούμε λοιπόν ότι η διαλειτουργικότητα δεν θα πρέπει να είναι αυτό σκοπό αλλά πάντα να εξυπηρετεί ε, το δημόσιο συμφέρον. Η μελέτη που αρχικά αναφέρεται στον γενικό στόχο ανάπτυξη πιο ευφυών και πιο ισχυρών πληροφοριακών συστημάτων για τα σύνορα και την ασφάλεια και μετά αναφέρει και άλλους πιο ειδικούς σκοπούς. να διευκολύνει το έργο των αξιωματούχων και την εύκολη πρόσβασή τους στις πληροφορίες θα διευκολύνουμε την ε, πρόσβαση των αρχών επιβολής του νόμου ε, σε βάση δεδομένων όταν αυτό είναι απαραίτητο για την διαρεύνηση και δύο ποινικών αδικημάτων και τέλος αντιμετώπιση λύσεων ε, για την ανείχνευση και αντιμετώπιση περιπτώσεων απάτης. Η, γενικούς, γενική λοιπόν στόχη της αστυνομικής έρευνας δεν ταυτίζονται πάντα με το δημόσιο συμφέρον. Για παράδειγμα, δυνάμει του άρθρου 52 της Χάρτας. Ούτε εξυπηρετούν τους σκοπούς επεξεργασίας δεδομένων βάσει του σχετικού ε, νομικού πλαισίου. Καλούμε λοιπόν την Επιτροπή να ξεκαθαρίσει ε, τους σκοπούς ε, των στόχων επεξεργαστεδομένων δεδομένων γιατί μπορεί να είναι χρήσιμη σαν διαδικασία, αλλά τελικά δεν μπορούν να καταναήσουν ενδιαφερόμενοι ποια δεδομένα τους τυχάνουν επεξεργασίες και για ποιους σκοπούς ή ποιες μπορεί να είναι συνέπειες. Να υπενθυμίσω ότι στο επίκεντρο της συζήτησης για τη νέα συμφωνία με τις ΗΠΑ ε, για το Privacy Shield η ομάδα εργασίας του άρθρου 29, στην οποία συμμετέχουν όλες οι αρχές προστασίας δεδομένων, έχει καταρτήσει έναν κατάλογο απαιτήσεων ε, για την προστασία δεδομένων. Οι αρχές λοιπόν έχουν διαμορφώσει ε, τις ευρωπαϊκές ε, δικλείδες ασφαλείας και στη συνέχεια έχουν ανακληθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ε, σε συγκεκριμένες υποθέσεις όπως το PNR με τον Καναδά. η επεξεργασία θα πρέπει να βασίζεται σε σαφείς, ακριβείς και προσβάσιμους κανόνες και θα πρέπει η επεξεργασία να είναι απαραίτητη και αναλογική. Κλείνοντας, να παριθμίσω τα πιο σημαντικά τμήματα των συστάσεών μας προς τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα σε ό,τι αφορά την ε, πρακτική χρήση της διαλειτουργικότητας. Είμαστε υπέρ αυτού του μηχανισμού όταν εφαρμόζεται με έναν ε, κατάλληλο τρόπο που να συμμορφούνται με τις αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας. Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την κάλυψη ορισμένων αναγκών, αλλά μπορεί και να μας ε, επιτρέψει να αποφύγουμε το, τις αλληλεπικαλύψεις συχνά θεωρείται τεχνική διαδικασία και λειτουργικότητα, όμως εμείς θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να αποφασίσουμε εάν θέλουμε να την εισαγάγουμε και ε, τι μέτρα θέλουμε να λάβουμε από νομικής άποψης. Βρισκόμαστε στην αρχή της ε, μακρόπνους αυτής της διαδικασίας και ό,τι και αν αποφασίσουμε να ε, δημιουργήσουμε αυτή τη στιγμή δεν θα καταληφθεί ποτέ. Όταν αξιοποιηθούν οι πόροι για την διασύνδεση των λύσεων, θα υπάρχουν νέες ιδέες αναπενταετία. Και σας ε, διαβεβαιώ ότι το 2020, 2022 ή και πιο νωρίς θα ξανασυναντηθούμε εδώ για να συζητήσουμε νέα στοιχεία. Μάλλον δεν πρέπει να το πω, αλλά αν δείτε μόνο το σημείωμα που δόθηκε στο Συμβούλιο του Φεβρουαρίου και αναφέρει τα πληροφοριακά συστήματα που θέλουμε να διασυνδέσουμε στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, έχουμε μία τεράστια γκάμα τέτοιων πληροφοριακών συστημάτων και θα έχουμε και άλλα ε, στο μέλλον. Και δεν λέω ότι οι αρχές προστασίας δεδομένων εν γέννη αντίκεινται ε, σε αυτή τη διαδικασία, όμως θα πρέπει να τα προσέξουμε. Τέλος, συγκεκριμένα ζητήματα διαλειτουργικότητας που θέλουμε να επιλύσουμε θα πρέπει πρώτα να τα προσδιορίσουμε στη μελλοντική νομοθεσία και ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εντοπίσει ορισμένα προβλήματα, όμως κάποιες φορές δεν περιγράφει λεπτομερώς τα ζητήματα αυτά και τις λύσεις ε, που προτείνονται σε πρακτικό επίπεδο. Τώρα, δεν ξέρω αν το πρόβλημα έγκυται στο νομικό πλαίσιο ή αν είναι τεχνικό το πρόβλημα. Και αυτό θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Και θα πρέπει να αναφέρονται οι ακριβείς σκοποί αξιοποίησης των δεδομένων. Ε, τώρα θέλουμε να κάνουμε μια πλήρη αξιολόγηση της λειτουργικότητας στα θεμελιώδη δικαιώματα, στην ε, προσωπική ζωή και την προστασία δεδομένων Όλα αυτά βέβαια θα γίνουν ε, όταν θα έχουμε και το πλήρες πλαίσιο και είμαστε διατεθειμένοι να σας δώσουμε γνωμοδότηση για αυτήν την νομοθετική διαδικασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ζίπλ. Ε, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Και τώρα άρχισε να σηκώνω το χέρι μου όταν φτάσατε στο κόστος και ότι ίσως είναι δυνατόν να μειώσετε το κόστος. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Και πρώτον, διότι ίσως την ερώτηση απαντήχα να κάνει στον Επίτροπο κύριο Κίνγκ, έχετε καμιά ιδέα σχετικά με το κόστος για να αρχίσει να λειτουργεί η διαλειτουργικότητα, διότι τα τεχνικά πρότυπα των διαφόρων σιλό είναι διαφορετικά για να υλοποιηθεί το δικαίωμα πρόσβασης καθώς και τα δικαιώματα όσων έχουν δικαίωμα να τροφοδοτούν τα σιλό με πληροφορίε Είναι λοιπόν πολύ ε, περίπλοκο το θέμα και ίσως χρειάζεται και ξεχωριστό λογισμικό αλλά και ε, μηχανήματα. Τώρα, για το ποιο έχει το δικαίωμα να τροφοδοτεί τα σιλό με δεδομένα. Επανέρχομαι στο ερώτημα της ποιότητας των δεδομένων που είπατε ότι και, εσεί, και μάλλον ότι είναι ακόμα πιο σημαντική από ό,τι τώρα διότι εάν εισαχθούν εσφαλμένα δεδομένα και ίσως και σε άλλα σιλό από αυτά τα οποία χρησιμοποιούνται τώρα, ίσως να οδηγηθούμε σε πολύ λανθασμένες πληροφορίες. Και πώς θα αντιμετωπίζουμε τότε αυτό το ενδεχόμενο. Το τεχνικό θέμα, εάν δηλαδή οι ειδικέ πληροφορίες θα πρέπει να ε, μπαίνουν σε διαφορετικά σιλό, αυτό θα γίνει σε ένα βήμα ή θα πρέπει να μπαίνουν σε διαφορετικά σύλλογα και τι γίνεται και με την διαγραφή των εσφαλμένων δεδομένων ή δεδομένων που δεν είναι πλέον επίκαιρα. Πρέπει να τα διαγράψω από τα διάφορα σύλλογα ή μπορεί αυτό να γίνει διαμιάς σε ένα βήμα. Και τέλος η ερώτηση που έκανε η κυρία Στίβενς στην προηγούμενη συζήτηση. Εάν βάλουμε όλα αυτά τα δεδομένα μαζί και τα διασυνδέσουμε αυτό αυξάνει τα προβλήματα από κυβερνοεπιθέσεις και χρειάζονται άλλου είδους προετοιμασίες για να αντιμετωπιστεί μια τέτοια ενδεχόμενη πρόκληση στο μέλλον. Ευχαριστώ. Εσείς κύριε εμπειρογνώμων, ευχαριστώ. Όταν μίλησα για μείωση του κόστους, εννοούσα το κόστος της έρευνας, όχι δημιουργίας του συστήματος. Έχετε δίκιο ότι η δημιουργία του συστήματος είναι δαπανηρή αν και δεν θα είναι ένα κεντρικό σύστημα, θα είναι η δυνατότητα διασύνδεσης των υφιστάμενων συστημάτων, αλλά και αυτή κοστίζει χρήματα. Αν υπολογίσουμε τώρα το κόστος όλων των ενεργειών που γίνονται τώρα μέσα στα συστήματα των ΣΥΛΟ, μπορεί ο στόχος επίτευξης, μάλλον η επίτευξη του στόχου μείωσης του κόστους να είναι δυνατή. Αν θα, πρέπει, αν θα μπορεί να γίνει με ένα κλικ ή με μια ενέργεια αυτό δεν είναι ερώτηση που πρέπει να απευθυνθεί στην ε, αρχή προστασία δεδομένων. Όμω, αν δεν είναι ο στόχο αυτό, τότε ποιο είναι. Υποθέτω ότι ο βασικό στόχο είναι όντω να μειωθούν τα βήματα, οι δράσεις που πρέπει να γίνουν για να έχουμε υψηλού επίπεδου προσβάσιμα δεδομένα υπέρ των χρηστών ως ε, ε, ε, αρχή προστασίας των δεδομένων μπορεί να έχουν κάποιες ερωτήσεις σχετικά με το ποιος θα έχει πρόσβαση στα δεδομένα και ασφαλώς και ελπίζω ότι η εισαγωγή των νέων μηχανισμών για την εργασία των ΣΥΛΟ θα σημαίνει ότι οι δράσεις αυτές μπορούν να ληφθούν την ίδια στιγμή. Δημιουργείται πρόβλημα σφάλματος που θα κατασπαρεί μετά σε όλα τα ΣΥΛΟ. Προβλήματα τέτοια πιθανότατα υπάρχουν. Το πρόβλημα που έχουμε για την ώρα είναι ότι τα δεδομένα μπορεί να διαφέρουν από το ένα σιλό στο άλλο. Και αυτό είναι πολύ πιο επικίνδυνο και για την ποιότητα των πληροφοριών και για την προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων των οποίων τα δεδομένα είναι αποδικευμένα εκεί αλλά και για τους χρήστες ε, των αρχών ε, επιβολής του νόμου. Δημιουργούνται προβλήματα ε, για τις κυβερνοεπιθέσεις και ναι και όχι. Δηλαδή το γεγονό και μόνο ότι μιλούμε για μεγάλα συστήματα ή συστήματα τα οποία διαχειρίζεται ένα κεντρικό σημείο δεν ανοίγει αυτό την πόρτα σε πρόσθετους κινδύνους. Μπορεί να μειώνει μάλιστα κινδύνους κυβερνοεπιθέσεων γιατί μειώνει τον αριθμό των σημείων από τα οποία μπορεί να εισέλθει η επίθεση. Αλλά όταν γίνει μια επίθεση και όταν επιτύχει την πρόσβαση, ίσως τότε ο κίνδυνος να είναι πολύ μεγαλύτερος παρά αν είναι το σύστημα χωρισμένο σε σιλό ξεχωριστά. Παρόλο που οι εμπειρίες των υπευθύνων για την ασφάλεια των ε, πληροφορικών συστημάτων λέει ότι όσο λιγότερο χρησιμοποιούνται τα σιλό, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα ότι κανείς δεν δει ότι έχει γίνει η επίθεση. Ευχαριστούμε κύριε Βιμπερόφσκι και για την παρουσίασή σας και για την απάντηση που δώσατε στην ερώτηση της κυρία Ζήπελ. Κάπως έχουμε βέβαια καθυστερήσει. Ας περάσω λοιπόν αμέσως στο επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη, αφού σας ευχαριστήσω και πάλι για την παρουσία σας. Και πρόκειται για δύο σημαντικά έγγραφα τα οποία θα παρουσιαστούν σε εσά σήμερα το απόγευμα και που συνδέονται άμεσα με το έργο της ε, Κοινοβουλευτικής μας Επιτροπής, θα ήθελα να συνεχιστεί η συνεδρίαση. Αν πρόκειται να αποχωρήσετε από την αίθουσα, παρακαλώ να το πράξετε εν σιγή. Λοιπόν, έλεγα ότι έχουν σχέση με την εργασία μας και mass surveillance. Το πρώτο της αρμόδιας αρχής εποπτείας από τις αρχές της Ένωσης και ο κ. Ελτχάιμερ καλώς ήρθατε θα παρουσιάσει την μελέτη και μετά θα, ακούσουμε άλλη μελέτη της ΣΤΟΑ για την δημιουργία βιομηχανίας ICT στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ξεκίνησε το 2016 με πρωτοβουλία των επικεφαλής της τώρα. Θα είναι η δεύτερη μελέτη αυτή λοιπόν. Πρώτος ο κύριος Ολτχάιμερ λοιπόν έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Θα θυμάστε ότι το 2013 έγιναν αποκαλύψεις για τον... Οι αποκαλύψεις του Έντορτ Σνόντιν ε, οδήγησαν ε, σε μεγάλη αγανάκτηση διό, διότι παρακολουθούνταν οι πολίτες κλπ. Οι απαντήσεις, οι κυβερνήσεις απάντησαν ότι η επιτήρηση ήταν αναγκαία για την αντιμετώπιση του κινδύνου τρομοκρατίας και πράγματι η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε είναι η προστασία των δικαιωμάτων μας με ταυτόχρονη προστασία της ασφάλειας και της ζωής των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην FRA αναγνωρίζουμε τον κεντρικό ρόλο των υπηρεσιών πληροφοριών. Το 2014 και 2015 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε δύο ψηφίσματα για την ηλεκτρονική μαζική επιτήρηση Ευρωπαίων πολιτών, ζητώντας από τις χώρες μέλη να εφαρμόσουν αυστηρές ε, αρχές προστασίας και βεβαίως ε, το μήνυμά σας αυτό παραμένει απολύτως επίκαιρο. Ταυτόχρονα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε από την FRA να κάνει σε βάθος έρευνα για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στα πλαίσια της επιτήρησης. Τα πρώτα μας συμπεράσματα τα δημοσιεύσαμε το 2015 και για πρώτη φορά χαρτογραφήσαμε την νομοθεσία συλλογής προφοριών στην Ένωση. Σήμερα, με μεγάλη μου χαρά, σας παρουσιάζω την τελική μας έκθεση μετά από 3,5 χρόνια ε, λεπτομερούς ερεύνης και αναλύσεως. Η έρευνα ήταν εξαιρετικά δύσκολη ορισμένες φορές και όχι μόνο λόγω των, ε, των ποικίλων νομοθεσιών αλλά και λόγω της εμπιστευτικότητας ε, ή του απορρίτου του τομέα. Με την μελέτη μας η... ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων σας ε, προσφέρει μια ανάλυση των ε, σχετικών νομοθεσιών και μετά από συζητήσεις με πολλούς επιρρογνώμονες σε πολλές χώρες μέλη. Η νομοθεσία για τις χώρες μέλη είναι πρόσφατη και βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Όπως θα δείτε από το χάρτη, με το βαθύ χρώμα δείχνουμε τις χώρες που έχουν κάνει μεταρρυθμίσεις από το 2015 και μετά. Ενώ όλες σχεδόν οι χώρες μέλη έχουν νομοθετικό πλαίσιο για την στοχευμένη επιτήρηση, ορισμένες χώρες μέλη, μεταξύ αυτών Γαλλία, Γερμανία, κάτω χώρες, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν εγκρίνει και νομοθεσία για την γενική επιτήρηση, παρακολούθηση αν θέλετε, των τηλεπικοινωνιών. Άλλες που κάνουν γενική παρακολούθηση δεν έχουν ε, νόμους αρκετά λεπτομερείς ώστε να μπορούν να αντέξουν ανάλυση διότι η έρευνά μας βασίστηκε αποκλειστικά ε, στην νομοθεσία που είναι δημόσιο κτήμα. Μόνο αυτά μπορούσαμε να σχολιάσουμε. Σε ό,τι αφορά τώρα την επιτήρηση παρακολούθηση, η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων έχει ανάγκη από νομιμότητα, εποπτεία και μέσα προσφυγής. Αυτά ερεύνησε η μελέτη μας. Για το πρώτο θέμα της νομιμότητας. Πολλοί από τους ανθρώπους με τους οποίους συνομιλήσαμε και θα δείτε ορισμένες παραθέσεις από αυτά που μας είπαν, επέκριναν την ασάφεια των ορισμών που περιλαμβάνονται στη σχετική νομοθεσία. Η έρευνα της FRA κατέδειξε ότι ακόμα και με νομική συμβουλή είναι δύσκολο να κατανοηθούν οι περιπλοκότητες των νόμων αυτών. Γαλλία, ε, Γερμανία, κάτω χώρες και ε, Ηνωμένο Βασίλειο έχουν μεταρρυθμίσει την νομοθεσία τους για να αντιμετωπίσουν και τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και απειλές, αλλά και για να απαντήσουν σε νέες απειλές, αλλά και για να βελτιώσουν την σαφήνεια. Και αυτό είναι κάτι το οποίο οφείλω να τονίσω. Άλλες χώρες μέλη, όπως η Φιλανδία, ακολουθούν. Όμως, οι συνομιλητές μας στις χώρες αυτές εξακολουθούν να περιγράφουν τους κανόνες που διέπουν την παρακολούθηση ως ασαφείς. Η βασική πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι νομοθέτες είναι να ρυθμίσουν τα των ε, αρχών συλλογής πληροφοριών χωρίς να αποκαλύψουν τις ιδιαιτερότητές τους διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ορισμένες χώρες μέλη το καταφέρουν αυτό καλύτερα από άλλες. Για ορισμένες η συμμόρφωση των εθνικών νομοθετικών πλαισίων με την Ευρωπαϊκή Συνθήκη για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα εξακολουθεί να αποτελεί ένα δύσκολο εγχείρημα. Στο δεύτερο θέμα της εποπτείας δηλαδή των υπηρεσιών συλλογής πληροφοριών, η FRA στόχευσε σε δύο τομείς. Έλεγχος της νομιμότητας των μέτρων παρακολούθησης και προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων τα εθνικά πλαίσια για την εποπτεία είναι πάρα πολύ ποικίλα μεταξύ των χωρών μελών. Όμω, συνήθως βλέπουμε τους ίδιου φορεί που βλέπετε στη διαφάνεια. Δηλαδή, Κοινοβουλευτική Επιτροπή, ανεξάρτητο δικαστικό σώμα, Data Protection Authorities και άλλους οργανισμούς που παρακολουθούν την σωστή εκτέλεση εποπτείας. Υπάρχουν βεβαίως ιστορικές και νομικές διαφορές που σημαίνουν ότι δεν υπάρχει ένα ενίο μοντέλο εποπτείας. Η έρευνά μας μας δείχνει ότι 16 χώρες μέλη έχουν δημιουργήσει ένα ή περισσότερους οργανισμούς, ανεξάρτητους οργανισμούς που ασχολούνται αποκλειστικά με την προστασία. Λύση η οποία είναι προτιμητέα σύμφωνα με την γνώμη της FRA. Οι εμπειρογνώμονες συνομιλητές μας θεωρούν ότι η αποτελεσματική υποπτία πρέπει να έχει τρία χαρακτηριστικά. Πρώτον, πλήρη ανεξαρτησία. Δεύτερον, ξεκάθαρες αρμοδιότητες. Τρίτο, διαφάνεια στον δημόσιο έλεγχο. Η νομική ανεξαρτησία των οργανισμών εποπτείας είναι αναγκαία για να μπορεί να λειτουργεί με αντικειμενικότητα και να αποκτήσει την εμπιστοσύνη του κοινού. Η έκθεσή μας τονίζει τα βασικά χαρακτηριστικά της πλήρους ανεξαρτησίας. Παραδείγματα είναι κοινοβουλευτικές επιτροπές, που θα, ο πρόεδρος θα προέρχεται από τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως. Επίσης να είναι εγκατεστημένοι οι οργανισμοί ε, εποπτείας σε άλλα κτίρια μη κυβερνητικά. Για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα χρειάζεται πλήρης πρόσβαση στα, στη συλλογή δεδομένων και ικανότητα πλήρους χρήσης των δεδομένων ανεπαρκής γνώση των μελών των οργανισμών εντοπίστηκε συχνά από τους συνομιλητές μας ως αντικείμενο κριτικής. Ταυτόχρονα οι εκπρόσωποι των οργανισμών εποπτείας εντοπίζουν και έλλειψη εμπιστοσύνης του κοινού στις δραστηριότητες λόγω της μυστικότητας των εργασιών αυτών. Γιατί χωρίς να είναι ανοιχτή στην δημόσια εποπτεία δεν επιτυγχάνουν να αποκτήσουν την εμπιστοσύνη του κοινού το οποίο υποτίθεται ότι προστατεύουν. Σημαντικές προκλήσεις στο εθνικό επίπεδο, ωστόσο ίσως από τα πιο ανησυχητικά συμπεράσματά μας ήταν η πολύ ασθενής εποπτεία της διεθνούς συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών συλλογής πληροφοριών. 17 από τις 28 χώρες μέλη δεν προβλέπουν στην ομοθεσία τους ανεξάρτητη εποπτεία για τα δεδομένα που λαμβάνουν από αλλοδαπές υπηρεσίες. Η ΦΡΑ θεωρεί ότι η ενίσχυση της εποπτείας και στο εθνικό και στο διεθνές επίπεδο είναι κρίσιμη σημασία για τα επόμενα χρόνια. Τέλος, για το τρίτο, δηλαδή για τα μέσα προσφυγής. Η έρευνα της ΕΦΑΡΕΗ βρήκε ότι τα άτομα αντιμετωπίζουν δυσχέρειες στα πλαίσια των εθνικών νομοθεσιών μη έχοντας μέσα προσφυγής, ιδίως για το δικαίωμα ειδοποίησης του προσώπου που παρακολουθείται και την προσβάση σε πληροφορίες. Οι 25 χώρες μέλη δίνουν τη δυνατότητα στο άτομο να προβεί σε καταγγελία σε μη δικαστικό οργανισμό βρήκαμε ότι το σύστημα, τα συστήματα αυτά είναι πολύ ποικίλα και δεν διαθέτουν επαρκή διαφάνεια. Και διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν πολλά παράπονα προσώπων που δεν γνωρίζουν σε ποιον φορέα πρέπει να απευθυνθούν. Και αυτά λόγω της έλλειψης διαφάνειας και λόγω της μυστικότητας σχετικά με τις διαδικασίες. Περιπτώσεις, οι υποθέσεις που έχουν σχέση με τη συλλογή προφοριών έχουν και άλλα ε, δυσχερή χαρακτηριστικά. Μπορεί τα άτομα να μην έχουν, μάλλον οι, οι υπηρεσίε να μην διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία ή να μην έχουν πρόσβαση σε ορισμένα στοιχεία πληροφοριών. Ορισμένε χωρισμένοι έχουν θεσπίσει εναλλακτικού μηχανισμού σε μια προσπάθεια να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια. Όμω, διαπιστώνει η μελέτη μα ότι λόγω του πολυτεχνικού χαρακτήρα των θεμάτων συλλογή πληροφοριών, οι δικαστέ εξακολουθούν να μην διαθέτουν την αναγκαία τεχνογνωσία για την κρίση των υποθέσεων αυτών. Αν και αυτό είναι προφανές ότι δηλαδή οι ανταλλαγές απόψεων μεταξύ των διαφόρων φορέων γίνονται, η έλλειψη τεχνογνωσίας των δικαστικών αρχών εξακολουθεί να εμποδίζει την αποτελεσματικότητα των μέσων πρόσφυγης των ένδικων μέσων. Εν τέλει, η έκθεσή μας εντοπίζει και κάποιες ε, λύσεις που μπορούν να είναι ως εξής. Πρώτο, θέσπιση λεπτομερών και προβλέψιμων κανόνων για ε, την εποπτεία. Δεύτερον, ανεξάρτητη και διαρκής εποπτεία των υπηρεσιών συλλογής πληροφοριών με απο, αποφορείς και πρόσωπα με την απαραίτητη τεχνογνωσία. Τρίτο, διαθεσιμότητα μηχανισμών προσφυγής ενώπιον δικαστικών ή μη δικαστικών αρχών με τις αναγκαίες εξουσίες. Θα βρείτε στη μελέτη μας 16 συστάσεις της FRA προς νομοθέτες και makers, ένα είδος εργαλειοθήκης που θα επιτρέπει την δημιουργία κατάλληλης και θέσπιση, και θέσπιση νομοθεσίας. Τα βασικά μας συμπεράσματα απηχούν την βαθιά πεποίθηση της FRA ότι οι μηχανισμοί αυτοί πρέπει να περιβληθούν τον ομαδία της νομιμότητας αν θέλουμε να εξασφαλίσουμε την ε, εποπτεία. Είμαστε πεπισμένοι ότι οι μηχανισμοί αυτοί μπορούν να θεσπιστούν με τρόπο που δεν θα οδηγήσει σε κίνδυνο τον, την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των θεμελιωδών αξιών μας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ολτχάιμερ για την παρουσίαση. Θα δώσω τον λόγο τώρα τους και στις συναδέλφους μου που επιθυμούν να παρέμβουν για τη μελέτη σας. Έχω τον κύριο Άλμπρεχτ πρώτο Παρακαλώ, έστε σύντομοι για να έχουμε τη δυνατότητα να τηρήσουμε το χρονικό μας πλαίσιο και να παρακολουθήσουμε και την παρουσίαση της επόμενης μελέτης και να διεξαχθεί και κάποια συζήτηση. Α, ο κύριος Αγγιλάρ πρώτος. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και τον κύριο Ότχαϊμερ. Ε, βέβαια, πολύ ενδιαφέρουσα η μελέτη. Εύστοχη και θα αποτελέσει πολύτιμο οδηγό για όλους όσοι προβληματιζόμαστε για αυτό το σκάνδαλο, γιατί παίζει σκανδάλο επρόκειτο τότε που μάθαμε για την μαζική παρακολούθηση από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών τον είπα που παρεδίασε το, το απόρριτο των δεδομένων, το ιδιωτικό βίο ε, και πολιτών απλών αλλά και φυσικά ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να σας μιλήσω ή να σας ρωτήσω τέλος πάντων για αυτό που είπατε για αυτά τα παραθυράκια, τα κενά στην νομοθετική ρύθμιση και στην έλλειψη ε, σαφήνειας. Γιατί αυτά τα παραθυράκια στην νομοθεσία όταν μιλούμε για το απόρριτο των επικοινωνιών αποτελεί έγκλημα. Έτσι το θεωρούν τα ποινικά δικαστήρια των κρατών μελών όταν κανένα παρεμβαίνει, επεμβαίνει σε επικοινωνία με οποιοδήποτε ε, τρόπο ταχυδρομείο, mail, ξέρω εγώ, στα κινητά, επαρέμβαση. Ε, οπότε, οπότε γίνει κάτι τέτοιο, όπου εις βάρος οποιοδήποτε πολίτη, και στην Ισπανία και παντού. Αλλά, άρα για πέστε μας. Έχετε υπόψη σας κάποιο είδους νομολογία. Μπορεί να μας βοηθήσει να εξαγάγουμε κάποια συμπεράσματα. αποφάσεις, νομολογία από δικαστήρια. Κάτι που θα μπορούσε να έχει κάποια σημασία. Θα μπορούσε αυτό να βοηθήσει το Ευρωπαϊκό τόσο ώστε να νομοθετήσει στο μέλλον, να νομοθετήσει από πλευράς ποινική. Οπότε αυτό θα αποτελεί προτέρα πολύτιμη εμπειρία. Ευχαριστούμε κύριε Κόλλιο. Σας ευχαριστούμε κύριε, ευχαριστούμε για την εισήγησή σας. Πρόκειται για δουλειά πολύ σημαντική και από ό,τι έχω καταλάβει είναι σημαντικό να ξέρουμε ξεκάθαρα το τι έχει γίνει και τι γίνεται με τις υπηρεσίες πληροφοριών να μην επανεθούν τα λάθη του παρελθόντος και τα κρατημέλη να έχουν επιλογές στη χάραξη πολιτικής. Όπως γνωρίζετε, έχει περιορισμένες αρμοδιότητες η Ένωση. Αλλά οι υπηρεσίες πληροφοριών ασχολούνται όλο και περισσότερο με την τρομοκρατία. Επομένω, είναι πολύ σημαντικέ οι αρμοδιότητέ μα σχετικά με αυτό. Έχω σα ρωτήσω τα, τα εξή ε, τρία. Πρώτα απ' όλα, εξηγήστε μου περισσότερο όσον αφορά το πώ αντιλαμβάνεστε την εθνική ασφάλεια και τη σχετική εξαίρεση που μπορεί να συντρέχει ε, για να παρακαμφθεί ή τέλο πάντων μπορεί να την επικαλεστεί όσον αφορά την εφαρμογή του κοινωνικού δικαίου. Μα υπάρχει τέτοια νομοθεσία. Τι γίνεται ας πούμε με το SIS. Θα, πρέπει, θα μπορεί κάποιος να επικαλεστεί αυτή την, ε, την, την ασφάλεια ούτω ώστε να παρακάμψει το σύστημα. Υπάρχει νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Επίσης ε, μας ε, είπατε ότι το δίκαιο προστασία δεδομένων το κοινοτικό αφορά και την συλλογή δεδομένων αλλά και η συλλογή δεδομένων από μόνη της είναι παρέμβαση, παράβαση. Άρα ισχύουν αυτά για τις σχετικές υπηρεσίες. Επίσης, γιατί πέντε κράτη-μέλη έχουν νομοθεσία όσον αφορά την παρακολούθηση των επικοινωνιών ή τηλεπικοινωνιών. Άρα τι γίνεται με την μαζική παρακολούθηση. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μπούχνερ έχει το λόγο. Πρώτα σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Έχω τρεις ερωτήσεις. Πρώτη, παλαιότερα στην Γερμανία υπήρχε μια σχετική νομοθεσία που προέβλεπε περιορισμό του αριθμού των δεδομένων που μπορούσαν να αποθηκευτούν ε, σχετικά με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, τουλάχιστον από κρατική πλευρά. Φαίνεται όμως τώρα η τάση να είναι ακριβώς η αντίθετη, δηλαδή οι κρατικές αρχές προσπαθούν να συλλέγουν όσο δυνατόν περισσότερα δεδομένα. Σκέπτομαι για παράδειγμα το κινέζικο social call system ή το ευρωπαϊκό που προσπαθεί να αξιολογήσει για παράδειγμα στην Κίνα την κοινωνική συμπεριφορά και να την επιβραβεύσει, να την τιμωρήσει. Και στην Ευρώπη γίνεται προσπάθεια με συλλογή τέτοιων δεδομένων να προβλέψουν την εγκληματική συμπεριφορά. Εγώ θεωρώ ότι αυτά ε, τραυματίζουν βαριά τι ε, βασικέ αρχέ για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Και το ερώτημα είναι τι μπορεί να γίνει. Δεύτερον, Google, Microsoft, WhatsApp και όλοι αυτοί οι μηχανισμοί. Ε, αυτοί συλλέγουν πλήθος μέγα δεδομένων η Microsoft έχει πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα ε, των ε, ηλεκτρονικών υπολογιστών σας. Το ίδιο Android. Πρόκειται για μια θεαζόνη, διότι ποιος σας λέει ότι δεν θα έχουν πρόσβαση κάποια στιγμή οι κρατικές αρχές σε, αυτά τα δεδομένα. Μπορεί να γίνει κάτι νομοθετικά. Και τρίτο, όπου σίγουρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, είναι βεβαίως αυτά που κάνουν οι αλλοδαπές μυστικές υπηρεσίες στην ε, Γερμανία και θυμίζω ότι έγινε με την Αμερικανική ε, υπηρεσία που παρακολουθούσε ε, κινητά τηλέφωνα και Γερμανών ηγετών. Ο κύριος Αλμπρέχτ. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κάτι σε σχέση με το πώς μπορούμε να νομοθετήσουμε, πώς μπορούμε να έχουμε ρυθμίσεις για τις επιβλήσεις πληροφοριών. Γιατί γνωρίζω ότι έχουμε το άρθρο 4 παράγραφος 2 ή 3 ε, της ε, ε, ε συνθήκης εκεί η εθνική ασφάλεια αποτελεί εξαίρεση. Δεν ρυθμίζεται, δεν υπόκειται στις ρυθμίσεις της ε, συνθήκης. Εσείς είπατε ότι αξιολογείτε το τι ισχύει όσον αφορά τον έλεγχο, όσον αφορά την νομοθεσία για τις περισσίες πληροφοριών Κοιτάξτε, ότι τα μελετήσατε και είπατε ότι υπάρχουν ε, διαφορετικέ ρυθμίσει, διαφορετικά συστήματα ελέγχου και ανεπάρκεια αυτού του ελέγχου. Οπότε, αν θέλετε να μεταβληθεί αυτή η κατάσταση, ε, τότε θα πρέπει να δούμε, ε, να έχουμε ευρωπαϊκά πρότυπα, ευρωπαϊκέ δίκτυες ασφαλεία. Οπότε, και εγώ αυτό θα ήθελα. Ε, αν υπάρχει κάποια πιθανότητα, δυνατότητα να πετύχουμε κάτι τέτοιο και ακριβώς επί τη βάση ότι οι αρχές συνεργάζονται ε, και στενά. Αξιολογήσατε και το ζήτημα της ε, έννοιας εθνική ασφάλεια. Έχουμε εκεί σύγκληση, έχουμε απόκληση διαφορές, τα σύνορα. Τι μπορούμε να κάνουμε για αυτήν την έννοια την ειδική ασφάλεια, τις ασφαλείας, την αστυνομία. Ο εισηγητής, ευχαριστώ πρόεδρε και ευχαριστώ και για τις ερωτήσεις. Να αρχίσω από την τελευταία ερώτηση. Αλλά ταυτόχρονα απαντήσω και στον κύριο Κόλλιο. Το Κοινοβούλιο ζήτησε να εξετάσουμε τις εθνικές νομοθεσίες. Εξού και η μελέτη μας. Παρακολουθήσαμε το τι ισχύει, πώς εξελίχθηκε η κατάσταση από το 2015 μέχρι σήμερα, τι προβλέπεται σε επίπεδο ένωσης. Δεν αναλύει η μελέτη, ε, τα, τα, τα, δεν υπησέρχεται ε, τις λεπτομέρειες των ορίων της κοινωτικής αρμοδιότητας και ακριβώς αυτό μας είπαν οι συνομιλητές μας ε, στα κρατημέλη. Το θέμα δηλαδή του ορισμού της έννοιας εθνική ασφάλεια. Πήγαμε σε πολλά κρατημέλη και σε πολλές περιπτώσεις το θέμα αυτού του ορισμού ανεδίθη. Ίσως όχι σε δικονομικά πλαίσια το κριτήριο δηλαδή του δικαστή που κρίνει αυτό. Ίσως ο δικαστής δεν έχει πρόβλημα με την έννοια. Το πρόβλημα είναι όταν δεν υπάρχει ορισμό στο δίκαιο. Οπότε, κοιτώντα το από πλευρά κοινωνικού δικαίου, υπάρχει το θέμα. Αυτό και ε, πρόκυψε. Δυστυχώ. Έχουν πολύ περιορισμένη νομολογία σε σχέση με αυτά τα όρια. Πάντως, Οργανισμός των Δικαιωμάτων αυτό προσπάθησε να κάνει. Να περιχαρακωθεί αυτό το, αυτό το, αυτή η έννοια και να βρεθεί ένας ορισμός της έννοιας εθνική ασφάλεια. Επαναρχόμαστε τώρα στο θέμα της ε, έλλειψης αφήνειας που έχει να κάνει και με την εθνική ασφάλεια. Να είναι παράδειγμα δηλαδή μια ενία η οποία χρειάζεται να διέπεται από περισσότερη σαφήνεια και έναν ορισμό. Οπότε η πραγματική πρόκληση είναι ότι χρειάζεται περισσότερη σαφήνεια στην νομοθεσία. Όπω σα είπαμε, πολλά μέλη πρόσφατα τροποποίησαν νομοθεσία τους για αυτό το πρόβλημα. Καταβάλλονται προσπάθειες προς τη σωστή κατεύθυνση. Και με αυτή την νομοθεσία για τις υπηρεσίες ασφαλείας έχουμε κάποιες τεχνικές που περιγράφονται και που εξηγούν τι γίνεται με τις αρμοδίτες των υπηρεσιών πληροφοριών και έτσι κανείς φέρνει ε, αποσαφήνιση, σαφήνεια στην ε, νομοθεσία και έτσι φροντίζει κανείς και την τήρηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Δεν βρήκα αρκετή νομολογία. Κύριε Λόπες Αγγιλιάρ, όπως είπατε κι εσείς. Και στην Ευρώπη και στα κράτη-μέλη λίγη νομολογία. Νομίζω το είπα και στην αρχή της ομιλίας μου. Το πρόβλημα είναι ότι πάρα πολύ λίγες είναι οι υποθέσεις που έχουν περάσει από τα δικαστήρια. Επίσης για τον κύριο Κοέλιο όσον αφορά την ε, παρέμβαση, επέμβαση και την εφαρμογή της κοινωτικής νομοθεσίας θέλουμε να φανεί διαφορά μεταξύ της έννοιας της ε, παρέμβασης και το κοινωτικό δίκαιο σε σχέση με τις σημείες ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πέραν δηλαδή των κανόνων προστασίας δεδομένων που προβλέπει το κοινωτικό δίκαιο. Ξέρετε, σήμερα το πρωί κιόλας κάπου αλλού το συζητήσαμε. Τι γίνεται όσον αφορά την εφαρμογή της ε, προστασίας των δεδομένων και όσον αφορά Τώρα τα ζητήματα προστασίας του ιδιωτικού βίου αυτά είναι πάρα πολύ αλληλοσχετιζόμενα. Είναι και θέμα συλλογή δεδομένων και επόμενος αναδύεται το θέμα της παρέμβασης. Βέβαια, δεν ισχύει η οδηγία για την προστασία δεδομένων, γιατί εδώ υπάρχει εξαίρεση εθνικής ασφάλειας. Τώρα επίση ε, είπατε για τα πέντε κρατημέλη που έχουν νομοθεσία όσον αφορά την παρακολούθηση των ε, επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών. Όχι, δεν έχουμε. Αλλά και στην έκθεση του 15 και στην ε, έκθεση που έχετε σήμερα αναχείρα, αυτό θέλουμε να δείξουμε. Ότι από πλευράς σύγκρισης και συγκρισιμότητας ο όρος μας για παρακολούθηση είναι χρήσιμος. Δεν είναι όμως νομικός όρος. Όσο μας βοηθάει να καταλάβουμε περισσότερο. Το τι κάνουν οι υπηρεσίες παρακολούθησης όταν συλλέγουν ε, πάρα πολλά δεδομένα. Α, ας πούμε, έχουμε ένα από τα λίγα γραφήματα που λέει που αναφέρεται σε αυτή τη μαζική παρακολούθηση. Έχουμε την νέα Ολλανδική νομοθεσία τα, τα έχετε αυτά στην εισήγησή μας, στην έκθεσή μας. Ε, εκεί βλέπετε τη διαδικασία στους εξεδομένων. Και για να σας απαντήσω, όχι, τα πέντε κρατημέλη που έχουν νομοθετήσει για τις παρακολουθήσεις των τηλεπικοινωνιών και επικοινωνιών δεν έχουν πει κάτι, δεν έχουν νομοθετήσει και για την μαζική παρακολούθηση. Τώρα όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα και τη συλλογή των δεδομένων Γι' αυτό μας ερώτησε κάτι ο κύριος Μπίχνερ. Ε, αυτό είναι θέμα το οποίο δεν εφήγει στην έκθεσή μας. Αυτό θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο άλλης μελέτης. Τα είπαμε το 2015 όμως. Συλλογή πληροφοριών από διάφορες συσκευές. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Και είναι και κάτι που γίνεται από τις δημόσιες αρχές. Τώρα, πώς κανείς πρέπει να νομοθετήσει σε νοσιακό επίπεδο. Α, όχι, συγγνώμη, γιατί μας είπατε κάτι για την παγίδευση του τηλεφώνου της κυρίας Μέρκελ. Όχι, όχι, δεν το εξετάσαμε αυτό ιδιαίτερα. Βέβαια υπάρχει η ανάλυση που την ξέρετε για την ανταλλαγή δεδομένων, για την παρακολούθηση επικοινωνιών, αλλοδαπών. σε σχέση με την εθνική νομοθεσία, σε σχέση με τον έλεγχο των ανεξαρτήτων αργών και να καταλήξουμε, να ολοκληρώσουμε με αυτά που είπε για την ανάγκη νομοθεσία σε κοινωτικό επίπεδο ο κύριος Άλμπριχτ. Κατελήγω στο συμπέρασμα, λαμβάνοντα υπόψη όλα αυτά και λαμβάνοντα και υπόψη την εξέλιξη της Ένωσης Ασφάλειας όπως είπε και για την τρομοκρατία του ο κ η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να εξασφαλίσει ότι κάθε νέα πολιτική λαμβάνει υπόψη αναβαθμίση της συνεργασίας των αρμοδίων υπηρεσιών το σύστημα εποπτείας, παρακολούθησης και δεδομένων. Αυτό θα μπορούσε να το προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση και για τις απαντήσεις. Ας περάσουμε τώρα στη δεύτερη μελέτη της ΣΤΟΑ σε ό,τι αφορά την επίτευξη ενό ε, κυρίαρχου και αξιόπιστου τομέα τεχνολογιών πληροφόρηση και επικοινωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα δώσουμε το λόγο στον ομιλητή, τον κύριο Ριβέρα Πάστο, να έρθει εδώ στο βήμα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 Thank you, Chair, and thank you to all of you for joining us. Ευχαριστώ. Είναι ένα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα που εξετάζουμε σήμερα για την Ευρώπη. Yeah, it's working. It's crucial because I think that... Πολύ σημαντικό λοιπόν γιατί θέλουμε να διασφαλίσουμε την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών ε, για την ολοκλήρωση μιας ε, υγιούς ε, ψηφιακής ενίας αγοράς. Και αυτό βασίζεται σε δύο στοιχεία. Πρώτον, θέλουμε να έχουμε τα εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε τον αυξανόμενο αριθμό κινδύνων στην κυβερνοασφάλεια και δεύτερον να διασφαλίσουμε τα θεμελιώδη δικαίωμα στην ιδιωτική σφαίρα ζωής και την προστασία δεδομένων. Εμείς κάναμε αυτή τη ε, μελέτη με τους εξής στόχους. Πρώτον, να περιγράψουμε το περιβάλλον σε ό,τι αφορά την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την προστασία δεδομένων στην Ευρώπη. Δεύτερον, να κατανοήσουμε τις βασικές προκλήσεις σε ό,τι αφορά την ε, βιομηχανία της ε, κυβερνοασφάλειας. Είναι σημαντικό για μας να ε, εξετάσουμε τις ε, υφιστάμενες πολιτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτούς τους τομείς, να μάθουμε, να αντλήσουμε δηλαδή διδάγματα και απόψεις και από τον κλάδο και από επιτυχείς πολιτικές σε άλλες ε, χώρες με τελικό σκοπό να βοηθήσουμε και να επιβάλλουμε προτάσει ε, στου υπεύθυνου χάραξης πολιτική. Ε, πρώτον, ε, έχουμε αναλύσει λοιπόν τι βασικέ απειλές για την ασφάλεια στην Ευρώπη. Δεύτερον, έχουμε αναλύσει το ευρωπαϊκό περιβάλλον τη ασφάλεια στην κυβερνοχώρα και από πλευρά προσφορά και ζήτηση σε τον κλάδο, την αγορά και του δημόσιου φορεί που εμπλέκονται. Τρίτον, έχουμε εξετάσει το σύστημα προστασία δεδομένων στην Ευρώπη και τέλος αναλύσαμε τις ε, πολιτικές για να εξετάσουμε επιμέρους ε, επιλογές πολιτικής. Έχουμε τέσσερις βασικές ε, κατηγορίες απειλών. Τρομοκρατία, κατασκοπία, έγκλημα και το λεγόμενο hacktivism, δηλαδή hacker ακτιβιστές. Υπάρχουν υποψίες ότι ακόμα και ξένες κυβερνήσεις μπορεί να υποκινούν κάποιες από αυτές τις ενέργειες και μάλιστα και οι πιο γνωστές και εδρεωμένες επιχειρήσεις απειλούνται κάποια στιγμή από τις κυβερνοεπιθέσεις. Ε, τα πιο βασικά οι βασικότεροι κλάδοι που πλήττονται είναι ε, ο κλάδος ε, των χρηματοοικονομικών, ε, τηλεπικοινωνίες, ενέργεια και ε, δημοσιοδιοίκηση. Για παράδειγμα, τον Δεκέμβριο του 2015 υπήρξε ε, επίθεση στο ηλεκτρικό δίκτυο της Ουκρανίας η πρώτη γνωστή λοιπόν κυβερνοεπίθεση σε δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και περίπου 230.000 άνθρωποι έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα για μια περίοδο έως 6 ώρες. Ενδιαφέρον είναι να δούμε ποιο ε, κυνηγάει ποιον λοιπόν, σε ποιου ε, απευθύνονται αυτές ε, οι επιθέσεις. Βάσει των στοιχείων του δεύτερου εξαμήνου του 2016 βλέπουμε ότι σημαντική επίθεση είδαμε από ρωσικές διευθύνσεις IP προς το Ηνωμένο Βασίλειο και τις κάτω χώρε, μάλλον τις ΗΠΑ και τις κάτω χώρες, συγγνώμη. Βλέπετε όμως πως αυτό μπορεί να γίνει σημαντικό και για τις ευρωπαϊκές χώρες. Υπάρχουν ορισμένες ε, σημαντικές ε, τεχνολογίες. Πρώτον έχουμε το διαδίκτυο των αντικειμένων και δεύτερον κυβερνοφυσικά συστήματα. Ο πρώτος κλάδος συμπεριλαμβάνει και συσκευές, κινητά τηλέφωνα, οχήματα, συσκευές, ε, οικιακές συσκευές και ο αριθμό των συσκευών αυτών αναμένεται να αυξηθεί από τα 2,9 δις το 2014 σε 21 δις το 2020. Και έτσι εδώ η ασφάλεια είναι σημαντικό ζήτημα. Ο σχεδιασμός τους ε, δεν ελάμβανε υπόψη τον τομέα της ασφάλειας. Αυτό λοιπόν θα αποτελέσει πρόβλημα τα επόμενα χρόνια. Για παράδειγμα, οι εφαρμογές των γεννών τηλεφώνων που περιλαμβάνουν ε, επικίνδυνο λογισμικό. Το 2016 ήταν 8,5 φορές μεγαλύτερος ε, από τον αντίστοιχο αριθμό το 2015. Μετά θα έχουμε και τεχνολογίες που θα δημιουργήσουν προβλήματα στο ψηφιακό περιβάλλον γιατί είναι σημαντικό ποσοστό των ευαίσθητων υποδομών, ε, δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεπικοινωνιών και πυρηνικών και όλα αυτά εξαρτώνται από τέτοιου είδου συστήματα. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυξάνονται οι επιθέσεις σε τέτοια συστήματα και φτάνουν το 50% σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο. Το εκτιμόμενο κόστος για την κοινωνία εν γέννη αναμένεται να αυξηθεί στα 6 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2021 σε σχέση με τα 400 δις σήμερα. Είναι, βλέπετε, τεράστια αυτή η αύξηση. Μετά πρέπει, θέλουμε να αναλύσουμε το σύστημα, ε, το περιβάλλον μάλλον ε, για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο στην Ευρώπη. Αφενός θέλουμε να δούμε την πλευρά της ε, ζήτησης από πολίτες και επιχειρήσεις. Βλέπουμε λοιπόν ότι η αντίληψη του κινδύνου είναι χαμηλή στην Ευρώπη πάνω από το 50% των Ευρωπαίων πολιτών θεωρούν ότι ε, δεν έχουν ενημερωθεί επαρκώς για αυτό το πρόβλημα. Βλέπουμε ότι οι άνθρωποι με χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο, οι γυναίκες και οι πολίτες της Νότιας Ευρώπης ε, δείχνουν ε, να προβληματίζονται λιγότερο από αυτά τα ζητήματα. Το 1 τρίτο των επιχειρήσεων στην Ευρώπη ε, έχουν ορίσει μία επίσημη ε, πολιτική ασφάλειας πληροφορική. Είναι χαμηλό αυτός ο συντελεστή, Εξαρτάται βέβαια από τη χώρα, από το μέγεθο και τον κλάδο της επιχείρηση. Οι περισσότερε μικρέ επιχειρήσει όμω δεν έχουν κάποια ε, πολιτική ασφαλείας για τα πληροφορικά του συστήματα. Βλέπουμε ότι είναι μια τεράστια αγορά. Το 2020 η αγορά αυτή θα ξεπεράσει τα 100 δις ε, δολάρια παγκοσμίω και στην Ευρώπη το 2018 θα κυμανθεί γύρω στα 25 δις δολάρια. Η αγορά αναπτύσσεται με ένα, σε ένα βαθμό 8% κάθε χρόνο. Όμως υπάρχει μεγάλος κατακαιρματισμός στην Ευρώπη. Περίπου το 1 τρίτο της αγοράς καλύπτεται από τους, ε, το top 15 των ε, παρόχων. Και υπάρχει μεγάλος αριθμός μικρών παρόχων που καλύπτουν την υπόλοιπη αγορά. Μεγάλος κατακαιρματισμός λοιπόν, με πολλές μικρές επιχειρήσεις. Παρουσιάζει λοιπόν ενδιαφέρον η εικόνα της ε, κυβερνοασφάλειας στην Ευρώπη. Αρχικά πρέπει να πούμε ότι η παρουσία της Ευρώπης στην αγορά είναι χαμηλή. Έχουμε δει ότι μόνο 10% των πιο σημαντικών επιχειρήσεων στον κλάδο αυτό είναι ευρωπαϊκές σε σχέση με το 35% που είναι από τις ΗΠΑ. Ο ρόλος λοιπόν της, ε, ε, του ευρωπαϊκού κλάδου σε αυτό το τομέα είναι πολύ χαμηλός έχουμε λιγότερες επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις μας είναι μικρότερες. 40% ε, των επιχειρήσεων στην Ευρώπη έχει κάτω, κάτω από 10 εργαζόμενους, ενώ στις ΗΠΑ που έχει μεγαλύτερες επιχειρήσεις, περίπου 10% είναι με πάνω από 500 υπαλλήλους. Όμω υπάρχει και ζήτημα χρηματοδότηση ε, στην Ευρώπη. Βλέπετε εδώ λοιπόν με το κόκκινο τι ΗΠΑ. Εκεί λοιπόν εδώ έχουμε μηχανισμούς ε, χρηματοδότησης ε, και μεγέθυνσης των επιχειρήσεων. Ενώ στην Ευρώπη, που βλέπετε με το μπλε, υπάρχουν οι προσέλκυση επενδυτών αφορά τα αρχικά στάδια της επιχείρησης και όχι μετά. Γι' αυτό και τα δεδομένα που ε, συγκεντρώνονται από την Ευρωπαϊκή Επιχειρήση και τα χρήματα μάλλον, οι πόροι, ε, είναι πολύ χαμηλότεροι από τους αντίστοιχους στις ΗΠΑ ή σε άλλες χώρες όπως το Ισραήλ. Ο μέσο όρο είναι το 50% των επιχειρήσεων κάτω από αυτή την τιμή, 1 εκατομμύριο στην Ευρώπη, το σημαίνει ότι 50% των επιχειρήσεων λαμβάνουν κάτω από 1 εκατομμύριο ευρώ για τη χρηματοδότηση τη εταιρεία σε σχέση με 8 εκατομμύρια, α πούμε, στι ΗΠΑ. Γι' αυτό εκεί οι επιχειρήσει είναι τόσο μεγάλε και έχουν τόσο μεγάλο μερίδιο τη αγορά. Ω εκ τούτου έχουμε ένα κενό ε, του, σε ό,τι φορά τον όγκο ρευστού που έχουν στη διάθεσή του επιχειρήσει στην Ευρώπη και στι ΗΠΑ για την περίοδο των τελευταίων 30 ετών είδαμε έχουμε μια τεράστια διαφορά. Στο Ισραήλ, για παράδειγμα. Το Ισραήλ είναι μια χώρα ε, για την οποία η κυβερνασφάλεια είναι πολύ σημαντική και έτσι επενδύουν πολύ σε αυτόν τον τομέα. Την ίδια περίοδο ε, έχουν επενδύσει 350 εκατομμύρια δολάρια. Το 60% των όσων έχουμε επενδύσει εμείς στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, σημαντικός ε, τομέας είναι το περιβάλλον της έρευνας στην Ευρώπη, γιατί πολλά από αυτά τα χρήματα, μάλλον από αυτά τα προγράμματα χρηματοδοτούνται από τέτοιους μηχανισμούς. Έχετε εδώ για παράδειγμα χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, ορίζον 2020. Βλέπουμε λοιπόν ότι κάθε χρόνο έχουμε περίπου 55 εκατομμύρια έως 110 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδότηση στην Ευρώπη. Αυτό μπορούμε να το συγκρίνουμε με τα όσα καταβάλει η Βρετανική κυβέρνηση που επενδύει τεράστια ποσά στην ασφάλεια, Εκείνοι λοιπόν δίνουν το τριπλάσιο, τους τριπλάσιους πόρους ε, από το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πρόγραμμα Horizon 2020 υπάρχει ένας νέος μηχανισμός εταιρική σχέση δημόσιο-δυτικού φορέα με σκοπό να προσελκύσει πολύ ψηλότερους πόρους. Οπότε ο δημόσιο τομέα δίνει για παράδειγμα 100 εκατομμύρια το χρόνο και ο ιδιωτικό τομέα αναμένεται να χρηματοδοτήσει με άλλα 300 εκατομμύρια το πρόγραμμα. Αυτό όμω δεν φαίνεται ρεαλιστικό γιατί στην πράξη βλέπουμε ότι η, η συνεισφορά του ιδιώτη, ιδίω ε, στην κυβερνοασφάλιση στην Ευρώπη, ήταν ιδιαίτερα χαμηλή τα τελευταία χρόνια. Οπότε δεν αναμένεται κάποια τεράστια αλλαγή με στα επόμενα χρόνια. Δεν θα αλλάξει λοιπόν τόσο δραματικά εικόνα σε ό,τι αφορά τις ε, εταιρικέ σχέσεις δημοσιοδητικού τομέα. Ε, κάτι άλλο το οποίο είναι σημαντικό για την έρευνα είναι ότι τα έργα είναι πολύ μικρά. Τα περισσότερα, το 75% είναι κάτω από το όριο των 4 εκατομμύριων ευρώ. Έχουμε μιλήσει και με πυρογνώμονε που μα είπαν ότι η καλύτερη επιλογή θα ήταν να χρηματοδοτηθούν μεγαλύτερα προγράμματα. Δεν ξέρω να ισχύει αυτό. Γιατί είναι η μοναδική πρόσβαση στη χρηματοδότηση και δυνατότητα επιτυχία αυτών των μικρών προγραμμάτων. Μετά, σημαντικό είναι ο ρόλος ε, των ε, ε, φορέων των δημοσίων φορέων. Έχει θεσπιστεί ένα πλαίσιο για τη βελτίωση της συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών φορέων και των κρατών μελών. Έχει συσταθεί και μια ομάδα συντονισμού και ένα δίκτυο. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο, ο ΕΝΙΖΑ, ε, υποτίθεται ότι ηγείται της όλας προσπάθειας, όμως ακόμα δεν έχει ε, γίνει πλήρως ανεξάρτητος ε, και μόνιμος φορέας και όχι μόνο γνωμοδοτικός. Είναι κάτι που προτείνεται και στην νέα πρόταση κανονισμού για τον οργανισμό που υπέβαλε η Επιτροπή πριν από μερικού μήνε και θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να έχουμε τέτοιο οργανισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μετά έχουμε την προστασία δεδομένων στην Ευρώπη. Εξετάζοντα τι κανονιστικέ ρυθμίσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία 20 χρόνια, η προστασία δεδομένων ε, βρίσκεται σε αυτό το έγγραφο από την αρχή. Είναι κάτι το οποίο έχει προβληματίσει ιδιαίτερα του υπεύθυνου χαράξη πολιτική στην Ευρώπη. Από την πρώτη οδηγία για την προστασία δεδομένων που υιοθετήθηκε το 1995. Ε, πριν από μερικούς μήνες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μία ε, ολική αναθεώρηση των κανόνων προστασίας δεδομένων και καταλήξαμε στον κανονισμό προστασίας δεδομένων που δημοσιεύθηκε πριν από μερικούς μήνες και νομίζω το Μάρτιο του 2018 θα περάσει από το Συμβούλιο. Και πάλι όμως ε, το πλαίσιο EDPR είναι ένα πολύ καλό πλαίσιο προστασίας δεδομένων των πολιτών, όμως υπάρχουν και προβλήματα. Πρώτον έχουμε την ισορροπία μεταξύ της προστασίας δεδομένων και της δημιουργίας καινοτόμων υπηρεσιών βάσει αυτών των δεδομένων. Πρέπει λοιπόν να βρούμε την κατάλληλη ισορροπία για να έχουμε ε, καλές υπηρεσίες στην Ευρώπη, η η Αμερική και η Κίνα θα καλύψουν αυτό το κενό που δεν ακολουθούν τόσο αυστηρούς κανόνες ως εμείς. Και το δεύτερο είναι η προκλήση που έχουμε για τι ε, ροέ προσωπικών δεδομένων. Γιατί τα προσωπικά δεδομένα από την Ευρώπη πάνε σε τρίτε χώρε. Εμεί έχουμε προσδιορίσει στρατηγικέ για την αντιμετώπιση του ζητήματο, όμω η αλήθεια είναι ότι μόνο το 1% των ε, σημαντικών παρόχων όπως η Google και η Amazon είναι από χώρες όπως οι Ηνωμένε Πολιτείε, Κίνα, Ιαπωνία που δεν έχουν τόσο αυστηρούς κανόνες προστασίας δεδομένων όσο η Ευρώπη. Είναι λοιπόν δύσκολο να επιβάλλουμε τους δικούς μας κανόνες σε αυτές τις χώρες. Οπότε υπάρχει σημαντικό κενό εδώ. Και θα είναι δύσκολο για εμάς να εφαρμόσουμε στην πράξη αυτόν τον κανονισμό όταν τα προσωπικά δεδομένα φεύγουν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, προσδιορισμός ε, κάποιων επιλογών πολιτικής στην Ευρώπη βάσει των πιο σημαντικών προκλήσεων που έχουμε εντοπίσει. Υπάρχουν κανονιστικές, ε, ερευνητικές και άλλες προκλήσεις στη μελέτη μας έχουμε καταλήξει ορισμένε προτάσει. αρχικά στις ε, θεσμικές πολιτικές για την ενίσχυση του ρόλου τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των εθνικών αρχών σε αυτά τα ζητήματα, για την εναρμόνιση της νομοθεσία. Μετά έχουμε τον ε, κλάδο της αγοράς. Ε, να έχουμε αρμόνιση των προϊόντων, ναι, των προτύπων και έχουμε και ορισμένες ε, βιομηχανικές πολιτικές γιατί ο κλάδος υπολείπεται του αντίστοιχου κλάδου άλλων χωρών και έχουμε ένα σύνολο πέντε πολιτικών για να αλλάξουμε αυτή την ε, τάση. Να ενισχύσουμε τα προϊόντα κυβερνοασφάλειας ανοιχτού λογισμικού να ενισχύσουμε ε, τη δημιουργία μηχανισμών, ε, επενδυτικών μηχανισμών, να ε, στηρίξουμε την ερευνητική δραστηριότητα και να τη φέρουμε πιο κοντά στην αγορά και να αυξήσουμε τη διαθεσιμότητα εργαζομένων στον τομέα της ασφάλειας. Γιατί υπάρχει σημαντική έλλειψη προσόντων και δεξιοτήτων σε αυτόν τον τομέα στην Ευρώπη. Και τέλος να ενημερώσουμε τους τελικούς χρήστες, τις μικρές επιχειρήσεις ε, που κατά πιθανότητα δεν θα είναι τόσο προστατευμένες. Έχουμε αξιολογήσει όλες ε, τις επιλογές πολιτικής βάσει μια σταθμισμένη μήτρας και ε, μπορεί αυτό να αποτελέσει ένα χρήσιμο και ωφέλιμο εργαλείο για τους υπεύθυνους χαρακτήρες πολιτικής. Αυτά είναι τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης μας. Πρέπει ε, να διασφαλίσουμε την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών και επιχειρήσεων, όμως έχουμε διαφορετικούς παράγοντες, όπως είναι ο κατακριματισμός της αγοράς, ανεπαρκείς στρατηγικές, έλλειψη χρηματοδότησης, που ε, ε, ενισχύουν την εξάρτηση από μη ευρωπαϊκούς παρόχους και έτσι δεν επιτρέπουν στην αγορά να αποκτήσει αντοχή και ανθεκτικότητα έναντι των κυβερνοεπιθέσεων. επιθέσεων. Ε, το πρόβλημα επίσης είναι ότι ε, μπορούν ε, να αξιοποιηθούν διάφοροι μηχανισμοί από ξένες κυβερνήσεις σε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο για τους δικούς τους σκοπούς. Έχει αναθεωρηθεί η νομοθεσία και για την κυβερνοασφάλεια με την οδηγία ΕΝΙΖΑ και με τον νέο κανονισμό προστασίας δεδομένων, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα αν θα καταφέρουμε να καλύψουμε την προστασία δεδομένων των πολιτών, γιατί ε, οι περισσότερε υπηρεσίε παρέχονται από μη ευρωπαϊκέ ε, χώρε. Έχουμε προτείνει διάφορε επιλογέ για να βελτιώσουμε αυτή την κατάσταση. Ε, Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ριβέρα Πάστορ. Ε, κυρία έχεις έχει ζητήσει το λόγο. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Ξυπνάμε σιγά σιγά και βλέπουμε πώς έχουν τα πράγματα. Για μένα είναι σαφές ότι κοιμούνται τα κράτη-μέλη, δεν υπάρχει καμία στρατηγική ενίσχυση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, ανάπτυξη τη δική μα τεχνολογία, γιατί επιτρέπουμε την πλήρη ε, παρίσπιση των ξένων επιχειρήσεων ε, και αυτό έγινε και στη χώρα μου πρέπει να έχουμε ένα ευρετήριο των ε, πλέον νευραλγικών υποδομών στην Ευρώπη, όπως τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας ή η η πυρηνικοί σταθμή, που μπορούν όντως ε, να αποτελέσουν στόχους ε, επιθέσεων. Και έτσι θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη μέρη για την προστασία τους. Μετά, έχουμε απαριθμίσει τις συμβάσεις που έχουν περάσει από τις ε, διοικήσεις μας με διάφορες ε, φές επιχειρήσεις από Ρωσία, Κίνα και αλλού που υποτίθεται ότι είναι πάροχοι ε, υπηρεσιών ασφαλείας στον κυβερνοχώρο που μάλλον στην πράξη είναι κυβερνοκατάσκοποι. Εγώ πιστεύω ότι ούτε καν έχουν γνώση του φαινομένου αυτού οι εθνικές κυβερνήσεις. Βλέπω να περνάνε από τα χέρια τους τέτοιες συμβάσεις, δείτε, στη χώρα μας, στην Πορτογαλία. Εξαφανίστηκαν δισεκατομμύρια σε μία offshore και τελικά βρέθηκε ότι είχε εμπλακεί ένας ε, εμπειρογνώμονα τη κυβερνοασφάλεια. Μπορεί να είναι και εγκληματία, αλλά κανεί δεν ενδιαφέρεται. Ε, πήγαμε με την ε, αντιπροσωπεία τη ΛΥΜΠΕ στην Ιαπωνία και είδαμε ότι εκεί η προστασία, το EDPR, είναι το μοναδικό σύνολο ε, διεθνώ αναγνωρισμένων προτύπων. Και στην Ιαπωνία είναι διατεθειμένοι να τηρήσουν αυτά τα πρότυπα γιατί θέλουν να διατηρήσουν τη θέση τους στην ευρωπαϊκή αγορά. Αν θέλουμε λοιπόν έχουμε τα μέσα να διασφαλίσουμε τη συμμόρφωση τη Ιαπωνία, των ΗΠΑ, οποιοδήποτε άλλο θέλει να δραστηριοποιείται στην ευρωπαϊκή αγορά. Άλλοι δεν έχουν ε, καμία ιδέα. Ο καθένα κάνει τα δικά του. Το θέμα είναι αν εμεί θα αξιοποιήσουμε τη δύναμη που έχουμε στα χέρια μα, την πρόσβαση δηλαδή στην αγορά μα, για να διασφαλίσουμε την τήρηση του EDPR όχι μόνο από εμάς αλλά και από όλους τους υπόλοιπους. Αυτό βέβαια απαιτεί πολιτική ισχύ. Αν οι κυβερνήσεις δεν κατανοούν καν το διακύβευμα, τι να πω. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Ε, πολύ φοβάμαι όμως ότι ακόμα βρισκόμαστε στα πρώτα βήματα. Ευχαριστώ. I will be very brief. Thank you, Chair. And thank you for your question. The truth is that there are a lot of national interests in this field. So... Είμαι πολύ σύντομος. αυτά που προτείνουμε είναι το να έχουμε μια πιο ευρωπαϊκή τοποθέτηση, γιατί νομίζουμε ότι αυτό είναι σημαντικό. Και νομίζω ότι αυτό το θέμα της κυβερνό άμυνας έχει σχέση με το στρατό, με την άμυνα. Συνήθως αυτά είναι θέματα εθνικών κυβερνήσεων. Και πρέπει αυτό να το εκχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά τέλος πάντων έχουμε αυτή εδώ την απαρίθμηση ε, των σημαντικών αποδομών. Όχι όμως δεν έχουμε κάποιο είδους απαρίθμηση, καταγραφή των εθνικών συμβάσεων, αλλά πρώτα πρώτα θέλουμε η πολιτική δημοσίων συμβάσεων να εναρμονιστεί. Να μπορούμε έτσι να έχουμε ανταγωνισμό σε περισσότερες ε, χώρες. Γιατί μπορεί κάποια εταιρεία να θέλει να προτείνει κάτι άλλο σε, κάτι σε μια χώρα και κάτι άλλο σε άλλη. Οπότε θα πρέπει για την κυβερνοασφάλεια να υπάρχουν τέτοιες ρυθμίσεις. Κάτι σαν το EDPS να φτιάξουμε. Δηλαδή να στείλουμε το μήνυμα και να καλύψουμε και ξένες εταιρείε για να έχουμε ποιοτικά προϊόντα. Γι' αυτό λέμε να τυποποιήσουμε τις διαδικασίες αυτές. Οι υπηρεσίες πληροφοριών βέβαια έχουν εθνικά πρότυπα, Άρα θα πρέπει να έχουμε ευρωπαϊκά πρότυπα για να αξιοποιήσουμε τις ε, πληροφορίες. Γι' αυτό λέμε να αναβαθμίσουμε την ενίσα ακριβώς γιατί είναι σημαντικό να έχουμε ευρωπαϊκή θέση. Thank you. Thank you very much for the presentation. Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εισήγηση και για τις απαντήσεις σας, κύριε Ριβέρα. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Είναι αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δίμευσης. Να δώσουμε το λόγο αμέσως στην εισηγήτρια την κυρία Γκρισμπέκ και να μας παρουσιάσει τι γίνεται με το θέμα, με τις τροπολογίες που είναι αρκετές. Και στη συνέχεια βέβαια να λάβουν τον λόγο οι άλλοι συνάδελφοι. Κυρία Γκρισμπέκ, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Συνάδελφοι, σας προσέξω πριν από ένα μήνα περίπου αυτό το σχέδιο έκθεσης όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά την αμοιβή αναγνώριση δέσμευσης και δίμευσης των σχετικών αποφάσεων. 25 ε, Δεκάτου έληξε η προθεσμία για τις τροπολογίες κατετέθησαν 210 δηλαδή συνέβαλαν όλες οι πολιτικές ομάδες για την πρόταση καονισμού δηλαδή διαμορφώθηκε η συνένεση γύρω από αυτόν τον κανονισμό το σχέδιο κανονισμού λοιπόν πολύ σημαντικό πρόκειται δηλαδή για ένα κείμενο κλειδί. Θα καταπολεμήσουμε τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και το οργανωμένο έγκλημα στην Ευρώπη. Δύσκολο να αναφέρω μία-μία ε, της τροπολογίας που είναι 210. Πάντως εκ πρώτης ε, απόψεως και θα τα συζητήσουμε και την επόμενη εβδομάδα ε, οι σκιώδες συζητητές και με εκείνους θα τα συζητήσω εις βάθος και θα βρούμε συμβαστικές τροπολογίες. Αλλά έχω κάποιες γενικότερες ε, παρατηρήσεις να σας τα πω πριν οι συνάδελφοι μιλήσουν. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν κάποιες τροπολογίες για την βελτίωση της ταχύτητας, την ε, αποτελεσματικότητα των ε, διαδικασιών αναγνώρισης αποφάσεων που αφορούν ε, το, το, τη δέσμευση και κατάσχεση προϊόντων εγκλήματος. Χρειάζεται δηλαδή συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων αρχών. Υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών. Βεβαίω και συμφωνώ με τη σχετική προσέγγιση. Και όλες οι τροπολογίες προς τα εκεί πηγαίνουν. Και είναι σημαντικό αυτό γιατί χρειάζεται ένα λειτουργικό νομοθέτημα να είναι συγκεκριμένο, να υπάρχει διαδικασία αποτελεσματική, γρήγορη και έτσι οι διοικητικές αρχές, οι δικαστικές αρχές, να μπορούν να δράσουν άμεσα. Κάθε φορά που έχουμε χρήματα ή αντικείμενα τα οποία είναι προϊόν διάπραξης εγκλήματος. Πρώτο αυτό. Μια δεύτερη δόση παρατηρήσεων. Έχουμε διάφορες τροπολογίες οι οποίες προέρχονται από όλο το πολιτικό φάσμα. Και οι συναδελφοί εκεί έχουν σταθεί στα θεμελιώδη δικαιώματα. Δηλαδή στο ότι να έχουμε την ε, ε, ρήτρα μη αναγνώριση και μη εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων για δέσμευση και δίμευση όταν παραβιάζονται τα θεμελιώδη δικαιώματα. Χαίρομαι που το ζητούν αυτό όλοι οι συνάδελφοι, γιατί το Κοινοβούλιο για αυτά θέλει εδώ και πολλά χρόνια. Μπράβο, συναδέλφους. Με τις τροπολογίες τους ακριβώς αυτό και τονίζουν. Τρίτη σειρά παρατηρήσεων, ας πούμε, ότι έχουμε κάποιες τροπολογίες που αφορούν το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού. Προτείνεται μια διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής. Απλά φορολογικής, αστικής, διοικητικής. Πολύ σημαντικό και αυτό. Αλλά τα θέματα βέβαια είναι κάπως πιο δύσκολα γιατί είναι δομικού, διαρροτικού χαρακτήρα. Οπότε να τα συζητήσουμε και να βρούμε ένα modus vivendi και να είμαστε έτσι συνεπείς σε σχέση με ε, το σώμα του κειμένου. Και αυτό το συζητήσουμε με τους σκιώδες ηγητές. Θα προσπαθήσουμε να συμφωνήσουμε όσον αφορά το θέμα της προληπτικής δίσμευσης, δέσμευσης και δίμευσης και πριν επέλθει κάποια καταδίκη δηλαδή. Επίσης, τέταρτη κατηγορία τροπολογιών και παρατηρήσεών μου θα πρέπει σε όλη την Ευρώπη, σε όλη την να έχουμε την καλύτερη δυνατή διαχείριση αυτών των ε, δεσμευμένων και δημευμένων ε, αγαθών. Επίση, προβλέπει πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάποια επαναχρησιμοποίηση για κοινωνικού σκοπού. Για αποζημίωση θυμάτων, των οικογενειών των θυμάτων, για τι επιχειρήσει που έχουν πέσει θύμα του οργανωμένου εγκλήματο ή τη τρομοκρατία. Οπότε να χρησιμοποιηθούν οι σχετικοί πόροι για να καταπολεμηθεί το οργανωμένο έγκλημα. Και πολλές τροπολογίες προς τα εκεί το πάνε. Πολύ σημαντικό αυτό να τις επεξεργαστούμε και να τις προωθήσουμε. 98, τόσο της εκατό, Δηλαδή σχεδόν 100 της εκατό των ε, προϊόντων εγκλήματος δεν κατάσχονται. Μένουν στα χέρια των εγκληματιών. Ε, είναι, καταλαβαίνει την τάξη μεγέθου του προβλήματο. Αυτά για το πνεύμα που διαπνεί αυτές τις 210 τροπολογίες. Σας είπα τις παρατηρήσεις μου, αυτές τις τέσσερις κατηγορίες παρατηρήσεων. Και πρέπει να ακούσω τις απόψεις συνάδελφοι για να δούμε πού θέλετε να σταθούμε, πού υπάρχουν ερωτηματικά όσον αφορά πιο συγκεκριμένα τις τροπολογίες. Πρόκειται και ένα νέο νομοθέτημα. Και αυτό θα είναι κομμάτι των όπλων μας, του πλουστασίου μας, για να καταπολεμήσουμε τρομοκρατία και οργανωμένο έγκλημα. Και ελπίζω η σωστή με τώρα δουλειά να συνεχιστεί. Κύριε Κρισμπέκ, σας ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα. Α, εδώ έχουμε όλους τους κοιόδους, οπότε να τους δώσουμε τον λόγο. Κύριος Πουλιέζε πρώτος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κατόπιν της ανάλυσης της εισηγήτριας για το πνεύμα αυτών των τροπολογιών είμαι απόλυτα ικανοποιημένος το ότι όλες οι πολιτικές πτέρυγες έχουν συγκλίνει για τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδίου κανονισμού της Κομισιόν. Θα πρέπει πάντως να υπάρξει σωστή διαχείριση αυτών των ε, προϊόντων εγκλήματος. Θα πρέπει αυτά τα προϊόντα εγκλήματος να χρησιμοποιηθούν υπέρ των κοινοτήτων που έχουν πληγεί από εγκληματίες και τρομοκράτες. Ε, νομίζω ότι το Ιταλικό δίκαιο αποτελεί πράγμα προς μίμηση γιατί η δέσμευση και η δημευστή γίνεται μόνο για να μην έχουν οι εγκληματίες τα οικονομικά αυτά όλα στοιχεία αλλά για να χρησιμοποιηθούν όπως σας είπα υπέρ αυτών των κοινοτήτων και στο 101 στην τροπολογία 101 ε, ε, το, αυτό το έχουμε προτείνει και το ξαναπροτείνουμε με ίσως καλύτερη διατύπωση το 253 επίσης 199 ε, 250 2 αφορούν το, την παρα 32 και το άρθρο 31 παράγραφος 4 όσον αφορά το τι πρέπει να κάνουμε για αυτά τα αγαθά, τα, τα προσωπικά στοιχεία τα οποία έχουν δεσμευθεί δημευτεί. Και οπότε ελπίζω ότι θα υποστηρίξετε τις τροπολογίες μου γιατί νομίζω ότι είναι θετικός αυτός ο οργανισμός. Είναι συγκεκριμένο αυτό το μήνυμα και αποτελεί πραγματική έκφραση αλληλεγγύης και μπορούν όλα αυτά τα περιουσιακά στοιχεία να αποζημιώσουν τους πληγέντες από το έγκλημα και έτσι θα έχουμε κάνει ε, ε, το καθήκον μας αλλά αυτό να απευθυνθεί και προς τους αστυνομικούς που κατά την εκπλήρωση του καθήκοντος έχουν υποστεί κάποια βλάβη και ακόμα και αναπηρία. Θα πρέπει επίσης να δούμε για το έγκλημα και την τρομοκρατία ότι θα πρέπει σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα κράτη-μέλη αυτά τα οικονομικά στοιχεία να τα βάζουν, να τα, να τα εντάσσουν στον κοινοτικό προϋπολογισμό και να αξιοποιούνται ε, υπέρ της Europol και των ε, συναρμοδίων αρχών. Έχουμε το 3 παράγραφος 1 και οπότε προτείνω να, ε, προσθέσουμε εδώ τα αγαθά, ε, συγγνώμη, τα εγκλήματα λαθρεμπορίας και τα εγκλήματα κατά της πνευματικής και βιομηχανικής διοκτησίας όπως ε, προβλέπεται στην Ιταλία. Τέλος. Σε σχέση με το άρθρο 31 παράγραφος 2 εδάφιο Β έχουμε την τροπολογία 246 και λέμε για το τι, πώς θα πρέπει να εκτελείται η απόφαση ε, η σχετική με ε, τα ποσά αξία πάνω από 10 ευρώ. Βλέπω ότι εδώ όλοι συμφωνούν με αυτή την ε, πρόταση, με αυτό που πρότεινε ο κύριος Παύλ και η κυρία Γκραπίνη με την τροπολογία 244 και επίσης ευχαριστώ ως και ο του ΕΛΚ ε, τους ε, άλλους συναδέλφους για αυτές τις τροπολογίες ιδίως τον κύριο Μέλο γιατί έχουμε 89, 92, 150 και άλλες τροπολογίες ε, τις οποίες μαζί κατεβάσαμε και ελπίζουμε να συμφωνήσει η συγκήτρια. Και επίσης έχουμε και την οδηγία 214 για την αμοιβαία αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων στα πλαίσια της δικαστικής συνεργασίας ε, στην ποινική δίκηση. Οπότε θα πρέπει ίσως να δανειστούμε αυτή την αμοιβή αναγνώριση για αυτές τις αποφάσεις χαίρομαι για ε, τα όσα γίνονται μέχρι τώρα και ελπίζουμε η αγαστή συνεργασία να εξηγηθεί και στις επόμενες συναντήσεις μας. Ευχαριστώ εσείς κύριε Μπάνερτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτον επιθυμώ να ευχαριστήσω την κυρία Γκρίσπεκ, η συγγήτρια και όλους τους κοιόδους εισηγητάς που εργάστηκαν για το θέμα αυτό. Νομίζω θα μπορέσουμε να συμβαστούμε σε πολλά από τα θέματα που αναφέρθηκαν. Έγινε συντονισμός μεταξύ των γραφείων μας για το θέμα που προέρχεται για το ε, ποσόν μάλλον προέρχεται από την δίμευση και ανάμεσα βέβαια στην ε, εκδούσα χώρα και την εκτελούσα χώρα. Από τα πιο σημαντικά είναι να γίνει σεβαστό και το πεδίο εφαρμογή του κανονισμού που αναφέρεται μοναχά στις ποινικέ διαδικασίες του 81-2α της συνθήκης. 82-1α διορθώνει ο Δερμηνέας. Και στις ε, σκιώδεις ε, συναντήσεις που θα γίνουν από την επόμενη εβδομάδα σε ό,τι αφορά την μη εκτέλεση των ε, αποφάσεων δέσμευση, πρέπει να κάνουμε σαφή διάκριση ανάμεσα σε υποχρεωτικούς νομικούς λόγους και σε αυτούς που είναι ε, κατ' επιλογή, όπως το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Χρειάζεται ευθυγραμμισμένη νομοθεσία για την αμοιβή αναγνώριση σε όλες τις χώρες της Ένωσης και να υπάρχει πλήρης προστασία και εγγύηση των θεμελιδών δικαιωμάτων. Εγώ θα εργαστώ ιδίω για την προστασία των ενδιαφερομένων μερών. Είμαι βέβαιο ότι θα καταλήξουμε σε ορθές συμβαστικέ τροπολογίε, όπω είπα στην αρχή και ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε τον μηχανισμό πολύ αποτελεσματικό για την καταπολέμηση του εγκλήματος και, την, και χρηματοδότηση τη τρομοκρατία. Η κυρία Μακοβέη Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητή Ναταλή Γκρίσπεκ, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη που εν τέλει θα καταλήξουμε σε κανονισμό ο οποίος θα είναι άμεση εφαρμογή σε όλες τις χώρες μέλη και με τον οποίο οι διαταγές δέσμευσης και δίμευση θα καταστούν εκτελεστές σε άλλες χώρες μέλη. Η αμοιβαία αναγνώριση λοιπόν και ε, εκτελεστότητα των αποφάσεων δέσμευσης και δίμευσης. Αυτό είναι το θέμα άλλωστε. Βεβαίως υπάρχει ένας αριθμός τροπολογιών που έχουμε καταθέσει ε, ορισμένοι εξημών, ορισμένες τις οποίες έχω καταθέσει εγώ για την ε, εν λόγω έκθεση αναφέρονται στην εφαρμογή του κανονισμού για την αναγνώριση των αποφάσεων ε, δέσμευσης και δίμευσης για όλες τις ε, περιπτώσεις, όλες τις υποθέσεις εκτεταμένης δέσμευσης και δίμευσης και δίμευσης που γίνονται ε, εκτός καταδίκης και στην βάση αστικών αποφάσεων. Επίσης, δημεύσει στα, στα χέρια τρίτων και επομένως όλα τα θέματα δέσμευσης και δίμευσης είναι αναγκαίο να καλυφθούν ώστε να μπορούν να ανακτώνται περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχουν αποκτηθεί μέσω απατών, ε, ξεπλήματος βρώμικου χρήματος ή με άλλα εγκληματικά μέσα. Άλλη τροπολογία δική μου αναφέρεται στις ξεκάθαρες προθεσμίες καθώς και στις ε, τυποποιημένες μορφές για όλες αυτές τις εθνικές διαταγές. Θα πρέπει όλες να είναι ίδιες, να έχουν τον ίδιο μορφότυπο, έτσι ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε περιττή καθυστέρηση, παρανοήσεις, εσφαλμένη ε, συμπλήρωση κάποιων ε, εντύπων που να οδηγήσει σε εσφαλμένη εφαρμογή από την άλλη μεριά. Χρειάζονται λοιπόν τυποποιημένα έγγραφα για όλες τις χώρες μέλη και ώστε όλες οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές που εκδίδουν τις σχετικές ε, αποφάσεις να μπορούν να τις συμπληρώνουν ορθά. Επίσης, μεταξύ των λόγων αναγνώρισης και εφαρμογής των εθνικών αποφάσεων δέσμευσης και δίμευσης, προτείνω εγώ οι λόγοι απόρριψης να μην είναι η ασυλία. Εάν δηλαδή στην χώρα μέλος όπου θα είναι εκτέλεση υπάρχουν διατάξεις του νόμου που αναφέρονται σε προνόμια ή ασυλίες ορισμένων αξιωματούχων ή βουλευτών η ασυλία να εξαιρεθεί από τους λόγους μη εφαρμογής όσον αφορά τα δικαιώματα των θυμάτων Σημαντικό είναι να αποζημιώνονται τα θύματα. Εγώ γνωρίζω το Ιταλικό σύστημα όπου μέρος των δημευωμένων χρημάτων χρησιμοποιείται για κοινωνικές αποζημιώσεις των θυμάτων για να μπορέσουν να βρουν δουλειά κλπ. Είναι σημαντικό αυτό να λυθεί υπόψη. Περιλαμβάνεται και στην οδηγία περί δέσμευσης και δίμευσης περιουσιακών στοιχείων που εγκρίθηκε το 2014. Αυτά είναι ολίγης σχετικά με τις τροπολογίες μου. Αλλά θα συνεχίσω να τα συζητώ στη συναντήση με τους άλλους και όλους Η κυρία Σπινέλη. Και πάλι ευχαριστούμε Ναταλή Κρισμπέτη, για αυτή την τόσο εύστοχη έκθεση και κυρίως για αυτές τις ε, τροπολογίες ε, αυτές που πρέπει να προστατεύσουν τα δημοσιονομικά δικαιώματα, τις ε, δικονομικές εγγυήσεις και τι γίνεται με αυτά τα δεσμευμένα, αντικείμενα ε, αγαθά. Ότι θα πρέπει δηλαδή να πάνε στις οικογένειες, στις πληγήσεις από τους εγκληματίες και τρομοκράτες. Οπότε ο, αυτός ο κανονισμός είναι ένα πολύτιμο εργαλείο, τόσο ώστε να έχουμε πιο θωρακισμένη δίωξη του οργανωμένου εγκλήματος στην Ιταλία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο της λειτουργία της δημοκρατίας και για την καταπολέμηση της ε, παρανομίας ε, για όλη τη χώρα. Αλλά θα πρέπει να καταδείξουμε το ότι όλες οι μαφίες και η ντραγκέτα ε, εκμεταλλεύονται κάθε παρανομία και παρανομία που δεν ονομάζεται μαφιόζικη και εκεί έχουμε αναδείξει το ότι αυτές οι συμμορίες δεν είναι αίτητες και άτρωτες. Ακόμα πιο σημαντική είναι η τροπολογία 31, Ναταλή, δική σου, που προσθέτει ε, στους λόγους ε, μη αναγνώρισης αποφάσεων εκτέλεσης κάποιες καταστάσεις όπου υπάρχουν σοβαροί λόγοι. Οπότε η εκτέλεση της απόφασης θα ήταν ε, ασυμβίβαστη με το άρθρο 6 ε, λόγω των υποχρεώσεων λοιπόν της ε, συγκεκριμένης χώρας εκτέλεσης απόφασης το άρθρου 6 του, του δικαιωμάτων. Επίσης θα πρέπει τα θεμελιώδη δικαιώματα να θωρακιστούν θα πρέπει να υπάρχουν οικονομικές εγγύσεις ιδίω όσον αφορά την αμοιβαία αναγνώριση ε, και τη διαδικασία ε, κατάσχεσης και δέσμευσης και λοιπά εκτός και προ και χωρίς ποινική καταδίκης τώρα επίσης έχουμε το δικαίωμα της ενημέρωσης όλων των ε, εμπλεκομένων που θα πρέπει να κατοχυρώσουμε. Σε ευχαριστούμε και πάλι Ναταλή. Ο κύριος Κοράου. Ευχαριστώ. Και εγώ να ευχαριστήσω την ε, εισηγήτρια για την αξιόλογη εργασία της και ακριβώς όπως είπαμε πολλές φορές και αυτός ο κανονισμός και άλλες νομοθετικές προτάσεις που έχουν πέρασει στο Κοινοβούλιο ε, ε, στόχο έχουμε να χτυπήσουμε την περιουσία αυτών των ε, εγκληματιών για να μην μπορούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, τη δράση τους τέλος πάντων. Και είπαμε τις τροπολογίες θα πρέπει να είναι γρήγοροι και και αποτελεσματική η εκτέλεση των αποφάσεων και αυτό θα πρέπει να υπάρχει αμοιβαία αναγνώριση. Θα πρέπει να υπάρχουν σχετικέ εγγυήσει και αυτό σε κάθε φάση της ε, διαδικασίας δέσμευσης, δίμευση και πέραν της ε, ποινική καταδίκη. Να υπάρχει επίσης ε, κατάσχεση ισχύρα τρίτων κλπ. κλπ. Οπότε θα πρέπει να έχουμε μια διαδικασία που να εφαρμόζεται από τους εθνικούς δικαστές και να έχει τα χαρακτηριστικά της ποινική διαδικασίας. Βέβαια το θέμα είναι το δικαστήριο που εφαρμόζει την νομοθεσία να έχει ποινικέ αρμοδιότητες, να είναι ποινικό δικαστήριο. Οπότε θα πρέπει να δούμε τι έχει γίνει στην Ιταλία για να καταπολεμήσουμε το επιθετικό οργανωμένο έγκλημα. Ε, πρόκειται για ένα εργαλείο που είναι πολύ αποτελεσματικό. Οι Ιταλικές αρχές το χρησιμοποιούν ακόμα για να πλήξουν τις μαφίες. Και αυτό είναι το να τις πλήξουν όσον αφορά την περιουσία τους. Να, που τώρα έχουμε την ευκαιρία και εμείς να νομοθετήσουμε σχετικά. Έτσι δρούν οι μαφίες και διασυνοριακά και δυστήριση στην νόμιμη οικονομία για όλα τα κράτη-μέλη. Οπότε θα πρέπει οι, οι, οι αρχές να σταματήσουν αυτές τις οργανώσεις από τη διείσδυση στην νόμιμη ε, οικονομία που είναι ένα καρκίνωμα. Οπότε θα κάνουμε διαπραγματεύσει, θα αποκρισταλώσουμε θέση στο Κοινοβουλίου και αυτό θα πρέπει να γίνει το συντομότερο για να περάσει όσο γίνεται πιο σύντομα αυτό ο σημαντικό κανονισμό. Επανέρχομαι στην εισηγήτρια. Κυρία και εσεί, μήπω θέλετε να προσθέσετε κάτι. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλες και όλους τους συναδέλφους για τις τροπολογίες καθώς και για τις παρεμβάσεις τους, στη συζήτηση εννοώ. Οι διαφορετικές ιδέες που κατέθεσαν, οι παρατηρήσεις τους, βεβαίως θα τις επεξεργαστούμε με λεπτομέρεια. Δεν θα επανέλθω στα όσα είπατε, έχω σημειώσει όμως η γενική ιδέα πάντως όλες και όλοι συμφωνείτε στο γεγονός ότι εκφράζεται την θέληση ε, να θεσπιστεί μια ισχυρή πολιτική για το σύστημα αποζημιώσεων των θυμάτων. Η ιδέα επίσης, όπως είπε ο κύριος Πολιέσε προηγουμένως, η δέσμευση και η δίμευση είναι σημαντικά, αλλά χρειάζεται και ένα σύστημα ανάκτησης από την Ευρωπόλ. Θα το δούμε με λεπτομέρειες. Το ίδιο για τα κίνητρα απόρριψης. Για πρόσωπα προνομιούχα ή που χαίρουν ασυλίας. Θα τα ε, συζητήσουμε και αυτά. Επίσης, βεβαίως έχω σημειώσει πολλά πράγματα από τα όσα είπατε και αυτά τα, αυτές οι σημειώσεις θα τροφοδοτήσουν και τη συζήτηση της Τρίτης. Μου άρεσε αυτό που είπε κάποιος και που δίνει νόημα στο κείμενο ότι δηλαδή πρόκειται για την υπεράσπιση της δημοκρατίας. υπεράσπιση δημοκρατίας, ευρωπαϊκής δημοκρατίας, με τα συστήματα άσκησης διώξεων κατά των μαφιών που δεν γνωρίζουν σύνορα και που μας αναγκάζουν να προβλέψουμε ευρωπαϊκή λύση αποτελεσματική με μηχανισμούς που θα επιτρέψουν με ακόμα μεγαλύτερη αυστηρότητα την δίωξη των εγκληματικών δραστηριοτήτων. Ευχαριστώ και πάλι όλες και όλους τους συναδέλφους. Συμφωνώ με την φόρμουλα του κ. Κοράου δηλαδή να προχωρήσουμε ταχαίω σε συμβαστικές τροπολογίε για να προχωρήσουμε μετά στην ψηφοφορία και αναμένω τη συνεργασία μαζί σας και την θεσμική συνεργασία με το Συμβούλιο Υπουργών. Αυτά με λίγα λόγια, αλλά βεβαίω η ουσία είναι η υπεράσπιση των θυμάτων αλλά και κυρίως των δημοκρατικών αρχών τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Γκρίσπε και ευχαριστώ και εσάς οι κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ερχόμαστε αμέσως στο επόμενο θέμα της σημερινής διατάξεως που είναι η παρουσίαση της συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μπαρμπούδα, ε, Μπαρμπάδος, Αντίγουα και Σεϊχελών και Μαυρικίου. Η νομοθετική διαδικασία επιτρέπει μόνο την εξέταση τροπολογιών. Η συγητής μα είναι ο κύριο Πάβελ. Θα δώσω πρώτα το λόγο στους εκπροσώπου Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να εξηγήσουν και μετά στον εισηγητή και σε όσους ευρωβουλευτές θέλουν να παρέμβουν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Αυτές οι συμφωνίες ατροποποιούν τις συμφωνίες που είχαν απογραφεί το 2009 ε, για την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βροχή διαμονή βασίζονται στις ε, ε, οδηγίες 2014 και βασίζονται σε ορισμένες τεχνικές τροποποιήσεις. Η βραχία διαμονή γίνεται πλέον 90 ημέρες σε οποιαδήποτε περίοδο 180 ημερών και έτσι ευθυγραμμίζεται με την Συμφωνία Σέγγεν και τις υπόλοιπες ε, αυτές συμφωνίες. Δεύτερον, τροποποιείται η τελική διάταξη για την αναστολή και έτσι ε, ευθυγραμμίζεται με τις συμφωνίες δεύτερης γενιάς για την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης που υπογράφηκε το 2009. Και το community γίνεται union, από κοινότητα πάμε σε ένωση. Μετά, Έχουμε ε, κάποιες κοινέ διακηρύξεις για τις ε, τρίτες χώρες και για την προσδιορισμό του διαστήματος της βραχίας διαμονής. Να σας ενημερώσω ότι έχει συμβεί από το 2010. Το Συμβούλιο πλέον έχει υιοθετήσει αποφάσεις για την ε, υπογραφή του στις 6 Νοεμβρίου και ο κύριος Ρούιτε έστειλε επιστολή το καλοκαίρι στον Πρόεδρο και εξετάζουμε αντίστοιχες ε, Τραποποιήσει με τη Βραζιλία. Έχουν οριστικοποιηθεί οι διαπραγματεύσει και έχουμε δύο διαδικασίες, μία για τα κανονικά διαβατήρια και μία για τα διπλωματικά. Έχουν ξεκινήσει από τα τέλη Οκτωβρίου. Αυτά ευχαριστώ. Thank you very much. Now I give the floor to the reporter, Mr. Pavel. Ο εισηγητής, ο κύριος Πάβελ, ευχαριστώ πολύ και την Επιτροπή. Χαιρετίζουμε την πρόταση της Επιτροπής για την για τις ε, αναφερμένες συμφωνίες με τις έξι αυτές ε, χώρες. Δεν θέλω να τις επαναλάβω. Οι συμφωνίες αυτές λοιπόν για την απαλλαγή υποχρέωση θεώρησης ε, για βραχίες διαμονή αφορά, αποτελεί το αποκορύφωμα των διαπραγματεύσεων με αυτές τις χώρες. Και έτσι παρέχουν τη δυνατότητα ε, να ταξιδεύουν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των έξι τον χωρών χωρίς θεώρηση για μια περίοδο 90 ημερών ε, σε οποιαδήποτε περίοδο 180 ημερών. Καλύπτονται όλες οι κατηγορίες ατόμων, κανονικά διαβατήρια, διπλωματικά, αξιωματούχοι, για όλους τους σκοπούς, εκτός από τους ε, σκοπούς ενέργειες επαμοιβή. Θα ήθελα να επισημάνω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα τροποποιήσουν όλες τις συμφωνίες όταν το σύστημα εισόδου-εξόδου θα είναι επιχειρησιακό. Για την Βουλγαρία και την Ρουμανία που δεν είναι ακόμα μέλη της ΕΝΓΕΝ, με τις διαπραγματεύσεις εισόδου-εξόδου ε, θα έχουν μια νέα ευκαιρία, ήδη έχουν παθητική πρόσβαση το ερώτημά μου λοιπόν είναι πώς αυτές οι αλλαγές ε, θα επηρεάσουν τις εξελίξεις. Ε, ε, Ευχαριστούμε. Η κυρία Βεργιά. Ναι, δεν ήθελα να πάρω το λόγο. Γιατί είναι καθαρά τεχνικός αυτός ο φάκελος. Πρόκειται για απλές προσαρμογές και τελικά διευκολύνουμε την ελεύθερη ε, κυκλοφορία των συμπολιτών μας που θέλουν να πάνε διακοπές στα πολύ ωραία αυτά νησιά. Κάνα πρόβλημα λοιπόν με όλα αυτά. Δεν νομίζω ότι ε, υπάρχει κάποιο άλλο ζήτημα. Όμως, άκουσα, γιατί είχα και την μεγάλη χαρά με την κυρία Γκάμπριελ να εργαστούμε από κοινού από αυτών των ε, συμφωνιών και είχαμε επιμείνει συστηματικά αυτές οι συμφωνίες να μας υποβληθούν όταν θα έχουν εφαρμοστεί. Και άκουσα ότι υπάρχει συμφωνία με τη Βραζιλία που μόλις ατέθησε ισχύ στις 31 Οκτωβρίου. Μήπως λοιπόν η Επιτροπή ε, συνεχίζει να κοροϊδεύει το Κοινοβούλιο. Πρέπει τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου να γίνονται σεβαστά και να μην ζητάτε τη γνώμη μα και την έγκρισή μας κατόπιν εορτή. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι σωστό. Το έχουμε αναφέρει και ε, στην ε, συνεδρία των συντονιστών. Πρέπει να υπάρξει επίσημη διαμαρτυρία εναντίον του Κοινοβουλίου ως προς αυτό το ζήτημα. Νομίζω ότι έχει γίνει και από την κυρία Γκάμπριελ πολλές φορές. Καλό θα ήταν λοιπόν κάποια στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη αυτήν την κατάσταση. Εμείς είμαστε εδώ για να κυρώνουμε αυτές τις συμφωνίες ε, εκ των προτέρων. Αλλιώς δεν έχει κανένα νόημα και το κείμενο των αισθητικών. Ευχαριστούμε κυρία Βαλέρο. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω σου ειδικά. Βάλτε λοιπόν τα ακουστικά σας. Εμείς ε, στους πράσινους φυσικά και στηρίζουμε την ε, απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για μια σειρά χωρών. Θέλουμε να έρθουν όσο γίνεται περισσότερα εμπόδια μεταξύ των χωρών. Τα ανοιχτά σύνορα είναι κάτι το θετικό, όχι μόνο για την Ευρώπη αλλά και για όλο τον κόσμο. Βέβαια αυτό επιτρέπει να αποκτήσουμε και πιο ανοιχτές κοινωνίες και ε, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αλλού να δημιουργήσουμε δεσμούς μεταξύ διαφορετικών κοινωνιών. Καθώς έχει ήδη υπάρξει απαλλαγή υποχρέωσης θεώρησης για τόσες πολλές χώρες και ελπίζουμε να συνεχίσουμε να αυξάνουμε τον αριθμό τους, υπάρχει και ένα παράλληλο σύστημα με τις ε, άδειες εισόδου Επομένως, κατά κάποιον τρόπο, από τη μία πλευρά κερδίζουμε κάτι με την απαλλαγή υποχρέωσης θεώρησης, από την άλλη κάτι χάνουμε με αυτό το άλλο σύστημα. Ελπίζω να ακολουθήσουμε ε, την άγουσα του Κοινοβουλίου και να αφαιρέσουμε κάποια τμήματα της πρότασης της Επιτροπής, ιδίως ό,τι αφορά κάποια στοιχεία για το, την εκπαίδευση στο ETRS. Το ETS τελικά μπορεί να δημιουργήσει πιο αυστηρές προϋποθέσεις από ότι ε, η Visa. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, εδώ έχουμε να κάνουμε με μία τροποποίηση αυτών των συμφωνιών που είναι τεχνικές, τεχνικής φύσεως και λαμβάνουν υπόψη τις αλλαγές στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Μετά τη θέση σε ισχύ της νομοθεσίας αυτής το 2014. Ωστόσο, αυτές οι συμφωνίες δεν λαμβάνουν υπόψη άλλες τροποποιήσεις σε σχετικές νομοθετικές πράξεις. Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι οι συμφωνίες μας με πολλές χώρες ε, είναι παροχημένες. Έχουν δημιουργηθεί εδώ και πολλά χρόνια. Είμαι σκιώδης συζητητής και νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε το πράσινο φως σε όλες αυτές τις ε, συμφωνίες. Ευχαριστώ. Τρέφουμε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να απαντήσει στα ερωτήματα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και για το ερώτημα για τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Αυτό μπορεί να μην αποτελέσει καν πρόβλημα για τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία μέχρι το 2020 όταν θα τεθεί σε ισχύ το σύστημα εισόδου-εξοδού, γιατί και οι δύο χώρες ενδεχομένως ήδη να πληρούν όλα, όλες τις προδιαγραφές για το σύστημα Σέγγεν. Αλλά ε, μπορεί αυτό να αφορά άλλες χώρες όπως η Κύπρος και αφορά όλες ε, τις ε, συμφωνίες απαλλαγή υποχρέωση θεώρηση, που είναι 30, όχι μόνο οι 6 που εξετάζουμε σήμερα. Θέλουμε αρχικά να εναρμονίσουμε όλε τι συμφωνίε Visa Waiver και για να απαντήσω και στην κυρία Βεγζιά. Αυτέ οι συμφωνίε πλέον ευθυγραμμίζονται με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία που ήδη έχει υιοθετηθεί και από το Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο. Είναι τεχνικής φύση λοιπόν. Όπως και να έχει δεν είχαμε εντολή να πάμε παραπέρα. Όπως ξέρετε το, σύστημα, το κανονισμός του σύστημα εισόδου-εξόδου υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο μόνο τη Δευτέρα εάν δεν απαιτούνται περαιτέρω τροποποιήσει, αυτέ θα πρέπει να προταθούν ω επόμενο βήμα μετά τη θέση ισχύ του κανονισμού και για όλες τις συμφωνίες απαλλαγή υποχρέωση θεώρηση. Για το δεύτερο ερώτημά σας, Νομίζω ότι πρόκειται περί παρεξήγησης να διευκρινίσω ότι οι συμφωνίες με τη Βραζιλία δεν έχουν τεθεί σε ισχύ. ενημερώσαμε το Κοινοβούλιο ε, στην αρχή των διαπραγματεύσεων με επιστολή της 8ης Αυγούστου του κυρίου Ρούτε προς ε, τον Πρόεδρο της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Και επί τη ευκαιρία, παρότι δεν ήταν στην ημερήσια διάταξη, θέλαμε να σας ενημερώσουμε ε, για τις εξελίξεις των διαπραγματεύσεων που τώρα έχουν κλείσει. απλώς για να λάβουμε υπόψη αυτές τις τεχ... τρεις τεχνικές τροποποιήσεις που ευθυγραμμίζουν αυτές τις δύο συμφωνίες με τη Βραζιλία με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Όπως και να έχει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ακόμα υιοθετήσει τις προτάσεις για την ε, απόφαση του Συμβουλίου για την υπογραφή και την ε, ε, συναπόφαση. Όταν, εν αυτό το χρόνο θα τα στέλνουμε αυτά στο Κοινοβούλιο και στο, στο Συμβούλιο και φυσικά και θα ε, απαιτείται η έγκριση του Κοινοβουλίου. Ευχαριστούμε. Ο εισηγητής θέλει να προσθέσει κάτι, κύριε Πάβελ. Όχι. Ωραία. Η παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης προβλέπεται στις 19 ε, και 20 Φεβρουαρίου στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ Ευχαριστώ συνάδελφοι. Και τελευταίο σημείο. Στη μεσοδιάταξη, ελπίζω να είναι όλοι εδώ για να ξεκινήσουμε. Είναι η έκθεση Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την πρόοδο στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία στο πλαίσιο του μηχανισμού συνεργασία και ελέγχου. Η τελευταία έκθεση λοιπόν που δημοσιεύθηκε στις 15 Νοεμβρίου του 14 από τον Διευθυντή, William Slash. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Χαίρομαι ιδιαίτερως που έχω την ευκαιρία να σας κάνω μια σύνοψη των διεκθέσεων. Πέρσι τον Ιανουάριο οι εκθέσεις έλαβαν μια νέα προσέγγιση. Οι τωρινές εκθέσεις πρέπει να θεωρηθούν ως μια επικαιροποίηση εκείνων ε, των εκθέσεων. Έχουμε ε, καταγράψει την κατάσταση ε, μετά από 10 χρόνια για να έχουμε μια συνολική εικόνα. έχουμε εντοπίσει ένα περιορισμένο αριθμό τελευταίων βημάτων που εάν ε, καλυφθούν θα επιτρέψουν στις δύο αυτές χώρες να ε, επιτύχουν τους στόχους τους. Και μετά η Επιτροπή θα δεσμεύσει ότι πρέπει να σταματήσουν αυτοί οι μηχανισμοί. Επίσης, συντάσσεται με τον στόχο να κλείσει το CVM κατά τη διάρκεια της ε, τωρινής θητείας της Επιτροπής. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή διατηρεί τη δέσμευση να εξετάσει προσεκτικά και σε στενή συνεργασία με τις ε, ρουμανικές και βουλγαρικές αρχές και λαμβάνοντας υπόψη τις γνώμες ε, της κοινωνίας των πολιτών και άλλων κρατών μελών. Λοιπόν, οι δύο εκθέσεις για τη Βουλγαρία. Η έκθεση του Ανωρίου είχε εντοπίσει 17 συστάσεις και αυτή η έκθεση καταλήξε στο ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος. Υπάρχει νέα όθηση ε, στην διαδικασία μεταρρυθμίσεων από το Μάιο και μετά ε, με ολοκλήρωση προσπαθειών που είχαν ξεκινήσει το 2016. Έχουν τεθεί ο στόχος μια σειρά μεταρρυθμίσεων μέχρι τέλη της χρονιάς. Επίσης είχαμε την εκλογή διαφόρων δικαστικών αρχών, το οποίο δίνει ευκαιρία νέων μεταρρυθμίσεων για αμερόληπτη και επαγγελματική λήψη αποφάσεων. Για πρώτη φορά εφαρμόστηκε η αρχή του ενός δικαστή και της μίας ψήφου, παρότι υπήρχαν επικρίσεις στο παρελθόν με το προηγούμενο σύστημα την κοινωνία των πολιτών. Τα άλλα ζητήματα αφορούσαν ε, τον ορισμό ε, μελών και υπάρχει πλέον ε, ένα νέο σύνολο αρμοδιοτήτων. Μετά έχουμε την παρακολούθηση σχέση με την περσινή ανεξάρτητη ανάλυση των εισαγγελικών αρχών και τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις στο σύστημα ποινικών διαδικασιών. Γενικά εξετάσαμε και τη σημασία της ε, νομοθετικής διαδικασίας χωρίς αποκλεισμούς με διαβούλευση με τους ε, ενδιαφερόμενους φορείς. Η κοινωνία των πολιτών έχει εκφράσει ορισμένε επικρίσεις και προβληματισμούς και αυτό είναι σημαντικό τμήμα της βιωσιμότητας της μεταρρύθμισης. Η διαφθορά έχει θυγεί στην ε, έκθεση γιατί θεωρήθηκε ότι είναι πάρα πολύ αργή η πρόοδος και η βασική σύσταση είναι το πώς θα γίνει μια συνολική μεταρρύθμιση της νομοθεσίας και έτσι να υπάρχει μία αρχή που να καταπονεί την φθορά. Οπότε τώρα εξετάζει σχετικό νομοσχέδιο το Κοινοβούλιο της χώρας Οπότε θα πρέπει να περάσει αυτό ο νόμο πριν τον νέο θεσμικό όργανο υπάρξει. Στι συστάσει επίση λέμε ότι χρειάζεται να υπάρχει ένα ξεκάθαρο χάρτη πορεία για την αντιμετώπιση της διαφθοράς και κάποιους μηχανισμούς... που να αφορά τη διαδικασία καταπολέμησης Και αυτό επίσης θα πρέπει να ρυθμίσει και το ρόλο της εισαγγελία σε αυτή την προσπάθεια για να μπορέσει να υπάρξει πρόληψη της διαφθοράς. Συγκεκριμένα διαβήματα για τις συμβάσεις και έχουν ήδη αναλυθεί ενέργειε. Τώρα όσον αφορά το τελευταίο στοιχείο και πολέμηση του εγκλήματος, τον Ιανουάριο του 2017 η έκθεση ανεγνώρισε ότι έχουν εξελιχθεί τα πράγματα όσον αφορά το έγκλημα τελευταία. Το 2012 ξεκίνησε η προσπάθεια ούτως ώστε να υπάρξει μια καταγραφή τη κατάστασης και να υπάρξουν και καταδίκες σχετικά. Επίση να γίνει και κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων των εγκληματιών. Θα πρέπει πάντως οι θεσμικές μεταβολές να αποτελέσουν εγγύηση επιτυχίας αυτών των προσπαθειών. Αυτά όσον αφορά την Βουλγαρία. Δεν μπορεί να καταλήξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ε, τα πάει καλά η χώρα σαν πρώτα διάφορα κριτήρια αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει σωστή κατεύθυνση, υπάρχει πολιτική βούληση και θα ολοκληρωθούν οι μεταρρυθμίσεις, ούτως ώστε η Βουλγαρία να παρακολουθήσει και να συμμορφωθεί με αυτές τις συστάσεις. Ρουμανία τώρα. Όσον αφορά την δεκαετή προοπτική, τον Ιανουάριο καταλήξαμε στο ότι έχει σημειωθεί πρόοδος. Υπάρχουν μεταρρυθμίσεις, έχουν ολοκληρωθεί και η δικαστική εξουσία επίσης έχει επιδείξει επαγγελματισμό και ανεξαρτησία. Οπότε και είχαμε και άλλες επιδόσεις των θεσμικών οργάνων για καταπολέμηση της ε, ε, εγκληματικότητας. Είχαμε 12 συστάσεις στην έκθεση του Ιανουαρίου επί τη βάση της λογοδοσίας, επί τη βάση των ευθυνών και είπαμε ότι υπάρχουν κάποιους ρήτρες διαφύλαξης και εξασφάλιση ούτω ώστε να υπάρξει εγγύηση συνέχιση αυτών των αποτελεσμάτων. Οπότε είπαμε ότι υπάρχει πρόοδο για διάφορες από αυτέ τι ε, συστάσεις και εξετάσαμε τους επιμέρου τομεί ένα προς ένα. Όσον αφορά τι χρηστές δικαιοσύνη, εστιαστήκαμε σε διάφορα ζητήματα. Πρώτα-πρώτα είπαμε να υπάρχει ανεξάρτητο, αμυρόληπτο σύστημα όσον αφορά τον διορισμό των ε, κορυφαίων εισαγγελέων και να υπάρχει σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής της Βενετίας. Πρόκειται για πάγιο θέμα που αφορά την νομοθεσία για την τάξη της δικαιοσύνης και εδώ εκκρεμούν κάποια θέματα. Επίσης είπαμε να υπάρχει μια, ε, ένας κώδικας ε, συμπεριφοράς, διοντολογίας να περάσει το Κοινοβούλιο, πέρασε τώρα και να δούμε όταν εφαρμοστεί ο κώδικας διοντολογίας κατά πόσον θα υπάρξουν ε, οι επιθυμητές συνέπειες. Σταθερότητα όσον αφορά την νομοθεσία, τους κώδικες, να υπάρχει διαδικασία νομοθεσίας που να είναι κρυστάλλινη για να ληφθεί υπόψη το ότι θέλουν δικαστικέ αρχέ για εμπλεκομένοι. Άρα έχουμε πρόοδο σε κάποια μέτωπα, αλλά είχαμε και κάποια γεγονότα που οδήγησαν σε αστάθεια όσον αφορά τη μεταρρύθμιση των κωδίκων ιδίω. Όσον αφορά το διάταγμα 13 του Φεβρουαρίου. Και είχαμε επίσης διάφορα μέσα τα οποία ελήφθησαν χωρίς να έχουν περάσει από συζήτηση και διαβούλευση τώρα υπάρχει μια ειδική επιτροπή του Κοινοβουλίου για να υπάρξει διάλογος με την δικαιοσύνη. Ίσως έτσι έχουμε περισσότερη προβληψιμότητα και περισσότερη συνενετικότητα στην διαδικασία. Εάν μεταρρυθμιστούν όπως πρέπει οι δικονομίες, αυτό θα είναι καλό δείγμα. θα πρέπει να μετρήσει γνώμη των δικαστών. Αυτό επίσης είναι ένα κριτήριο. Τώρα, το Δικαστικό Συμβούλιο τον Ιανουάριο άρχισε τη θητεία του. Θα έπρεπε από την αρχή να προσαρμοστεί στην αλλαγή του τοπίου, αλλά έχουν ληφθεί σημαντικές αποφάσεις. Ακαιρεώτης. Και πάει μια νέα πρωτοβουλία πρόληψη, ούτω ώστε να μην έχουμε σύγκρουση συμφερόντων σε σχέση με τις δημόσιες συμβάσει. Τα πρώτα αποτελέσματα ήδη υπάρχουν. Διαφάνεια στον κοινοβουλευτικό έλεγχο σε θέματα όπως σύγκρουση συμφερόντων. Ακόμα εκκρεμούν κάποιες υποθέσεις. Το Κοινοβούλιο ακόμα δεν έχει επιβάλει τις σχετικές κυρώσεις ούτως ώστε να έχουμε πρόοδο και για αυτήν την σύσταση. Όσον αφορά την διαφθορά υψηλού επίπεδου, τον Ιανουάριο είχαμε τη σχετική σύσταση και είπαμε ότι έχουμε μόνο μία τέτοια σύσταση όσον αφορά τη λογοδοσία, την άρση ασυλιών στο Κοινοβούλιο και έχουμε σύσταση κάποιων κριτηρίων για την, για την άσκηση ποινική δίωξη. Και εδώ επειδή έχετε βελτίσει η κατάσταση καταλήξαμε. Τώρα όσον αφορά την διαφθορά, γενικά θεωρούμε ότι είναι θετική η εθνική στρατηγική, αλλά και εδώ χρειάζονται περισσότερες προσπάθειες και περισσότερη έντονη πολιτική βούληση. Τελευταία σύσταση αφορά την υπηρεσία για την διαχείριση των ε, κατεσχεμένων και δεσμευμένων. Και αυτό ε, αποτελεί σήμα πρόοδου. Άρα βλέπουμε πρόοδο για πολλές συστάσεις. Και υπάρχουν ακόμη και επισεκκριμότητες που νομίζαμε ότι είναι κεκτημένα. και προβληματιζόμαστε για το αν θα ισχύσει τελικά η εξαρτησία τη δικαιοσύνη. Χρειάζεται συνεργασία των διαφορών θεσμών οργάνων στη χώρα. Και χρειάζεται η πολιτική βούληση ούτω ώστε να αξιοποιηθούν τα όσα έχουν επιτευχθεί. Δικαστική εξαρτησία. ούτω ώστε ό,τι συστάσει δεν έχει εκπληρώσει, να, η χώρα να το κάνει στο εγγύ μέλλον. Άρα μπορούμε να θεωρήσουμε ότι με τις δύο εκθέσεις ε, ε, κάνουμε το πρώτο βήμα, θα κάνουμε άλλες εκθέσεις του χρόνου και θα συνεργαστούμε, θα παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις στις δύο αυτές χώρες. Ευχαριστώ πολύ κύριε εκπρόσωπε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τέσσερα ονόματα έχω εγγεγραμμένα συναδέλφων που επιθυμούν να παρέμβουν. Μακοβέη πρώτη η κυρία Ζήπελ, επίσης Σεφ Ας δώσουμε πρώτο λόγο στην κυρία Μακοβέη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρόκειται για το πιο αυστηρό μήνυμα που έχει αποστείλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη Ρουμανία. Και μιλώ για όλες τις εκθέσεις MCV μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποιεί ότι υπάρχει κίνδυνος να ξανανοίξουν θέματα τα οποία είχαν θεωρηθεί ότι είχαν κλείσει πλέον στην τελευταία έκθεση CVM όπως εξήγησε μόλις ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα να ανοίξουν ξανά κεφάλαια τα οποία έχουν κλείσει αποτελεί ένα βήμα προς τα πίσω. για την ίδια τη χώρα και σε αυτό ευθύνεται η κυβέρνηση. και παραβιάζει τις υποχρώσεις της ε, χώρας. Λέει η, Ευρωπαϊκή, λέει η κυβέρνηση ότι δεν χρειαζόμαστε CVM για την Ρουμανία. Όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασκεί την εποπτεία και υπάρχει CVM που όμως οι πολιτικοί μας θεωρούν ότι χρειάζεται θα πρέπει να γίνονται σεβαστές οι συστάσεις της εκθέσεως. Και βεβαίως η CVM κάποια στιγμή θα λήξει. Στην έκθεση της Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η δικαιοσύνη στην Ρουμανία αποτελούν σημαντική πηγή ανησυχία. Εμείς αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει αυτό και θα πω σε λεπτομέρειες. Μιλούμε για την τροποποίηση της νομοθεσίας σχετικά με την δικαιοσύνη και μάλιστα με ε, κατεπήγοντα χαρακτήρα. Πού, βρέθηκε, ο κατεπήγον χαρακτήρας. Οι τροποποίησεις αυτές υπάγουν την ε, δικαιοσύνη στην πολιτική. ενώ την τελευταία δεκαετία η δικαιοσύνη τα πήγε καλά με τις μεταρρυθμίσεις προσπαθώντας να εξασφαλίσει την ισονομία. Τώρα, οι πλειοψηφίε του Κοινοβούλιο οδηγούν τη χώρα προς τα πίσω. Υπάρχει απόσταση μεταξύ της πολιτικής βούλησης και των θεσμών. Τώρα όμως η σημερινή κυβέρνηση κάνει βήματα προς τα πίσω και δεν ενδιαφέρεται καθόλου για τις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας είπε ότι προεβδομάδος όταν δημοσιεύτηκε η έκθεση ζητήθηκε από το Ρωμανικό Κοινοβούλιο ζήτησε το Ρωμανικό Κοινοβούλιο από την Επιτροπή της Φενετίας να κάνει συστάσεις. Τώρα όμως, για την τροποποίηση της νομοθεσίας περί δικαιοσύνης, τώρα όμως, ο πρόεδρος της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής στη Ρουμανία που μέσα στη νύχτα έκανε ε, μεταρρυθμίσεις σαν κλέφτης λέει ότι δεν θα ζητήσει στάσεις από την Επιτροπή της Βενετίας και αμέσως την εβδομάδα όπου μας λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα πρέπει να ζητηθούν οι, θα ζητηθεί τη Επιτροπή Βενετία. Και ο ίδιο ο πρόεδρο τη Κοινοβουλευτική Επιτροπή στη Ρουμανία λέει όχι. Αυτό που θέλω να πω εν τέλει για τους Ρουμάνους πολίτες είναι ότι οι συστάσεις πρέπει να εφαρμοστούν, όχι να αγνοηθούν. Και αυτό διότι η χώρα μας θα πρέπει να προχωρήσει προς τα εμπρός. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να σύρεται προς τα πίσω από ορισμένους πολιτικούς. Οι πατριώτες ε, Ρουμάνοι πρέπει να συμβάλλουν σε μια πρόοδο της χώρας προς τα εμπρός και όχι αυτά που κάνουν τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού. Εσείς τώρα κύριε, ευχαριστώ. Πολιτική σταθερότητα, αποφασιστικότητα και πρόοδος. Αυτά ζητούνται στις συστάσεις. Αυτά περιλαμβάνονται στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την πρόοδο της Βουλγαρίας για την CVM. Σημειώσουμε ακόμη ότι πρόκειται για την πιο θετική έκθεση πιθανότατα σχετικά με την πρόοδο της Βουλγαρίας στα πλαίσια του Μηχανισμού Συνεργασίας και Επαλήθευσης. Η έκθεση προβαίνει σε θετική αποτίμηση των όσων έχει πράξει η κυβέρνηση. Μπορέσαμε δηλαδή να καλύψουμε τις καθυστερήσεις που οφείλονταν στις πρόορες εκλογές. Συγχαίρω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την συνέχεια που εμφανίζει στις τελευταίες δύο εκθέσεις της, οι οποίες περιλαμβάνουν ξεκάθαρα κριτήρια και κάτι το οποίο δεν ήταν ε, ίσως προφανές στις προηγούμενες εκθέσεις. Πάντως, η σημερινή έκθεση δεν περιλαμβάνει νέες συστάσεις και για πρώτη φορά προσφέρει μια ξεκάθαρη προοπτική για, την, για το μηχανισμό συνεργασίας και επαλήθευσης και την λήξη της ισχύω του που θα επέλθει όταν συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις με τον ίδιο ρυθμό που διεξάγονται τώρα. Με τις συστάσεις ε, για τις οποίες μιλούμε εφόσον αυτές ληφθούν υπόψη, ο CVM θα λήξει. Ο CVM έχει εξαντλήσει τη χρησιμότητά του και είναι πλέον διακριτικός, ε, δηλαδή ε, σημαίνει διάκριση. Χρησιμοποιήθηκε από τα κόμματα στις προεκλογικές εκστρατείες. Πέρσι ε, απευθύνθηκε έκκληση για δημιουργία νέου μηχανισμού που θα εφαρμόζεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και όχι μόνο στην ε, Ρουμανία και Βουλγαρία. Και ελπίζουμε ε, να δούμε το μηχανισμό αυτό να εφαρμόζεται. Ευχαριστώ. Να μην σας υπενθυμίσουμε ότι αυτά τα πράγματα συνεχίζονται από το 2007. Για μένα μου φαίνεται σαν συμμετοχή σε μια ιεροτελεστία ή για να το πω μια ε, γιορτή της επόμενης έκθεσης. Δηλαδή, τη μια χρονιά σημειώνονται παραλήψη στη συμπεριφορά των ρουμανικών αρχών που εξισορροπούνται όμως από άλλη αξιοσημείωτη πρόοδο. Την επόμενη χρονιά έχουμε σημαντική και αξιόλογη πρόοδο η οποία εξορροπείται πάλι με τη σειρά από παραλήψεις της κυβέρνησης. Μια χρονιά η Ρουμανία βαθμολογείται άσχημα, την άλλη χρονιά βαθμολογείται άσχημα η Βουλγαρία. Εάν το εγχείρημα είναι άχρηστο. Είναι άχρηστο, εγώ νομίζω όχι. Διότι υπάρχουν δύο συνέπειες και οι δύο βεβαίω αρνητικές. Η πρώτη εκ των συνεπειών αυτών είναι ότι η Ρωμανία και η Βουλγαρία παραμένουν εκτός χώρου Σέγγεν επαόριστον. Η δεύτερη συνέπεια που κατά τη γνώμη μου είναι ακόμα πιο σοβαρή είναι ότι και οι δύο χώρες, μάλλον οι δύο κυβερνήσεις, η Ρωμανική και η Βουλγαρική, θα συνεχίσουν να παραβαίνουν τον νόμο και να δρουν με διεφθαρμένο τρόπο εν γνώση τους και θεωρώντας ότι δεν πειράζει και ό,τι και να κάνουν ή να παραλείψουν ο δεν θα επιβάλλεται ως αποτέλεσμα της συμπεριφοράς τους, παρά μόνο ως αποτέλεσμα πολιτικών αποφάσεων που ξεφεύγουν από, την... από τα χέρια των κυβερνήσεων. Μακάρι να ήταν επιτυχή στο μου Φοβούμαι όμως ότι δεν είναι. Ε, ευχαριστώ κυρία Σίπελ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δυστυχώς είχα διάφορες ευκαιρίε να παρακολουθήσω τις εκθέσεις CVM e ξανά και ξανά και θυμούμε την τελευταία περίπτωση, τελευταία τέτοια ευκαιρία δηλαδή, ότι στην έκθεση λεγόταν ναι υπάρχει κάποια πρόοδος αλλά χρειάζεται και άλλη δουλειά. Και εν προκειμένου συμφωνώ με τον συνάδελφό μου που μόλις μίλησε για τα προβλήματα και εγώ θεωρώ ότι ναι μεν έχει επιτελεστεί πρόοδος ξανά και ξανά τα τελευταία χρόνια υπάρχει όμως μια πολιτική απόφαση να μην λήξει ο CVM, διότι οι χώρες μέλη δεν θέλουν Βουλγαρία, Ρουμανία να, μπει στο χώρο, να μπουν στο χώρο Σέγγεν. Όμως υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία πρέπει να θίξουμε. Και θέλω να κάνω ένα σύντομο σχόλιο για το ερώτημα εάν ορισμένες χώρες μέλη θα πρέπει να έρθουν σε επαφή και να συνεργαστούν με την Επιτροπή της Βενετίας. Εν προκειμένου θέλω να τονίσω ότι υπάρχουν πάνω από μια ή δύο χώρες που δεν θέλουν να ακούσουν την Επιτροπή Βενετίας, ούτε θέλουν να συνεργαστούν μαζί της. Η διαφορά είναι ότι οι χώρες αυτές δεν αντιμετωπίζουν CVM. Αυτή είναι η μοναδική διαφορά. Όταν πρόκειται για τη Ρουμανία λοιπόν, στην περίπτωση αυτή όπου ακούμε ότι σημειώνεται κάποια πρόοδο, αλλά μετά ακούμε και κάποιες αρνητικές θέσεις, θα ήθελα να γνωρίζω, να αναγνωρίζω σαφώς, διότι διεξήχθη προμηνών εδώ στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου συζήτηση για τη Ρουμανία. Δυστυχώ δεν μπόρεσα να παρακολουθήσω ολόκληρη την εκθέση. Θέλω να μάθω όμω, ποιε είναι οι προτάσει για νομοθετικέ ρυθμίσει τότε και ποιε είναι οι συγκεκριμένε νομοθετικέ προτάσει τώρα, ποιε είναι οι διαφορέ από τότε όταν διεξήχθη η συζήτηση για τη Ρουμανία και ποια είναι η κατάσταση και ποιοι είναι οι κανόνε τώρα. Μπορείτε να μα δώσετε παραδείγματα για το τι έχει αλλάξει εν τω μεταξύ, εάν έχει αλλάξει κάτι στην πράξη ή εάν αναφέρεστε στις κατατεθειμένες προτάσεις που βρίσκονται στο τραπέζι. Κυρία Γκόμες. θέλω να σχολιάσω. Την ε, πολιτικού χαρακτήρα στρατηγική τα προηγούμενα χρόνια, όπως ε, υπενήχθη στις προηγούμενες παρεμβάσεις, πρέπει όμως να σας πω τα όσα αποκόμισα από την επίσκεψή μου στη Ρουμανία στις αρχές ε, του μήνα, κατόπιν πρόσκλησης ε, του συναδέλφου Καταλήν Ιβάν, όπου συνομίλησα με εκπροσώπους κοινωνίας των πολιτών και με τα μέσα ενημέρωσης για τα ζητήματα που υπάρχουν στη Ρουμανία σε ό,τι αφορά την αντίληψη για τη διαφθορά και την ε, έλλειψη καταπολέμησης διαφθοράς. Μπορούμε να πούμε ότι ο κόσμος ε, εντύχεται κατά της διαφθοράς. Μέσα στο καταχύμωνο βγήκαν ε, και διαμαρτυρήθηκαν και διαδήλωσαν κατά της ε, διαφθοράς. Ε, συνάντησα λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους και πραγματικά εντυπωσιάστηκα από την ποιότητα των ε, παρατηρήσεών τους και των ε, ερευνών που διεξάγουν υπό πολύ δύσκολες συνθήκες. Και εκείνοι αναγνώρισαν ε, ότι πράγματι υπάρχει βελτίωση σε ό,τι αφορά τη δικαιοσύνη. Όμως παραμένουν ιδιαίτερα ανήσυχοι για την πάλι κατά τη διαφθορά συνολικά. Εγώ θα μιλούσα για τις ε, προσπάθειές μας, ε, ιδίως ό,τι αφορά την νομοποίηση παρανομών εσόδων ε, και για τα έγγραφα του Παναμά. και με προβλήματα που έχουμε στη χώρα μας ό,τι αφορά την εφαρμογή της τέταρτης οδηγίας για την νομοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητε. γιατί υπάρχουν πολλές ε, συμβάσεις ε, που αφορούν εκτάσεις γης με τεράστιο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και πολλές φορές εμπλέκονται και ευρωπαϊκά κονδύλια. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν αφορά μόνο τη Ρουμανία, ε, ούτε μόνο την αξιοπιστία την αξιοπιστία ε, των δημοσίων αρχών στα μάτια των Ρουμανών πολιτών, είναι και η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής. Οπότε χρειαζόμαστε μια πραγματική πολιτική προσέγγιση Και αν για να το κάνουμε αυτό πρέπει να πιέσουμε την ε, Επιτροπή της Βενετίας για να κάνει τη δουλειά της και να ε, παρεμβεί, έστω. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει έτσι διεκπαιρεωτικά ε, και να αλλάζουμε από την μια χρονιά στην άλλη βλέπουμε ότι οι Ρουμάνοι πολίτε προβληματίζουν ιδιαίτερω και είναι διατεθειμένοι να λάβουν ε, το μερίδιο τη ευθύνη του Πρέπει να του βοηθήσουμε. Ευχαριστούμε κύριο ε, Στάνισερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είχα το προνόμιο, ή μάλλον όχι και τόσο προνόμιο, να παρακολουθήσω αυτή την έκθεση από την αρχή αυτή τη σειρά εκθέσεων από την αρχή του το 2007. Γενικά καταλήγω ότι αν από την αρχή της διαδικασίας ο μηχανισμός αποτελούσε ισχυρό κίνητρο για τις ε, κυβερνήσεις στη Βουλγαρία για να προβούν τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, ε, τελικά βλέπουμε ότι όλα αυτά γίνονται πλέον λίγο τελετουργικά, χωρίς να αλλάζει κάτι στην ουσία. Γιατί ε, στην αρχή στη χώρα μου υπήρχε μεγάλο άγχος και προσμονή για την, για την κάθε έκθεση. Ε, τώρα πια έχει γίνει λίγο ρουτίνα. που δεν επιφέρει κάποια θετική τουλάχιστον αλλαγή. Και να θεωρώ ότι το πρόβλημα είναι και, αφορά και την γενική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί ένα από τα κριτήρια που υιοθετήθηκε από την αρχή είχε αποφασιστεί τότε, το 2007, για την ε, συνταγματική αναθεώρηση. Πουθενά δεν αναφέρθηκε ότι αυτή η παράγραφος έχει ήδη γίνει. Έχει ήδη ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και νομίζω ότι αυτό είναι ανησυχητικό. Ο μηχανισμός λοιπόν συνεχίζεται χωρίς ε, κάποια σαφή κάποιο σαφές χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωσή του, ενώ βλέπουμε ότι τα κριτήρια τη Κοπεχάη στην Ευρωπαϊκή Ένωση που καλύπτουν ζητήματα δημοκρατία, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κράτου δικαίου, παραβιάζονται σε πολλά από τα μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν θέλουμε λοιπόν τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι ε, αποτελεσματικά και αξιόπιστα πρέπει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση να αξιολογούνται αυτά τα ζητήματα. Να μην γίνονται όλα αυτά επιλεκτικά και ούτε να αξιοποιούνται όπως σε αυτή την περίπτωση με το CVM απέναντι στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία ως μέσω πίεσης για άλλους πολιτικούς σκοπούς. Ήδη αναφέρθηκε το θέμα της Σέγγεν. Και το λέω ευθέως. Αυτό που συμβαίνει στο Συμβούλιο με την ε, επιχρόνια τώρα αναστολή ή μάλλον ε, καθυστέρηση της ε, προσχώρησης των δύο αυτών χωρών στη ζώνη Σέγγεν, ενώ ξέρουμε ότι πληρούν όλα τα κριτήρια για τη συμμετοχή τους, είναι σκανδαλώδες, υπονομεύει την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνει ξεκάθαρα την εντύπωση των δύο μέτρων και δύο σταθμών και δημιουργεί ακόμα και εγχώρια ζητήματα σε χώρες. Γιατί από τη μία είχαμε εκλογέ στη μία χώρα, μετά στην άλλη, μετά στην τρίτη, άρα λέμε πρέπει να ε, ανασταλεί. Να αναβληθεί μάλλον αυτό το θέμα. Και όταν πρόκειται για ζητήματα που είναι ευρωπαϊκή αρμοδιότητα, αυτό είναι σίγουρα ένα από τα ε, βασικά παραδείγματα. Ευχαριστούμε ο κύριος Βούντα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Δεν είμαι μέλος ε, της Επιτροπής σας, αλλά εφόσον γίνεται λόγος για τη Ρουμανία, με ενδιαφέρει. Αυτή η έκθεση ορίζει με μεγάλη ευκρίνεια κάποια ζητήματα και κάποια φαινόμενα στη Ρουμανία Υπάρχει κάποια βελτίωση, αλλά δυστυχώς ε, ήμουν και εγώ Πρόεδρο τη Επιτροπή Δικαστικών Υποθέσεων στο Κοινοβούλιο. Προσπαθούσα να εφαρμόσω την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για να κλείσει η διαδικασία CBM. Δυστυχώς όμως... Υπάρχουν καταχρήσεις από πλευράς ε, κυβέρνησης, η οποία προσπαθεί να ε, πολιτικοποιήσει ε, τη δικαιοσύνη και να την θέσει, να θέσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης ε, στην υπηρεσία άλλων. καθώς και την εισαγγελία. Υπάρχουν βέβαια και θετικές εξελίξεις, όπως το όριο ηλικίας, για την πρόσβαση στο δικαστικό σώμα, όμως δυστυχώς υπάρχουν ακόμα σοβαρά προβλήματα με την τομέα τη δικαιοσύνη. και καλό είναι να ε, υπάρχει κάποια παρακολούθηση από την Ευρώπη, υπάρχουν σημαντικά ζητήματα και με άλλες χώρες όπως την Πολωνία και αλλού. Όμως, κάτι το οποίο θεωρώ πραγματικό είναι ακριβώς η προσχώρηση στη ζώνη Σέγγεν. Είναι απαράδεκτο. Και να θυμάστε ότι αυτό είναι κάτι που πραγματικά βαραίνει συναισθηματικά τους ε, πολίτες ότι υπάρχει διασύνδεση μεταξύ τη ΕΝΓΕΝ και του CVM. Η Ρουμανία έχει επενδύσει εκατομμύρια ευρώ ε, σε εξοπλισμό από άλλες χώρες για να διασφαλίσει τη σταθερότητα ε, στην ευρύτερη περιφέρεια. Παρόλε τι προσπάθειές μας δεν μα αφήνουν να μπούμε στι ζώνη ΕΝΓΕΝ, το οποίο είναι πραγματικά άδικο. Και να πω προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βέβαια δεν αφισβητώ τις ενέργειές της, αλλά θα μπορούσε στην Επιτροπή Ρέτζι και Αγρί όταν μιλούμε για την απορρόφηση πόρων, πρέπει να βρούμε τρόπους για τα κάτι μέλη, ε, ούτως ώστε αυτό που συμβαίνει σε μία χώρα να μην ε, εξαρτάται από το τι συμβαίνει σε μία άλλη. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένας κώδικα δοντολογία και βέλτιση των πρακτικών σε ό,τι αφορά ε, την ε, πρόσβαση ε, και την απορρόφηση των ευρωπαϊκών πόρων. Η κυρία Μακοβέ, υπήρξε ένα σφάλμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποτέ δεν συνέδεσε τις εκθέσεις CVM με την πρόσβαση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στη ζώνη Σένγκεν. Ποτέ. Μόνο ένα κρατός μέλος, 100 χώρες, πριν από 4-5 χρόνια, είχε πει ότι θα θέλαμε 2-3 διαδοχικές θετικές εκθέσεις CVM. Ποτέ δεν το έχει πει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως. Δεν ισχύει λοιπόν ότι δεν μα επέτρεψαν να προσχωρήσουμε στη ζώνη Σέγγεν εξαιτία αυτού. Όχι, δεν είναι γι' αυτό το λόγο. Είναι επειδή εμεί έχουμε πολιτικού που λένε ψέματα, που, κλέν, που κλέβουν. Δεν έχει καμία σχέση με το CVM που αφορά την ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Και οι πολίτε αυτό θέλουν, δικαιοσύνη. Και εγώ θέλω βέβαια να μπει η Ρουμανία και η Βουλγαρία στη Σέγγεν, αλλά να πω σε όλου όσοι πιστεύουν ότι υπάρχει διασύνδεση μεταξύ των δύο ότι αυτό δεν ισχύει. Κυρία Σίπελ, συγγνώμη, αλλά κατόπιν όλων αυτών θα ήθελα να προσθέσω ότι ίσως δεν υπάρχει επίσημο έγγραφο. Όμως, τα κράτη-μέλη μας είπαν ε, πολλές φορές πέρσι ότι εξαιτία του CVM δεν θα επιτρέψουν στα δύο κράτη-μέλη να ε, έχουν πρόσβαση στον χώρο Σέγγεν. Να μην λέμε με ψέματα λοιπόν εδώ στην ε, αίθουσα και επειδή ο συνάδελφο ανέφερε την Πολωνία, να μην ξεχνάμε ότι εδώ και έξι χρόνια έχουμε προβλήματα με την Ουγγαρία. Και συμφωνώ ότι αν αρχίσουμε να κατανομάζουμε κράτη-μέλη, να, να τους λέμε όλου. Να λέμε όλα τα κράτη-μέλη που υπάρχουν προβλήματα και όχι επιλεκτικά, ανάλογα με τις ε, συμπάθειε και αντιπάθειές μα. Να ξέρω ότι για την Ουγγαρία υπήρξαν πολλέ συστάσει τη Επιτροπή Βενετία, λέει ο Κύριος Λέσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας. Θα θυμάστε ότι ο πρόεδρος Γιούγκερ στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης ε, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο κράτος δικαίου. Είναι λοιπόν ένα γενικό οριζόντιο μέλημα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, βέβαια, είναι ιδιαίτερο το πλαίσιο του CVM. που οδηγεί τελικά και στη συνδέξη των εκθέσεων. Ο πρόεδρο Γιούνκερ στην ομιλία του επίση ξεκαθάρισε και την ε, θέση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προσχώρηση τη Βουλγαρίας και τη Ρουμανία στην ε, ζώνη Σέγγεν. Νομίζω ότι πραγματικά ξεκαθάρισε το τοπίο και στην έκθεση του Ιανουαρίου υπάρχει ρητή αναφορά στο γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν συνδέει τα δύο ζητήματα. Γι' αυτό εξακολουθεί να αποτελεί τη θέση της Επιτροπής. θα ήθελα να τονίσω ένα σημείο για τις συστάσεις. Πράγματι, οι συστάσεις που έκανε η Επιτροπή τον Ιανουάριο είναι ακριβώς οι ίδιες με τις συστάσεις αυτή τη στιγμή. Οπότε δεν έχει αλλάξει κάτι στις συστάσεις. είναι τα ίδια βήματα που θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα πρέπει να ε, γίνουν για να θεωρήσουμε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις. Θέλουμε λοιπόν ε, να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με τα δύο κράτη-μέλη προκειμένου ε, να πληρωθούν αυτές οι συστάσεις ε, το συντομότερο δυνατόν. Ευχαριστούμε πολύ. Φτάσαμε στο τέλος ε, της σημερινής συνεδρίασης. Να ανακοινώσω μόνο ότι η επόμενη συνεδρία θα γίνει στις 27 και 28 Νοεμβρίου. Καλό σας βράδυ.